Σας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

Αγαπητοί συνάδελφοι, καλωσορίζατε στη συνεδρίαση της Επιτροπής μας. Εχθές ήταν αργία στο Βέλγιο, εξού και η εβδομάδα αρχίζει για μας μόλις σήμερα. Äh, για το σημείο 1 της ημερήσιας διάταξης έχω να πω τα εξής. Αύριο το πρωί ε, θα έρθει εδώ ο κύριος Δήμας, 11 ε, με 12.30 και το σημείο 6 έχει αποσυρθεί. Τα καλλιντικά και η αντίστοιχη οδηγία αναβάλλεται για ευθετότερο χρόνο. Εγκρίνεται έτσι την ημερήσια διάταξη. Ωραία. Ε, ούτως θα προχωρήσω γλώσσες όλες εκτός από εστονικά, λετονικά και μαλτέζικα. Επίσης έχουμε και ένα τηλεοπτικό συνεργείο της φλαμαδικής τηλεόρασης που παρακολουθεί και ακολουθεί και συνοδεύει τις συναδέλφους Φάντεν και Τελάνχε αν δεν διαφωνείτε θα τραβήξουν κάποια πλάνα. Έτσι κι αλλιώ είμαστε στο διαδίκτυο, στη διάθεση της ανθρωπότητα παγκοσμίω. Μπορεί ο καθένας να παρακολουθήσει τις ε, εργασίες μας. και έρχομαι στο σημείο 2. Το μόνο που θα ήθελα να σας πω είναι ότι την πέρασμένη εβδομάδα έγινε η σύνοδος κορυφής της Βρυξέλλης και εκτός από τη συνθήκη της Σαββόνας ασχολήθηκε και με την προστασία του κλίματος και από πλευρά μας ε, πρέπει να πούμε ότι μας χαροποιεί που τα 27 κράτη-μέλη είναι προσιλωμένα στο πακέτο για το κλίμα. 30% μείωση δηλαδή μέχρι το 2020 να δεσμευτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση αν τα άλλα βιομηχανικά κράτη κάνουν αντίστοιχες ρυθμίσεις. Είναι σημαντικό αυτό παραμονές της Κοπεχάγης και Δεύτερον, για τη χρηματοδότηση του συνολικό πακέτο αυτό των 100 δισεκατομμυρίων ευρώ για το έτος 2020 έγινε δεκτό. Βέβαια, ακούσαμε όλοι και είδαμε ότι το συγκεκριμένο μερίδιο που αναλογεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση εκκρεμεί. Παρέμεινε ανοιχτό εν μέρη και για λόγους τακτικούς, αλλά και επειδή υπάρχει μια διαμάχη ποιος θα πληρώσει πού και πόσα και μέχρι την Κοπενχάγη χρειάζεται να γίνει ακόμα δουλειά. Περνώ όμως στο άλλο θέμα που θα συζητηθεί την Πέμπτη εκτενέστερα η αντιπροσωπεία της Επιτροπής μας στην Ουάσιγκτον και συζήτηση με τους συναδέλφους στο Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Ευρώπη παραμένει ηγέτης το θέμα της ε, προστασίας του κλίματος και καταπολέμησης κλιματικής αλλαγής. Άλλοι χρειάζονται να εργαστούν πολύ περισσότερο. Εμείς έχουμε και νομοθεσία και θα θέλαμε και συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Για την αντιπροσωπεία όμως και το ταξίδι αυτό θα συζητήσουμε περισσότερο και θα φερώσουμε περισσότερο χρόνο την Πέμπτη το πρωί. Έρχομαι λοιπόν στο σημείο 3 τώρα. Έγκριση των πρακτικών της 30 Σεπτεμβρίου. Αν δεν έχετε επιφυλάξει, μέχρι το τέλος συνεδρίασης ε, θα θεωρηθούν εγκριθέντα τα πρακτικά και πάμε στο πρώτο ουσιαστικό σημείο του απογεύματός μας. Ανταλλαγή απόψεων με τον κύριο Χέρτ Ντάνσετ, που είναι εκτελεστικός διευθυντής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων στο Ελσίνκι. Καλώς ορίσατε θερμά. Εσείς και οι συνεργάτες σας. Ε, το REACH ήταν από τα προγράμματα μαμούθ ε, της ε, περασμένης θητείας. Πολλοί ε, από τους βουλευτές που ήταν μέλη και στην προηγούμενη θητεία έκαναν πολλή δουλειά, αφιέρωσαν και πολύ χρόνο σε αυτή την υπόθεση και στην τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής μας είχαμε ήδη κάνει ένα γύρο ερωτήσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εφαρμογή του REACH, οπότε είναι πάρα πολύ επίκαιρο που ε, μας κάνετε επίσκεψη σήμερα για να μπορέσουμε να εμβαθύνουμε στη συζήτηση αυτή. Είστε από τους σημαντικούς οργανισμούς στην Ευρώπη που μας χρειάζονται για να ανταποκριθούμε στο έργο μας και στο καθήκον μας και είμαι βέβαιος ότι η Επιτροπή μας θα ενδιαφερθεί πάρα πολύ να σας ακούσει πώς έχετε αναπτύξει τη δουλειά σας, ε, ποιες είναι οι προτεραιότητες και σίγουρα θα κάνουν και ερωτήσεις. Παρακαλώ, έχετε αμέσως το λόγο. Dear Chairman, members of the committee. Αγαπητέ Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη της Επιτροπής, χαίρομαι ιδιαίτερα που έχω την ευκαιρία να σας μιλήσω για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στον οργανισμό μας μετά από την τελευταία μας ανταλλαγή απόψεων τον Ιούλιο του περασμένου έτους. Θα ήθελα να ξεκινήσω καταρχήν ευχαριστώντας σας και να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου για την υποστήριξή σας κατά τη διάρκεια της ε, διαδικασίας ε, ε, του προϋπολογισμού γιατί χρειαζόμαστε αρκετούς ικανούς πόρους για τον επόμενο χρόνο που θα είναι ο πιο κρίσιμος για την εφαρμογή του REACH. Η Επιτροπή σα ξεκίνησε τη διαδικασία διόρθωση που οδήγησε στην πρώτη ε, ψηφοφορία με πρώτη ανάγνωση την 1η Οκτωβρίου και βασίζομαι στην συνεχιζόμενη σα υποστήριξη ώστε να διασφαλίσουμε πως το αποτέλεσμα αυτό θα επικυρωθεί στη δεύτερη ανάγνωση αργότερα φέτο σε δεύτερο λόγο θα ήθελα να σας ε, να ευχαριστήσω σε πιο προσωπικό επίπεδο την κυρία Χάση ε, για την υποστήριξή της και την προσήλωσή της στα θέματά μας τα τελευταία δύο χρόνια, αλλά και τους ε, δύο εκπροσώπους σας, τον κύριο Λάγκη και τον Αλεξάνδρου οι οποίοι συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο και που μας βοήθησαν στην διαδικασία κίνησης λειτουργίας του οργανισμού. Να καλωσορίσω και όλα τα νέα μέλη του Διοικητικού μας Συμβουλίου, τον Guido Σακώνη και τον κύριο Νασάουερ που είναι δύο από ε, του βασικού σχεδιαστέ του ΡΙΤΣ κατά τη διάρκεια τη προηγούμενη θητεία. Είναι εξαιρετικά ε, ε πολύτιμοι γιατί έχουν μεγάλη εμπειρία στα θέματα και θα μας βοηθήσουν έτσι να αντιμετωπίσουμε τις μελλοντικέ προκλήσεις. Πριν να δούμε το μέλλον θα ήθελα να σας θυμίσω την προέλευση του οργανισμού και πόσο πολύ έχουμε προχωρήσει. Ο ιδιωτικό κανονισμός του ΕΚΑ, το ΡΙΤΣ, υιοθετήθηκε το Δεκέμβριο του 2006 με μεγάλη υποστήριξη από Συμβούλιο και Κοινοβούλιο. Το ΕΚΑ νομικά εδρεώθηκε τον Ιούνιο του 2007. Ήταν και η πρώτη μου ημέρα εργασίας στο Ελσίνκι χρόνο μετά, την 1η Ιουνίου 2008, μια αρχική ομάδα, 35 υπαλλήλων της Κομισιόν και περίπου 70 προσωρινοί υπάλληλοι, με επιτυχία διαχειρίστηκαν την έναρξη λειτουργίας του οργανισμού και την μετατροπή από την προηγούμενη νομοθεσία. Την ίδια μέρα η ΕΚΑ ήταν έτοιμη να δεχτεί ηλεκτρονικές υποβολές ε, ε, εγγραφών και εγγραφών ε, χημικών ουσιών. Ξεκινήσαμε λοιπόν με πολύ καλή αρχή. Έξι μήνες μόλις μετά, την 1η Δεκεμβρίου 2008, ο οργανισμός με επιτυχία ολοκλήρωσε την περίοδο προεγγραφής, ενώ δέχτηκε 2,7 εκατομμύρια υποαιτήσεις σε έναν ε, μη αναμενόμενο οργανισμό και όπως καταλαβαίνετε ο όγκος αυτός ήταν 30 φορές μεγαλύτερος από τον αναμενόμενο και έφτασε τις τελευταίες εβδομάδες, πράγμα το οποίο απέτησε πολύ μεγάλη ευελιξία και πολύ σκληρή δουλειά από όλους τους συναδέλφους. Είμαι πολύ περήφανος για αυτούς και για το, τα όσα καταφέραμε όλοι μαζί. Οι εταιρείε που, που ήθελαν να προεγγραφούν εγκαίρω το μπόρεσαν να το κάνουν. Τον Οκτώβριο του 2008 εκδόθηκε η πρώτη ε, εκδοχή ε, για τις ε, πολύ επικίνδυνες ουσίε που περιλαμβάνει 15 ε, ουσίες από 17 κράτη-μέλη για τον περαιτέρω έλεγχο κινδύνου. Την 1η Ιουνίου 2009 ε, ο ΕΚΑ έστειλε τις πρώτες συστάσεις για τις 7 από τις 15 αυτές ουσίες προς την Κομισιόν ώστε να συμπεριληφθούν στον κατάλογο ε, αδειοδότησης. Πέρα από αυτές τις μεγάλες ε, προθεσμίες που είχαμε και που ορίζονταν από τον κανονισμό REACH, υπάρχει φυσικά και η καθημερινή εργασία της, ε, του οργανισμού ΕΚΑ, ε, καθημερινής βάσης οι ευρωπαϊκές χημικές εταιρείες αλλά και μη ευρωπαϊκές εταιρείες υποβάλλουν ε, μέχρι και εκατοντάδες φακέλους μέσω του REACH για... και μάλιστα εκπονούμε εμείς ε, επιστημονικές αξιολογήσεις για πάνω από το 5% εξ αυτών. Υπάρχουν περιορισμοί, αδειοδοτήσεις, αναρμονισμένη ταξινόμηση και ετικετοθεσία των χημικών ουσιών. Όλα αυτά έχουν ξεκινήσει και ο κατάλογος των υποψηφίων αυτή τη στιγμή στιγμή ενημερώνεται για πρώτη φορά και ο ΕΚΑ προετοιμάζεται ώστε να ανταποκριθεί στον αυξανόμενο όγκο εργασία λόγω όλων αυτών των διαδικασιών τα επόμενα χρόνια. Ο ΕΚΑ επίση συμβάλλει στι συνεδριάσει τη Κομισιόν με τι αρμόδιε αρχέ και φέτο οργάνωσε τρει ειδικέ ε, συνεδριάσει του δικτύου ώστε να συμφωνήσουμε για μια κοινή προσέγγιση για την αξιολόγηση, τον περιορισμό αλλά και την αδειοδότηση και να μπορέσουμε να ενεργοποιήσουμε περισσοτερα περισσότερα κράτη-μέλη για τα θέματα αυτά. Ένα σημαντικό τμήμα της καθημερινής μας εργασίας γίνεται σε συνεργασία με τις επιτροπές και τα δίκτυα που συγκεντρώνουν την Κομισιόν, τα κράτη-μέλη και τους ε, ενδιαφερόμενους φορείς το Διοικητικό Συμβούλιο, οι τρεις επιστημονικές επιτροπές και το Φόρουμ για την επιβολή του ΡΙΤΣ, καθώς και τα τρία άλλα δίκτυα ε, συνεδριάζουν τακτικά στο Ελσίνκι. Αυτές οι συνεδριάσεις βοηθούν στο να εξαπλωθούν οι καλές πρακτικές και να βελτιωθεί ο συντονισμός ολόκληρη την Ευρώπη. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι είναι χαρά μου που βλέπω τόσο ψηλού επίπεδου πυρογνώμονες από ολόκληρη την Ευρώπη να συνεργάζονται στο Ελσίνκι με στόχο να βελτιώσουν την ασφαλή χρήση των χημικών προϊόντων σε ολόκληρη την Ένωση, ενώ ταυτόχρονα ε, προσπαθούν ώστε να επιτευχθούν και οι υπόλοιποι στόχοι του κανονισμού REACH. Ο ΕΚΑ ε, επίση ε, κάνει μια προοδευτική πολιτική για τη συμμετοχή των φορέων και του, και του ευρύτερου κοινού. Εμεί έχουμε δύο ημερίδες των ενδιαφερόμενων φορέων κάθε χρόνο, ώστε να μπορεί καθένα να συμμετέχει και ε, συμμετέχουν και εκπρόσωποι των κρατικών ε, οργανισμών που θέλουν να συμμετέχουν. Ακόμα και αποζημιώνουμε το κόστος συμμετοχής ε, όλων των ε, εκπροσώπων των ενδιαφερόμενων φορών. Είμαστε περήφανοι που διαφυλάσσουμε την διαφάνεια του κανονισμού REACH. Εμείς ε, ε, καθοδηγούμε και τις εταιρείες για το πώς να πληρούν τις ευθύνες τους υπό τον κανονισμό REACH. 600 ερωτήσεις απαντούμε κάθε μήνα. Δίνουμε κατευθύνες γραμμές βασικά σε όλες τις ευρωπαϊκές τις γλώσσες της Ένωσης και επίσης κάνουμε και διάφορα σεμινάρια. Η διαχείριση, η διοίκηση του ΕΚΑ εισήγαγε και διάφορα διαχειριστικά εργαλεία ώστε να παρακολουθούνται οι διάφορες διαδικασίες και οι αναφορές. Είναι πολύ σημαντικά αυτά τα, ε, αυτές οι εργασίες και ο έλεγχος της ε, Κομισιόν απέδειξε πως ακολουθούμε τις καλύτερες πρακτικές. Μετά από αίτημα της Κομισιόν, ο ΕΚΑ συμβάλλει και στις διεθνείς δραστηριότητες της Ένωσης για, τη, ε, για την ασφαλή χρήση των χημικών προϊόντων, κυρίως στο πλαίσιο του ΟΣΑ. Ενώ οι συμμετέχοντες φορείς και οι παρατηρητές αναγνωρίζουν πως ο ΕΚΑ έκανε πολύ επιτυχημένη αρχή, χάρη και στην ε, πολύτιμη υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι οι μεγαλύτερες προκλήσεις βρίσκονται μπροστά μας. Και θα σας παρουσιάσω ποιες είναι αυτές. Τον επόμενο χρόνο, ο επόμενος χρόνος, μάλλον θα είναι ο πιο δύσκολος μάλλον και αυτό γίνεται ενώ εκπαιδεύουμε πάνω από 100 νέους υπαλλήλους. Κατά τη διάρκεια του 2010 θα πρέπει να χειριστούμε δεκάδες χιλιάδες φακέλους εγγραφής και εκατοντάδες και μάλλον και εκατομμύρια ε, αιτήσει για ταξινόμηση και διοδότηση. Θα πρέπει να ανταποκριθούμε σε δύο σημαντικέ προθεσμίε με ένα μήνα μόνο διαφορά μεταξύ του, με τα Χριστούγεννα ανάμεσα. Πολύ μαζικό έργο που δεν έχει γίνει ποτέ άλλοτε πουθενά στον κόσμο. Και αυτό θα το κάνουμε στο τρίτο, τρίτο έτος λειτουργίας μας, πριν ακόμα να έχουμε συμπληρώσει το απαραίτητο προσωπικό μας. Άρα λοιπόν η ετοιμότητα του επιστημονικού προσωπικού μας αλλά και του, των ηλεκτρονικών μας προγραμμάτων θα είναι πολύ κρίσιμα για να μπορέσουμε να τηρήσουμε τις προθεσμίες που περιλαμβάνονται το κανονισμό. Φυσικά εμείς στον ΕΚΑ δεν είμαστε οι μόνοι που δουλεύουμε σκληρά για να λειτουργήσει το και οι εταιρείε συνεργάζονται όσον αφορά τα φόρα ε, Ενημέρωση για τις ουσίες ώστε να προετοιμάσουν όλες ε, τις κοινοποιήσει τους για τι ετικετοθεσίες ε, και ταξινόμηση των ουσιών. Σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να καταγραφούν όλα τα στοιχεία ώστε να μην υπάρξουν ε, περιτές δοκιμές και κόστος. την Άνοιξη η βιομηχανία μας κάλεσε να τους, βοηθήσουμε, να τους σε αυτό το φόρουμ γιατί η εργασία δεν λειτουργούσε αρκετά γρήγορα. Αποτελούν όμως τα φόρα αυτά τόσο πολύ ουσιαστικό τμήμα της διαδικασίας εφαρμογής του ΡΙΤΣ που η ΟΕΚΑ μαζί με την Κομισιόν ξεκίνησε μια εκστρατεία ενημέρωσης με τον τίτλο ε, «Το ρολόι τρέχει, φτιάξτε το φόρουμ σας τώρα». Χρειάζεται λοιπόν να δουλέψουμε πολύ γρήγορα γιατί χρειάζεται πολύς χρόνος για να ετοιμαστεί ένα ντοσχέ καταγραφής. Ο ΕΚΑ συνεχίζει να υποστηρίζει τις βιομηχανίες, για παράδειγμα παρέχοντας ειδικέ υπηρεσίες για την ε, καταγραφή των ουσιών, καθώς και για να βοηθήσει τα κράτη-μέλη να βοηθήσουν και αυτά με τη σειρά τους τις μικρές εταιρείες στα φόρα ε, αναγνώρισης των ουσιών το Δεκέμβριο θα ξεκινήσουμε και μια νέα εκστρατεία ενημέρωσης για την ετικετοθεσία. Ε, θέλουμε να θυμίσουμε στις επιχειρήσεις τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με τον νέο κανονισμό κυκλοθεσίας και συσκευασίας που υιοθετήσατε εσείς στα τέλη του περασμένου χρόνου. Προετοιμάζοντας αυτές τις κρίσιμες λοιπόν ε, προθεσμίες και ε, περιόδους εχμής, εμείς εργαζόμαστε και για το σύστημα πληροφορικής μας ώστε να μπορούμε να χειριστούμε μεγαλύτερους όγκους καταγραφής και κοινοποιήσεων ουσιών. Επίσης αναπτύσσουμε μια ολόκληρη σειρά επιστημονικών εργαζόμενων εργαλείων ε, πληροφορικής για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε για την καταγραφή και την επιβολή. Προοδεύουμε επίσης πολύ καλά με ένα πιλωτικό πρόγραμμα για τη διάδοση πληροφοριών ε, για τις ήδη εγγεγραμμένες ουσίες ε, προς το κοινό. Πράγμα που θα ξεκινήσει πριν το τέλος του τρέχοντος έτους και όπου θα μας βοηθήσει και μια ομάδα εργασίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Ταυτόχρονα γνωρίζουμε απόλυτα την ανάγκη προστασίας ε, των εμπιστευτικών πληροφοριών των εταιριών, εταιριών που πρέπει να μας υποβάλουν ε, τα στοιχεία αυτά ως τμήμα της διαδικασίας REACH. Ο ΕΚΑ πολύ σοβαρά διερευνεί τα θέματα της ασφάλειας των πληροφοριών και απαιτεί παρόμοια μέτρα από πλευρά των κρατών και ε, της Κομισιόν πριν τους δώσει την άδεια για πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές. Εν τέλει, όπως ε, θα καταλάβατε, έχουμε μεγάλη πίεση, έχουμε κάνει εξαιρετική αρχή, αλλά οι προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε το 2010 είναι τεράστιες. Αυτές οι πραγματικές προκλήσεις όμως δεν είναι οι μόνες που αναμένουμε. Αύριο η Επιτροπή σας θα συζητήσει για πρώτη φορά ένα νέο νομοθετικό, ε, μια νέα νομοθετική πρόταση για τα βιοκτώνα. Νέα δουλειά λοιπόν για την υπηρεσία μας και μια νέα επιστημονική επιτροπή προβλέπεται εκεί. Είναι μια ευθύνη την οποία ευχαρίστως αναλάβουμε με την προϋπόθεση ότι θα έχουμε και τους απαραίτητους πόρους φυσικά. Είμαι βέβαιος ότι η δική μου παρουσίαση δεν έκανε παρά να αναφέρει όσα κάνουμε για να προστατεύσουμε την ε, ανθρώπινη υγεία. Ξέρω επίσης ότι το Ρίτς είναι το μωρό πολλών από εσά και θέλω να σας αποδείξω πόσο καλά το φροντίζουμε και γι' αυτό με ευχαρίστηση θα ήθελα να επισήμως να σας καλέσω να έρθετε και να επισκεφτείτε τον οργανισμό μας στο Ελσίνκι, πράγμα που θα σας επιτρέψει σε εσά και σε εμά να σας ενημερώσουμε με περισσότερες λεπτομέρειες για τη δουλειά μας και να επιτύχουμε τους στόχους του Ρίτς. Θα ήμουν ευγνώμων αν οι συντονιστές και η γραμματεία διευκόλυναν μια τέτοια επίσκεψη για το πρώτο ήμιση του 2010. Πριν να κλείσω την ομιλία μου, θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας τις τρεις μεγαλύτερες μου ανησυχίες, όπου πραγματικά χρειάζομαι την υποστήριξή σας. Καταρχήν, οι συνάδελφοι και εγώ αντιμετωπίζουμε μεγάλες προκλήσεις για το 2010 και, και δεν γνωρίζουμε ακριβώς την κλίμακα της πρόκλησης μέχρι ότου να την αντιμετωπίσουμε πραγματικά. Εξαρτάται από τον αριθμό και το χρονισμό των ε, αιτήσεων που θα υποβληθούν για καταγραφή. Κατά την άποψή μας, μπορεί να κυμανθούν ανάμεσα στην αρχική πρόβλεψη της Κομισιόν και 300% περισσότερες. Η πίεση βέβαια θα ασκηθεί σε εμά ακόμα περισσότερο αν η βιομηχανία περιμένει μέχρι το τελευταίο μήνα για να υποβάλει τι αιτήσει. Χρειαζόμαστε λοιπόν ευελιξία και πόρου κατά τη διάρκεια των επόμενων ετών. Περισσότερε εγγραφέ σημαίνει περισσότερα έσοδα για τα επόμενα χρόνια, αλλά μπορεί να χρειαστούμε περισσότερο μόνιμο προσωπικό για να μπορέσουμε να χειριστούμε όλη αυτή τη δουλειά. Μπορεί λοιπόν να χρειαστώ την υποστήριξή σα και περισσότερου ανθρώπινου πόρου τα επόμενα χρόνια. Δεύτερον, αυτή η διαβεβαιότητα όσον αφορά τον όγκο και τον χρονισμό των αιτήσεων θα χρειαστεί να θα μας οδηγήσει σε συχνή αλλαγή προτεραιοτήτων μέσα στο 2010. Μπορεί να μην μπορέσουμε να προοδεύσουμε σε όλα τα μέτωπα με την ίδια ταχύτητα καθόλου όλη τη διάρκεια του χρόνου και έχω συμφωνήσει με το Διοικητικό μου Συμβούλιο ότι θα του ενημερώνω για, σε κάθε συνάντηση που θα έχουμε καρδιέρ και το 2010 για τον όγκο τη εισερχόμενη δουλειά και τι πιθανέ ανάγκε για αλλαγέ στι προτεραιότητε, ώστε να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να συμμορφωνόμαστε με τι προθεσμίε του ΡΙΤΣ. Είμαι ευγνώμων που το Διοικητικό Συμβούλιο συμπεριλαμβάνει εκπροσώπους και του Κοινοβουλίου και της Συμβουλίου και τη Κομισιόν που μπορούν να μα βοηθήσουν όσον αφορά την θέσπιση προτεραιοτήτων για τα επόμενα έτη. Απλώ χρειάζομαι να με υποστηρίξετε εσεί, να υποστηρίξετε τα μέλη σα στο Συμβούλιο μα για να μπορούν σωστά να μα ενημερώνουν και εκείνοι, για να μα βοηθήσουν. Και ε, οι προθεσμίες του επόμενου έτους απέχουν ένα μήνα μόλις η μία από την άλλη και είναι τόσο αβέβαιες και επικίνδυνες που έχουμε ξεκινήσει, όπως σας είπα, σε πολύ μεγάλες, σχεδιασμό μάλλον, συντονιστικό σχεδιασμό και υπάρχουν διάφορες βαθμίδες πιθανότητων και αντικτύπου, ωστόσο θέλουμε να είμαστε έτοιμοι για το χειρότερο, ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε οτιδήποτε και να συμβεί. Ωστόσο, ό,τι σχεδιασμό και να κάνουμε μπορούμε μόνο να προβλέψουμε μια ε, κάλυψη του κινδύνου στο μέτρο του λογικού. Δεν ε, μπορούμε να είμαστε βέβαιοι 100% και τέλος αυτή η επαναστατική νομοθεσία την οποία εσείς ε, ε, φτιάξετε θα λειτουργήσει μόνο αν όλοι μαζί συνεργαστούμε. Δηλαδή οι νομοθέτης, οι ε, αρμόδιοι για την πολιτική και οι ενδιαφερόμενοι άμεσα φορείς. Εγώ ως διευθυντής του Οργανισμού Χημικών Προϊόντων μπορώ μόνο να σας διαβεβαιώσω ότι εμείς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε από τη δική μας πλευρά για να επιτύχει το ρίτσι. Ξέρουμε ότι οι εταίροι μας προσβλέπουν σε εμά για έναν καλύτερο κόσμο για τις μελλοντικές γενναίες. Σας ευχαριστώ ευχαριστώ για τη συνεργασία σας και προσβλέπω στο διάλογο μεταξύ μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ντανσέτ. Νομίζω ότι έγινε σαφές ότι η υπηρεσία σας έχει τεράστιο έργο σε όλο τον κόσμο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει τόσο προηγμένο σύστημα όσο αυτό της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτό σίγουρα έχουμε ηγετικό ρόλο. Σημαντικό είναι λοιπόν να πετύχει το όλο εγχείρημα. 20 φορές περισσότερες ε, προεγγραφές είχαμε από ό,τι περιμέναμε. Αυτό βέβαια ε, δημιουργεί προβλήματα για το επόμενο στάδιο, ιδιαίτερα όσον αφορά τα λεγόμενα SIFs. Δηλαδή, την έκκληση προς τις εταιρείες να υποβάλουν μαζί με τους ανταγωνιστές τους, ε, τους σχετικούς φακέλους για τις, ε, δραστικές ουσίες, για τις ίδιες δραστικές ουσίες. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε το χρονοδιάγραμμα των επόμενων ετών. Ε, μπορεί ενδεχομένως ε, να ε, αναφερθείτε στο θέμα αυτό αργότερα. Η κυρία Ιούτα και ήρθε ακριβώς τη στιγμή που μιλούσατε για τις δαπάνες και τον προϋπολογισμό. Θα ήταν ενδιαφέρον να ξέρουμε πώς εκτιμάται το σύνολο των τελών που συλλέγεται και την ανάγκη πόρων από τον προϋπολογισμό μας. Όπως ήταν αναμενόμενο, έχουμε έναν μακρύ κατάλογο με ερωτήσεις, έχουμε μία μισή ώρα μέχρι τις πέντε η ώρα. Ο Ρίχαρτ Ζίβαρ είναι ο πρώτος, μετά όλοι με τη σειρά. Ρίχαρτ, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ήθελα να αναφερθώ σε ένα πρόβλημα με την διερμηνία από, την, ε, από το γερμανικό κανάλι έβγαινε άλλη γλώσσα. Μήπως μπορεί ο τεχνικός ε, να το διορθώσει το θέμα αυτό. Μιλάτε πολύ σιγά και γι' αυτό ήταν απαραίτητο να σας παρακολουθώ από τα ακουστικά μου. Αλλά ως προς την ουσία, ευχαριστώ για την παρουσίαση κύριε Διευθυντά. Ήδη αναφερθήκατε στο γεγονός ότι του χρόνου θα μπούμε στη φάση όπου θα έχουμε τις πρώτες προθεσμίες. Ε, η πρώτη είναι 30 Νοεμβρίου 2010 για την καταχώρηση και εάν δεν γίνει η καταχώρηση εγκαίρως δεν θα επιτρέπεται να παράγονται πια οι χημικές ουσίες. Αυτό λοιπόν θα έχει συνέπειες για το σύνολο του τομέα και όπως είπατε αυτά τα ΣΥΦΣ δεν λειτουργούν πολύ καλά. Από ό,τι ξέρω το 1 πέμπτο το, το, 1 πέμπτο ε, των διαδικασιών έχει ολοκληρωθεί σωστά. Τι μπορείτε να κάνετε εσείς για να προωθήσετε το θέμα, ώστε να μην καταλήξουμε στην κατάσταση οι εταιρείε, ιδιαίτερα οι μικρομεσαίες, ε, να μην καταχωρήσουν ε, τα προϊόντα τους εγκαίρως ε, και να μην μπορούν πια να συνεχίσουν την παραγωγή. Μπορείτε Επίσης, να μας πείτε το εξής, από ό,τι ξέρω, από τις πληροφορίες που έχω, 20 ε, φορές περισσότερες ε, καταχωρήσεις ε, έχουν ζητηθεί από ό,τι περιμένατε. Αυτό είναι δικαιολογημένο και μία ερώτηση προς εσάς όσον αφορά το σύνολο της διαδικασίας για να διεξαχθεί ομαλά. Τι προτάσεις έχετε συγκεκριμένα πώς μπορεί καλύτερα να συμμετέχουν οι ενδιαφερόμενοι, οι επιχειρήσεις, η βιομηχανία, ώστε να αποφευθούν ε, ε, αυτά τα προβλήματα, οι καθυστερήσεις, οι συμφορήσεις. Τι μπορεί να γίνει ώστε να αποφευθούν οι δυσάρεστες καταστάσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα ακούσουμε τρεις-τρεις τις ερωτήσεις. Η Λίντα. Ευχαριστώ για την παρουσίασή σας σχετικά με τη λειτουργία της υπηρεσίας. Δύο γρήγορες ερωτήσεις. Η πρώτη, γιατί υποτιμήσαμε τον αριθμό των αιτήσεων σε τέτοιο βαθμό. Είπατε ότι λάβατε 20 φορές περισσότερες. γιατί συνέβη αυτό. Ε, ζητούν καταχώρηση οι, οι επιχειρήσεις που δεν χρειάζεται να το κάνουν. Ε, υπήρχε πρόβλημα στην νομοθεσία. Δεύτερον, υπήρχε η ανησυχία σχετικά με τις δοκιμές σε ζώα. Μπορείτε να αναφερθείτε στο θέμα αυτό. Έχουν βρεθεί λύσεις. Πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα και τι λύσεις μπορούν να βρεθούν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ η Όλγα Κράμερ. Ο κύριος, ε, ε, ε, ο κύριος Χόλκερ Κράμερ. Ευχαριστώ. Είναι πολύπλοκη η νομοθεσία που θα πρέπει να εφαρμοστεί και ήδη συναντούμε μια πρώτη σειρά δυσκολιών. Προσωπικά δεν με εκπλήσουν οι δυσκολίες που συναντούμε. Ήδη κατά τη διάρκεια της νομοθετικής διαδικασίας ε, έγιναν υποδείξεις ε, σχετικά με αυτές. Πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις Πιθανότατα όχι απλά να έχουν δυσκολίες, αλλά να ε, ε, αδυνατούν να εφαρμόσουν την νομοθεσία. Ε, ε όπως και ο κύριος Ρίχαρτ Ζήπερ, θα σας παρακαλούσα να ε, μας απαντήσετε πιο συγκεκριμένα. Καταρχήν, έχετε την εντύπωση ότι οι επιχειρήσεις στην Ευρώπη ασχολούνται με την εφαρμογή του κανονισμού, είναι συνεργάσιμες, πληρούν τις υποχρεώσεις τους. Δεύτερον, όσον αφορά τα ΣΥΦ, συμμερίζεστε τη θέση ότι η διαδικασία για τη δημιουργία τους είναι πιθανότατα υπερβολικά πολύπλοκη και ότι υποτιμήσαμε την όλη κατάσταση. Και η επόμενη μου ερώτηση είναι η εξής να το πω προσεκτικά, είπατε ότι θα έχουμε προβλήματα ως προς το χρονοδιάγραμμα. Μιλήσατε για προτεραιότητες, μιλήσατε για ε, προγράμματα ε, έκτακτης ανάγκης. Τι θα γίνει εάν έχουμε φτάσει στην ε, ημερομηνία της προθεσμίας και δεν έχουν κλείσει οι φάκελοι. Πώς μπορούμε να αντιδράσουμε, τι δυνατότητες έχουμε. Θα ήθελα να μου πείτε πιο συγκεκριμένα και τέλος θα Ήθελα να αναφερθώ στις ε, κατευθυντήρες γραμμές ε, της ε, υπηρεσίας σας. Οι κατευθυντήρες αυτές γραμμές είναι πάνω από χίλιες σελίδες. Μπορούμε πράγματι να απαιτήσουμε από μικρομεσαίες επιχειρήσεις να κάτσουν να τις διαβάσουν. Λειτουργεί αυτό και στην υπηρεσία σας υπάρχουν σχέδια και πόσο συγκεκριμένα είναι αυτά σχετικά με την διαδικασία καταχώρησης, ε, με τη διευκόλυνση της διαδικασίας καταχώρησης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και ε, τελευταία μου πρόταση, ε, όταν θέλει κανεί ε, να έρθει σε επαφή με την υπηρεσία σα, αυτό λειτουργεί μόνο με email. Είναι αδύνατο να σου πάρουν τηλέφωνο ε, και ε, καθυστερεί πάρα πολύ απάντηση στα email και όταν την λάβουν οι επιχειρήσει δεν είναι ικανοποιητική. Νομίζω ότι έχουμε μπροστά μα πολλή δουλειά. Θα ήθελα να μου πείτε πόσο κρίσιμη είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Περιμένουμε τις απαντήσεις σας. Ευχαριστώ. Να ξεκινήσω με τις ερωτήσεις του κυρίου Ζήπερ. Πράγματι, είναι αλήθεια ότι το REACH λέει εάν δεν υπάρχουν δεδομένα δεν υπάρχει αγορά. Δηλαδή οι επιχειρήσεις θα πρέπει να καταχωρήσουν τα προϊόντα τους εγκαίρως ώστε να έχουν τη δυνατότητα να παραμείνουν στην αγορά. Οι αρχές επιβολής ε, του νόμου των κρατών μελών θα πρέπει να φροντίσουν μόνο οι ε, επιχειρήσεις που έχουν καταχωρήσει τα προϊόντα τους να παραμείνουν στην αγορά. Αυτό δεν είναι καθήκον της, ε, της υπηρεσίας μας. Ένα στοιχείο της απάντησής μου λοιπόν... Μπορούμε όλοι να είμαστε ικανοποιημένη εάν στο τέλος της διαδικασίας γίνει παράταση της ε, πρώτης προθεσμίας ε, κατά έξι μήνες. Το εξάμεινο αυτό που παρήχανε οι νομοθέτες, εσείς και το Συμβούλιο δηλαδή, ε, αυτούς τους έξι μήνες τους χρησιμοποίησε η βιομηχανία για να καταλάβει πώς ακριβώς θα πρέπει να διαμορφώσει τα ΣΥΦ. Αυτή η προθεσμία δόθηκε δηλαδή, διότι πολλή ε, χρόνος έχει χαθεί ε, ε, για να βρεθεί η σωστή διαδικασία, διότι οι κατευθυντήρες γραμμές δεν εξηγούσαν επαρκώς πώς θα έπρεπε να γίνει κάτι τέτοιο. Και τελικά, στην πραγματικότητα, έχουμε δει πολλούς, δυνατούς, πολλούς πιθανούς τρόπους ε, λειτουργίας των ε, ΣΥΦ. Χρειάστηκε λοιπόν πολύς χρόνο ε, για να καταλάβουν επιχειρήσει τι πρέπει ακριβώ να κάνουν. Και έτσι επανέρχομαι στην ερώτηση όχι μόνο στη δική σα αλλά και σε άλλων. Υπάρχει ακόμα αρκετό χρόνο για ολοκλήρωση των φακέλων των αιτήσεων. Η γνώμη μου είναι ότι ναι, αρκεί ο χρόνος. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να χαθεί βέβαια πολύς χρόνος και μάλλον θα πρέπει να καταβάλουμε προσπάθειες ώστε να ανακτηθεί μέρος του χαμένου χρόνου. Και πώς μπορεί να γίνει αυτό. Νομίζω ότι αυτό ήδη το κάνουμε με διάφορους τρόπους. Οργανώσαμε σχετικό εργαστήριο, σεμινάριο, ε, οργανώνουμε όμως και σεμινάρια μέσω του διαδικτύου όπου εξηγούμε ακριβώς τις διάφορες διαδικασίες που πρέπει να πραγματοποιηθούν για να γίνει η καταχώρηση. Δηλαδή, καταρχήν μιλάμε για τον εντοπισμό των ε, ουσιών, ε, την ε, συμφωνία πάνω σε έναν ορισμό, το το πείρασμα των πληροφοριών καθώς και τις ε, απαιτήσει από την ε, διαδικασία πληροφόρησης. Δεύτερον, έχουμε σχεδιάσει άλλο ένα μέσο πληροφορικής, το οποίο δεν ζητήθηκε, αλλά είναι ένα chat box. Ε, ουσιαστικά θα πρέπει οι επιχειρήσεις να συνομιλούν μεταξύ τους. Δεν θα πρέπει να επανεφεύρει κανείς ε, τον τροχό και εμείς έτσι δημιουργήσαμε την υπηρεσία μας. Ε, μάθαμε από άλλες υπηρεσίες και γι' αυτό φτάσαμε εδώ που φτάσαμε τόσο γρήγορα. Το ίδιο λοιπόν μπορούν να κάνουν και άλλοι. Κάποιοι ηγούνται, κάποιοι βρίσκονται πιο μπροστά, γιατί λοιπόν να μην βοηθήσουν τους άλλους. Και αυτός ήταν ε, ο στόχος του εργαστηρίου LEAD καθώς και της αίτησή μας, ώστε να μπορεί δηλαδή ο ένας να θέτει ερωτήσεις στον άλλον. Μπορούμε να κάνουμε κάτι περισσότερο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, συνήθως ε, δεν είναι ο κύριος καταχωρητής, ο κύριος ετών της καταχώρησης, ε, συμμετέχουν στην διαδικασία και θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα που συντάσσουν οι μεγάλες επιχειρήσεις. Ε, το θέμα είναι λοιπόν να υπάρχουν δίκαιοι κανόνες και η καθοδήγηση για ε, την ε, για την ανταλλαγή πληροφοριών προβλέπει έναν τρόπο πώς μπορεί να γίνει αυτό. Θα πρέπει οι διάφοροι όμιλοι, οι διάφορες κοινοπραξίες να δημοσιοποιήσουν τους υπολείπους τα αποτελέσματα της δουλειάς τους. Νομίζω ότι κάτι τέτοιο θα μας οδηγήσει σε καλά αποτελέσματα στο μέλλον. Μετά από την πρώτη προθεσμία, μετά από την προθεσμία για την πρώτη καταχώρηση, θα πρέπει να εξετάσουμε πώς θα οργανώσουμε το σύστημα στο μέλλον. Διότι όσο μικρότερος ο όγκος, ε, διότι όσο προχωράει ο χρόνο, τόσο περισσότερε μικρομεσαίε επιχειρήσει θα συμμετέχουν στη διαδικασία και θα πρέπει να ηγηθούν τη διαδικασία. Γι' αυτό θα θέλαμε στο μέλλον να δώσουμε περισσότερη υποστήριξη στη διαδικασία αυτή. Θα πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε δημιουργικά για το πώς μπορούμε να ε, παρέχουμε τέτοιου είδους υποστήριξη. Και αυτό με οδηγεί στην ερώτηση του κυρίου Κράμερ σχετικά με τον προσανατολισμό που δίνουμε. Είναι όσο γίνεται πιο πλήρης και γι' αυτό έχει τόσο μεγάλο όγκο. Δεν χρειάζεται όμως όλοι να διαβάσουν το σύνολο του οδηγού. Χρειάζεται να διαβάσει ο καθένας το κομμάτι του οδηγού που αφορά ένα συγκεκριμένο φάκελο και γι' αυτό ακριβώς ο οδηγός αυτός, το εγχειρίδιο αυτό, παραπέμπει τον αναγνώστη στα σημεία που τον ενδιαφέρουν περισσότερο που ενδιαφέρουν περισσότερο την επιχείρησή του δηλαδή ή το συγκεκριμένο ΣΥΦ. Οι πληροφορίες είναι επίσης πιο εύκολα προσβάσιμες επειδή έχουμε δώσει μια περίληψη του οδηγού Έχουμε επίσης συντάξει κάποια φυλάδια πληροφόρησης. Έχουμε δηλαδή δημιουργήσει κάποια εργαλεία που κάνουν τις πληροφορίες πιο προσβάσιμες, ώστε οι επιχειρήσεις να μπορούν να καταλάβουν τι ακριβώς χρειάζονται. Πρόκειται για ένα μενού κατά κάποιο τρόπο. Δεν χρειάζεται να φάει κανείς όλα τα φαγητά στο μενού, θα αρρωστήσει κανείς. Αν τα φάει όλα. Μπορούν, μπορούν λοιπόν οι επιχειρήσεις να επιλέξουν κάποια σημεία από το μενού. Να επανέλθω στις, ε, αιτήσεις, ε, στις προκατακτικές αιτήσει καταχώρησης, οι οποίες ήταν 20 φορές περισσότερες από όσες περιμέναμε. Υπήρχαν πολλοί λόγοι γιατί είχαμε τόσο πολλές αιτήσει. Κάποιες επιχειρήσεις δεν χρειαζόταν να καταχωρήσουν τα προϊόντα τους. Ε, θεώρησαν όμως ότι θα μπορούν να βγάλουν λεφτά πολλώντας, πολλώντας καταχωρήσεις ε, σε άλλους. Κάποιες επιχείρησεις λοιπόν προσπάθησαν να υποφεληθούν από το σύστημα αυτό, δημιουργώντας διάφορες εταιρείες εντός του συστήματος πληροφορικής μας για όσο γίνεται περισσότερες ουσίες. Δεν είναι δυνατόν όμως να ε, μεταβιβαστεί η καταχώρηση από μία εταιρεία σε άλλη. Οι επιχειρήσεις αυτές λοιπόν παρεξήγησαν το όλο σύστημα. Επίσης, σε κάποιες περιπτώσεις η νομοθεσία προέβλεπε ανάγκη για διπλή προκαταχώρηση, προκαταρκτική καταχώρηση, όπως για παράδειγμα για κάποιους τομείς της βιομηχανίας, Χρειαζόταν λοιπόν σε κάποιες περιπτώσεις για μία ουσία δύο επιχειρήσεις να κάνουν την προκαταθήκη ε, καταχώρηση. Ε, τελικά όμως ε, θα καταλήξουμε σε μία αίτηση αναπροϊόν για κάθε αλυσίδα προμήθειας. Επίσης κάποιες επιχειρήσεις έλεγαν ότι εμείς εμπορευόμαστε πολλά μείγματα και δεν ξέρουμε ποιες ουσίες περιέχονται σε ποιο μείγμα. Για να είμαστε λοιπόν ασφαλείς, ας τα καταχωρήσουμε όλα. Και βέβαια τελικά δεν θα γίνει καταχώρηση για όλες τις ουσίες αυτές, αλλά οι προκαταρκτικές καταχωρήσεις ήταν δωρεάν. Όταν λοιπόν παρέχει κανείς μια τόσο εύκριστη υπηρεσία δωρεάν, τελικά καταλήγει σε πολύ περισσότερες αιτήσει από ό,τι χρειάζονται. Όταν λοιπόν εξετάσαμε όλες τις πληροφορίες, όταν εξετάσαμε όλο το υλικό και όταν Προσπαθήσαμε να δούμε πόσε αιτήσει θα έχουμε το 2010 και είδαμε ότι θα είναι περισσότερε και ότι θα είναι πολύ περισσότεροι οι φάκελοι. Αρχίσαμε να διαγράφουμε ό,τι δεν ήταν απαραίτητο, ό,τι δεν ήταν χρήσιμο. Καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι δεν θα καταχωρηθούν μέχρι το 2010 περισσότερες ουσίες από ό,τι ήταν η αρχική μας εκτίμηση. Το... Μιλάμε για περίπου 9.000 ουσίες. Αυτό όσον αφορά και την ενδιάμεση και την τελική καταχώρηση. Μπορεί και να υπάρχουν κάποιε επικαλύψει. Όσον αφορά του φακέλου, η Κομισιόν έκανε υπολογισμό για 25.000 το 2010. Αυτή τη στιγμή έχουμε διατηρήσει αυτόν τον αριθμό φακέλων, δεδομένου ότι είχαμε μια καθυστέρηση στην ε, διαδικασία, αλλά θα δείτε ότι στο πρόγραμμα εργασίας μας για το 2010 έχουμε και ένα σενάριο για 50.000 φακέλους καθώς και ένα για 75.000 ε, φακέλους. Έχουμε δηλαδή τρία σενάρια και προσπαθούμε να, εντοπίσουμε τους, ε, να υπολογίσουμε τους πόρους που χρειαζόμαστε για κάθε τέτοιο σενάριο ώστε να ενεργήσουμε ανάλογα. Έτσι λοιπόν λειτουργούν τα σενάρια μας. Και νομίζω ότι έτσι απαντώ στον κύριο Κράμερ. Όσον αφορά τα σενάρια αυτά, Θα θυμάστε ότι και κατά διάρκεια τη προκαταρκτική καταχώρηση όλοι ήθελαν να έχουμε ένα δεύτερο σύστημα πληροφορική σε περίπτωση ε, που, ε, που χαλάσει το δικό μα. Ε, θέλαμε δηλαδή ένα δίκτυο ασφαλεία. Έτσι λοιπόν και τώρα θα αναπτύξουμε ένα εναλλακτικό σύστημα Σε περίπτωση λοιπόν ε, που δεν λειτουργεί το δικό μας σύστημα θα έχουμε έναν άλλον τρόπο να ε, διαχειριστούμε τους φακέλους αυτούς. Αυτό θα στοιχήσει πόρους και όσον αφορά το ανθρώπινο δυναμικό και όσον αφορά τα χρήματα. Θα Πρέπει όμω να είμαστε έτοιμοι δεδομένου ότι η νομοθεσία καθορίζει πολύ συγκεκριμένα τι προθεσμίε. Και να αναφερθώ και στι δοκιμέ σε ζώα, στα πειράματα σε ζώα. Θα θέλαμε καταρχήν να επιβεβαιώσουμε ότι σε αντίθεση με ό,τι δημοσιεύθηκε σε κάποιες επιστημονικές εφημερίδες, σε κάποια επιστημονικά περιοδικά, συνεχίζουμε να πιστεύουμε ότι δεν θα χρειαστεί να γίνουν περισσότερες δοκιμές σε ζώα από ό,τι εκτιμήθηκε κατά την έγκριση της νομοθεσίας. Έχουμε δημοσιεύσει ένα ανακοινωθέν τύπου, όπου εξηγούμε γιατί δεν θα ξεπεράσουμε τις αρχικές εκτιμήσεις. Ταυτόχρονα, προωθούμε ενελεκτικούς τρόπους δοκιμών. Και γι' αυτό μία πτυχή της εργασίας μας είναι να εξηγήσουμε στην βιομηχανία πώς μπορεί να αποφύγει νέες δοκιμές σε ζώα. Θα πρέπει δηλαδή να γίνει ευρύτερη χρήση των ε, δεδομένων που ήδη υπάρχουν. Στο παράθυμα 11 αναφέρονται και εναλλακτικοί τρόποι. Έξυπνη χρήση των δεδομένων που υπάρχουν μπορούν να οδηγήσουν σε αποφυγή δοκιμών σε ζώα. Από την ιστοσελίδα μας και από τα ανακοινοθέντα τύπου μας μπορείτε να δείτε ότι όταν μια επιχείρηση προτείνει παρόλα αυτά να να κάνει αίτηση για δοκιμές. Ε, έχουμε πρώτα διαβουλεύσεις με το κοινό προτού εγκρίνουμε αυτές τις νέες δοκιμές σε ζώα που έχουν ζητηθεί. Χρησιμοποιούμε λοιπόν τα εχέγγυα που έχετε εγκρίνει στην ομοθεσία. Νομίζω λοιπόν ότι και εδώ είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μάρτιν Κάλ. Επόμενος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον κύριο Ντάνσερτ για την παρουσίασή του και τις τόσο ενδιαφέρουσες απαντήσεις του μέχρι στιγμής. Πήγα και επισκέφθηκα μια μικρή χημική, μικρομεσαία επιχείρηση στην περιοχή μου την περασμένη εβδομάδα. Είναι πολύ εξειδικευμένη στη βιομηχανία πετρελοειδών, παράγουν ουσίες που οι περισσότερες εξάγονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μου λένε εκατοντάδε χιλιάδε σερλίνες θα τους κοστίσει για να καταχωρήσουν την ουσία αυτή. Έχουν και πολλούς ανταγωνιστές οι οποίοι δρεύουν όλοι εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό σημαίνει ε, πολλά έτη κερδών που θα πρέπει να χρησιάσουν και με την ε, τρέχουσα οικονομική τους κατάσταση. Τι τους συμβουλεύετε, είναι σε πολύ δεινή οικονομική θέση, δεν έχουν τα χρήματα να καταχωρήσουν αυτή την ουσία που είναι τελείως ε, ε ασφαλής, έτσι κι αλλιώς αυτό θα φανεί από την καταχώρηση. Όμως οι ανταγωνιστές, επαναλαμβάνω, δεν επομίζονται τέτοιο κόστος και έχουν και τους ίδιους Πελάτε. Είναι πολύ δύσκολο το δίλημά του. Εσείς τι του συμβουλεύετε. Ευχαριστώ. Καρλ Σλίτερ. Ευχαριστώ. Χαιρετίσματα από τη Σάτου Χάση. Δυστυχώς σήμερα κολλείται και αποσιάζει. Για τους ανθρωπίνους πόρους. Το 2010 λέτε θέλετε 100 νέους υπαλλήλους. Πόσοι από όλους αυτούς θα κάνουν αξιολόγηση για εκτίμηση, πόσοι θα είναι οι επιστημονικοί συνεργάτες και επιρρογνώμονες για να εγκρίνουν τα πειράματα και να τα ελέγχουν. Πόσοι άνθρωποι σας χρειάζεται για να κάνουν αυτή τη δουλειά. Νομίζω ότι εμεί αυξήσαμε τον προπολογισμό στην ψηφοφορία. Θα με διορθώσει η Γιούτα Χάουκ. Ε, πείτε μας αν θέλετε περισσότερα χρήματα. Υποθέτω ότι έχετε υποχρηματοδότηση μέχρι να αρχίσετε να εισπράτετε από τα τέλη, αλλά θα είναι πολύ αργά για τη στελέχωσή σας. Αυτό μπορείτε να μας απαντήσετε. Το δεύτερο, για τη λίστα υποψηφίων. 15 ουσίες ε, αναφέρατε, ενώ υπάρχουν χιλιάδες ουσιών. Είναι πολύ σημαντικό για τους πολίτες ε, να ξέρουν, για να ενημερώνονται, να υπάρχουν πολλές ουσίες στις υποψήφιες προς έγκριση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε πέντε και μία μόνο κατέληξε σε αυτό τον κατάλογο. Μα υπάρχουν τέσσερις ψυχρές πίσες, ε, λεγόμενες κόλταρς, που ε, ανταποκρίνονται ε, στα κριτήρια. Αν δεν δίνει αρκετή ενημέρωση ο κλάδος, η βιομηχανία για να αποφασίσετε, να τους υποχρεώσετε. Δεν θα πρέπει να επιβραβεύεται η βιομηχανία όταν δεν σας ενημερώνει σωστά για να κάνετε καλά τη δουλειά σας. Αναφερθήκατε και στις 7 ουσίες που προτείνετε. Ε, τρεις είναι φθαλικές ουσίες και μια άλλη επίσης επισφαλής. Τον Ιούνιο δεν αποφασίσατε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν επανήλθε. Στο ΡΙΤ, στον κανονισμό, έχετε εσείς προθεσμία για να αντιδράσετε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όχι. Τι προτείνετε και πότε ε, που αναμένεται η απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής γιατί έχουν αρχίσει να συζητάνε αυτό το καθοδηγητικό έγγραφο ε, το 2007. Πώς μπορούμε να επιταχύνουμε αυτή τη διαδικασία και πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε. Την περασμένη φορά ε, στη συνεδρία της Επιτροπής μας μίλησα για κριτήρια PBT και άλλων ουσιών και έφερα σε δύσκολη θέση την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί είπατε και εσείς και τα κρατημέλια ότι χρειάζεται καλύτερη πληροφόρηση για τα κριτήρια και Μιλάμε και για ε, οργανισμούς υδρόβιους, αλλά θα πρέπει ε, να μιλήσουμε και για αερόβιους οργανισμούς. Τι είναι όλα αυτά τα κριτήρια, πώς μπορούν να ε, αναθεωρηθούν, που πρέπει να αναθεωρηθούν το σύντομότερο. Αυτά προς το παρόν. Πολλές ερωτήσεις κάνετε, λέει ο πρόεδρος. Τώρα, ο Ζήλ Περνιό. Δύο λόγια μόνο. Έχουν γίνει πολλές ερωτήσεις ήδη και πολλά θέματα θίξαν. Στην εισαγωγή σας είπατε ότι ήταν το μωρό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το ΡΙΤΣ. Και εσείς πολύ καλή μεμπισίτερ είστε. Έχω την εντύπωση ότι η θελησιοκρατία σας δεν είναι αρκετή. Δεν είστε καλή νταντά. Δεν φροντίζετε καλά το μωρό μας παρόλη τη βούληση που εκφράσατε προηγουμένως. Γιατί ακούμε την Ένωση Χημικών Βιομηχανιών που λέει ε, ότι δεν γίνεται 1500 ε, 1.500 φάκελοι έχουν, εγκριθεί, έχουν καταχωρηθεί και 9.000 ε, ε, ε, θα έπρεπε. Εκκρεμούν πάρα πολύ, δηλαδή διαμαρτύρονται και μας φέρουν μπροστά σε τελεσμένα γεγονότα. Γιατί η διελκυστίδα αυτή είναι υπέρ εκείνων. Εγώ θα επιθυμούσα, ε, βγαίνοντας από εδώ, να μας πείτε ποιες είναι οι σημαντικές διατάξεις ε, και τα μέτρα που θέλετε να λάβετε και να εφαρμόσετε. Για παράδειγμα, σε μία από τις απαντήσεις σας είδαμε το πρόβλημα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Μας λέγουν ότι οι μικρομεσαίες δεν μπορούν να καταχωρήσουν τις ουσίες τους γιατί είναι πάρα πολύ περίπλοκο οι διαδικασίε και οι φάκελοι. Και εσεί μα είπατε ότι μπορούν να έρθουν σε επαφή με τι μεγάλε χημικέ βιομηχανίε που μπορούν να τι βοηθήσουν. Ναι, αλλά αν έχετε αυτή την πληροφόρηση, τι λένε οι μεγάλες χημικές βιομηχανίες. Αν δεν γίνεται οι να μπορέσουν να αντιδράσουν, μα τότε θα πρέπει ο οργανισμός να ασχολείται. Και με τρόπο έτσι πιο συγκεκριμένο να υποδεικνύει στις μικρές επιχειρήσεις ε, ποια είναι τα στοιχεία που θα πρέπει να καταχωρούν. Όπως προηγουμένως ε, θύμισε ο συνάδελφος Σλούτερ. Θα μπορούσατε λοιπόν ενδεχομένω να μας πείτε ποια θα είναι τα ε, μέτρα, τα υποχρεωτικά, αγκαστικά ε, για να υποχρεώνετε ε, ε, τις εταιρείες να σας ενημερώνουν, που είναι και υπερημών με Y και υπερημών με Ήτα. Ο Καλ Χάινς Φλόρενς. Μάλιστα. Κύριε Γενικέ, Διευθυντά, εάν σας κατάλαβα καλά, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις φταίνε για όλα. Και ο οργανισμός σας θα έχει κάνει όλα σωστά. Ε, δύσκολα μπορώ αυτό να το πουλήσω στην ιδιαίτερη πατρίδα μου, γιατί άλλα ακούω από τους μικρομεσαίους. Και ο συνάδελφος να έχει δίκιο. Όταν λέγει ότι το σύστημα στην Ευρώπη ε, είναι πολύ φιλόδοξο, αυτό που στήσαμε, γνωρίζοντας όμως ότι θα έχουμε ενδεχομένως στρεβλώσεις του ανταγωνισμού. Αλλά από ό,τι φαίνεται, μερικοί το έχουν ήδη ξεχάσει αυτό. Βεβαίως και θέλουμε την καταχώρηση αυτή και δεν το αμφισβητώ, αλλά δεν μπορούν να είναι τόσο δαπανηρά όλα αυτά και όσο περίπλοκα και τόσο χρονοβόρα για λόγους γραφειοκρατικούς. Αν θέλετε 1100 σελίδες για να περιγράψετε και μόνο τον οργανισμό σας, ε, αυτό δεν εντάσσεται στη Λισαβόνα, ας πούμε. Μπορεί να εντάσσεται σε έναν οργανισμό που λειτουργεί καλά, αλλά είπαμε ότι θέλουμε να κάνουμε την Ευρώπη τι είναι ισχυρότερη ήπειρο του κόσμου κτλ. Ε, πιστεύω λοιπόν ότι τα εμπόδια που υπάρχουν τώρα θα πρέπει κάπου να οφείλονται. Αν δεν έρχονται οι επιχειρήσεις ή αν δεν μπορούν να προχωρήσουν, ε, υπάρχει κάποιος λόγος. Είτε δεν μπορούν να δώσουν τα στοιχεία, είτε φοβούνται. Μπορώ να τους καταλάβω. Όταν κάποιος μικρός και έχει 100 εργαζομένους και πολύ υψηλή πνευματική ιδιοκτησία, ε, δεν πάει να την καταθέσει κάπου χαίρεται δεν είναι μόνο ε, βασικές ουσίες, πρώτες αλλά είναι πολύ περίπλοκες ε, ουσίες, τις οποίες βασίζεται καμιά φορά η ύπαρξη ολόκληρης της Ε, από ό,τι φαίνεται δεν προχωράει αυτή η υπόθεση. Ε, τα στοιχεία είναι πάρα πολύ ε, διεισδυτικά αυτά που ζητάτε και παραβιάζουν ε, την έννοια της πνευματικής ιδιοκτησίας. Εκεί θα ήμουν πάρα πολύ προσεκτικός εγώ. Ο Χόρστ Σνέλχαρτ. Ευχαριστώ. Είχα αρχίσει να ανησυχώ. Γιατί δεν είχα καταλάβει τι σειρά είχα και με ποια σειρά δίνεται το λόγο. Αλλά δεν πειράζει, εσύ είναι. Ο ένας μετά τον άλλον λέει η σειρά, <laughs> λέει ο πρόεδρος. Ευχαριστώ για την ενημέρωση. Νομίζω ότι έχει γίνει σαφές το εξή. Ε, πάει καλά ε, ο οργανισμός ε, στο αρχικό του στάδιο, αλλά εκπλήσωμε ε, για αυτά που λέτε. Ε, λέτε ότι έχετε σχέδια, δεν ξέρετε πόσες αιτήσει θα πάρετε, τι θα κατατεθεί και λέτε δεν δούμε περισσότερο χρόνο, θα προλάβουμε. Μπράβο για το θάρρος σας. Αλλά ε, Μήπω χρειάζεται και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινοβούλιο ένα σχέδιο έκτακτη ανάγκη για να επιμηκυνθεί κάπω ο χρόνο, να δοθεί κάποια παράταση, γιατί προέχει η ποιότητα τη ταχύτητα, Χρειαζόμαστε σαφή δεδομένα, σαφεί δεσμεύσει και υποδείξει. Και δεν νομίζω ότι θα μας φτάσει ο χρόνο ακριβώ, γιατί το ακούσαμε επανελειμμένα σήμερα, η συνεργασία, οι δυσκολίε, οι επιφυλάξει που μπορεί να έχουν μικρομεσαίε επιχειρήσει είναι δεδομένε. Ακούω πολύ συγκεκριμένα πράγματα από τον κόσμο που λέει μόνο στα αγγλικά μας στέλνουν τους φακέλους. Και θα πρέπει να τα δώσουμε να μεταφραστούν. Δηλαδή κάθε μικρομεσαία επιχείρηση, αν δεν έχει ένα συνεργάτη αγγλόφωνο που μπορεί να τα ανταλλάσσει, πρέπει να μεταφράζει όλα αυτά τα χαρτιά, επιπλέον κόστος κτλ. Δεν θα μπορούσαμε... Το είπατε κι εσείς προηγουμένως σε όλες τις επίσημες γλώσσες να μεταφράζεται, να εφαρμόζεται και αυτό, γιατί είμαι πεπισμένος ότι δεν γίνεται αυτό. Σε πολλές περιπτώσεις δεν αποστέλλονται στη γλώσσα των ενδιαφερομένων τα έγγραφα και οι φάκελοι. Οπότε θα παρακαλούσα εκεί να δώσετε μεγαλύτερη προσοχή, να διευκολύνετε τη δουλειά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Γι' αυτό θα βοηθήσει να τηρούνται και οι προθεσμίες. Αλλιώς Νομίζω θα πρέπει να έχουν και ένα σχέδιο εκτακτή ανάγκη και το Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μπορείτε να με διαψεύσετε, εγώ το σημειώνω, αλλά θα το παρακολουθήσω. Αλλιώ δεν θα προκάνομαι, λέω εγώ. Ευχαριστώ. Ο κύριο Ντάνσερτ. Okay, thank Σας ευχαριστώ. Να ξεκινήσω με το πρώτο συγκεκριμένο παράδειγμα του κύριου Κόλεγκαν για τη μικρο, αυτή μικρομεσαία που παράγει μία μόνο ουσία σε έναν, μία παγκοσμιοποιημένη αγορά στην πετρελοβιομηχανία. μηχανία. Όντως πρόκειται για μια παγκόσμια αγορά, όπου όμως η Ευρώπη είναι μέρος της ε, και όλες οι άλλες εταιρείε θα έπρεπε να εγγραφούν που ε, λειτουργούν στην ίδια αγορά. Αφού κάτι τέτοιο φαντάζομαι. Οπότε θα πρέπει να υπάρχει κάποιος καταμερισμός του κόστους και συνεργασία, εκτός και αν η αγορά είναι τόσο ειδική Εσείς λέτε πως δεν υπάρχει αγορά για την ουσία αυτή στην Ευρώπη. Λέτε πως εξάγεται το 99% του προϊόντος. Αλλά αν το 1% είναι απαραίτητο, στην Ευρώπη θα μπορούσε αυτό να είναι ένα θέμα. Αλλά πάντως μπορούμε αυτό να το εξετάσουμε, τη συγκεκριμένη περίπτωση. Εν γέννη, όσον αφορά τη στήριξη των μικρομεσαίων, θέλω να πω ότι οι μικρομεσαίες ε, δεν, είναι, δεν έρχονται μεμονωμένα και δεν καταχωρούνται μεμονωμένα. Εάν είναι επικεφαλής της καταχώρησης, η συμφωνία μας με τις Εθνικά Γραφεία Βοήθειας είναι ότι θα πρέπει εκείνοι να αναλάβουν, μιλούν τη δική τους γλώσσα, εμείς τους βοηθούμε, εμείς τους καταρτίζουμε και μπορούν να τους βοηθήσουν το Εθνικό Γραφείο και για τη χρήση του συγκεκριμένου τύπου πληροφορικής με όλα τα εργαλεία που έχουμε σε όλες τις γλώσσες και αυτό είναι κάτι που θέλω να τονίσω ότι προσπαθούμε να μεταφράσουμε όσο γίνεται περισσότερα από τα έγγραφα επίσης τους επόμενους μήνες θα μεταφράσουμε τα περισσότερά μας εγχειρίδια τα οποία ε, είναι προσανατολισμένα στην ε, χρήση της πληροφορικής και μπορεί να είναι και αυτά βοηθητικά. Επίσης ξέχασα να μιλήσω για το πώς ερχόμαστε σε επαφή με τις εταιρείε που έχουν πρόβλημα. Από τα μέσα του έτους, εμείς ερχόμαστε σε επαφή με κάθε εταιρεία που έχει πρόβλημα στην υποβολή κάποιου ε, φακέλου. Τους καλούμε άμεσα και μπορείτε να έρθετε σε επαφή με εταιρείε που έχουν ήδη υποβάλει ε, ντοσχέ και έχουν κάπου ε, σταματήσει στην πορεία. Εμείς τους καλούμε. Και είναι πολύ θετική για τον τρόπο με τον οποίο ερχόμαστε σε επαφή μαζί τους. Πιστεύω πως και αυτό είναι ένα συν. Όσον αφορά την στελέχωση του οργανισμού, έχουμε 100 νέα στελέχη και από όσο θυμάμαι είναι 25 εξ αυτών, ένα τέταρτο δηλαδή θα ασχοληθεί με την αξιολόγηση το 2010, όμως θα πρέπει να καταλάβετε επίσης ότι άλλα 15 με 20 άτομα θα ασχοληθούν πρώτα με την καταχώρηση και τον επόμενο χρόνο θα πάνε στην αξιολόγηση. Άρα τον επόμενο χρόνο θα καταρτιστούν εν μέρη για την εργασία αξιολόγηση. Είναι άνθρωποι που ε, προσωρινά θα μας βοηθήσουν στην καταχώρηση και τον επόμενο χρόνο θα προχωρήσουν στην αξιολόγηση. Που θα είναι ο μεγαλύτερος όγκος εργασίας από το 2011 και μετά. Οπότε πιστεύω πως αυτή την πτυχή της αξιολόγησης ε, την αντιμετωπίζουμε έτσι. Φυσικά, όπως σας είπα, οι πόροι ξεκολουθούν να μας ενησυχούν και θα σας ενημερώνουμε βέβαια, αλλά φυσικά εργαζόμαστε ώστε να κάνουμε πιο ακριβείς υπολογισμούς ε, και σίγουρα η Γενική Διεύθυνση που είναι υπεύθυνη για μας μας παρακολουθεί μηνιαίως για να δούμε πόσα χρήματα θα χρειαστούν ε, για τον επόμενο χρόνο και πόσα έσοδο θα έχουμε για να μπορέσουμε να χρηματοδοτήσουμε το κόσμο γιατί είναι πραγματικά απρόβλεπτο το πότε ακριβώς θα αρχίσουν οι πληρωτές καταχωρήσεις. Αυτή τη στιγμή συζητάμε για ακόμα 15 ουσίες τώρα στον κατάλογο για τη σχετική ερώτηση των ουσιών. Έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε περισσότερα στο μέλλον, αλλά τα όσα έχουμε κάνει για να επιταχύνουμε αυτή τη διαδικασία νομίζω ότι διευκόλυναν τη συζήτηση ανάμεσα στους υπεύθυνους για τη, λήψη των, ε, για τη χάραξη πολιτικής, τα κάτι μέλη και την Κομισιόν για το πώς θα καταμεριστεί η εργασία μεταξύ τους για την προετοιμασία των ντοσιέ ε, για την λίστα των υποψηφίων. Έχουμε κάνει νομίζω ένα μεγάλο βήμα στη διευκόλυνση της πολιτικής συζήτησης και έτσι ώστε να γίνεται καλύτερος καταμερισμός εργασίας στο μέλλον. Αυτή ήταν η φετινή μας ε, συμβολή. Το τέταρτο τρίμηνο δεν τα καταφέραμε γιατί δεν είχαμε αρκετές πληροφορίες από τον ε, κλάδο για την ταυτότητα των ουσιών, για να μπορέσουμε δηλαδή να εντοπίσουμε σωστά την ουσία, αλλά και για την χρήση και την έκθεση στις ουσίες. Πρόκειται όμως απλά για μια καθυστέρηση. Ε, θα, θα καταχωρηθούν αυτά έτσι και λίγο στον επόμενο χρόνο και πρόκειται απλώς για μια μικρή καθυστέρηση. Δεν κερδίζουν δηλαδή και τίποτα αλλά για μας είναι εξαιρετικά σημαντικό να τοποθετηθούν οι σωστές ουσίες, να έχουμε σωστή αναγνώριση της ουσίας ε, όταν μπαίνει στο λίστα, να μην υπάρχει αμφισβήτηση για το κατά πόσο σωστά έχουμε ορίσει την κάθε ουσία. Όσον αφορά τις οδηγίες για την διοδότηση. Η διαδικασία της Κομισιόν για την πρώτη εκδοχή του καταλόγου αδειοδότησης αδειοδοτήσεων μάλλον, θα πρέπει να ε, ρωτήσουμε ακριβώς γιατί υπάρχουν καθυστερήσεις στην Κομισιόν. Εμείς ε, τις επιθυμούμε ακόμη περισσότερο από ό,τι εσείς διότι χρειάζεται να επεξεργαστούμε τις διαδικασίες και πιέζουμε όσο μπορούμε ώστε να επιταχύνουμε την ολοκλήρωση των ε, οδηγιών. Ελπίζουμε πως θα έχει ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία μέχρι το Φεβρουάριο του επόμενου έτους και όσον αφορά τα κριτήρια του BBT, εμείς λαμβάνουμε τα μέτρα ώστε να δημιουργήσουμε μια επιστημονική ομάδα μέσα στο πλαίσιο των επιστημονικών μας επιτροπών για το θέμα αυτό και πάλι θα κάνουμε το δικό μας μερίδιο σε αυτό το πλαίσιο, μερίδιο εργασίας σε αυτό το πλαίσιο. Γιατί τώρα έχουμε 1500, ε, ενώ έπρεπε να είχαμε 2000 και ενώ προβλέπονταν 9000 ε, αρχικές καταχωρήσεις. Αυτό δεν οφείλεται στο ότι υπάρχουν μόνο 9000 ΣΥΦ ε, που έχουν δραστηριοποιηθεί. Υπάρχουν πολλά περισσότερα. Όμως, δουλεύουν μόνο με ένα υποσύνολο των ανθρώπων που έχουν καταχωρηθεί. Δεν υπάρχει μία ε, ε, δεν, δεν έχει γίνει ακόμα επισήμως ορισμός του υπεύθυνου για την καταχώρηση και άρα δεν έχει επισήμως δημιουργηθεί το ε, ΣΥΠ. Σε άλλες περιπτώσεις έχει να κάνει με το γεγονός ότι η Ένωση, η, και αυτό ισχύει για την πετρελαιομηχανία ότι εκείνοι κάνουν την περισσότερη δουλειά για να προετοιμάσουν τα ντοσιέ, αλλά δεν έχουν αναθέσει τα διάφορα ε, ντοσιέ στους υπεύθυνους καταχώρησης. Δηλαδή το υπάρχει, αλλά ο υπεύθυνο καταχώρηση δεν υπάρχει, δεν έχει οριστεί. Έχουμε συμφωνήσει μαζί με την Επιτροπή να ενημερώσουμε όλους ε, τις ενώσεις που εργάζονται για τα ΣΥΦ ώστε να ολοκληρώσουν τον ορισμό του υπευθύνου και να μπορέσουν έτσι και άλλες εταιρείε να μπουν σε αυτά τα κονσόρσια της συμπράξης, ώστε να γνωρίζουμε ακριβώς πώς λειτουργούν σήμερα. Αυτό έχουμε υπόψη μας να κάνουμε. Uh, Ωραία. Ωραία, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Διευθυντά. Θεωρήσατε, περιγράψατε το ρίτσο ως επαναστατικό. Ε, αυτό σίγουρα είναι κάπως περίεργο. Σκοπό είχε να προωθήσει την καινοτομία και τη μακροπρόθεσμη προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος από την ε, δράση κάποιων χημικών. Καταλαβαίνω ότι βρισκόμαστε ακόμα σε πρώιμο στάδιο, αλλά εσείς ως διευθυντής έχετε στοιχεία ότι η νομοθεσία αυτή προωθεί την καινοτομία ότι οδηγεί στην απόσυρση από ε, την αγορά ε, κάποιων χημικών που προκαλούν ανησυχία και την αντικατάστασή τους με λιγότερο βλαβερές ουσίες. Ευχαριστώ. Πέτερτε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Διευθυντά, σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσίασή σας και συγχαρητήρια για την καλή έναρξη των δραστηριοτήτων σας. Ακούγοντάς σας, θυμήθηκα ένα φίλο μου, χημικό μηχανικό, που εργαζόταν σε μια ε, εταιρεία, σε ένα εργοστάσιο ε, τεχνητών αρωμάτων και έλεγε ότι κάθε ουσία που έπαιρνε ε, σε ένα ράφι Είχε την ακροκεφαλή επάνω που έλεγε δηλητήριο και προσοχή. Τελικά, το τελικό προϊόν όμως, το άρωμα, δεν είχε αυτό το, ε, την ένδειξη, αυτό το σήμα. Δεν ήταν επικίνδυνο, γιατί τα λέω αυτά, ότι είναι σοβαρά πράγματα. Εσείς μιλήσατε με τρόπο και με πνεύμα πολύ ανοιχτό και πρόθυμο, αλλά θέλω να σας ρωτήσω, οι πολίτες ενδιαφέρονται ε, να μάθουν ποια είναι η δουλειά σας, τι κάνετε και σε ποιο βαθμό συμμετέχουν και ρωτούν και οι, οι φορείς, οι οργανώσεις κοινωνίας των πολιτών. Ποια είναι η σχέση σας. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Πρέπει να σας πω και ομολογώ δημόσια, ομολογώ, ε, δεν το θεωρώ κακό, ότι το καταψήφισα το Ρίτς. Και διαφώνησα και με την πολιτική μου ομάδα. Διότι έβλεπα αυτό το κείμενο ότι δεν ήταν βιώσιμο, ατελές, με θέματα πάρα πολύ συγκεκριμένα και ασαφή. Για παράδειγμα αυτά τη συμπνευματική ιδιοκτησία. Ένα έγγραφο με τόσο μεγάλη ευθύνη και τέτοιο αντίκτυπο στην κοινωνία δεν μπορεί να αφήνει τα πράγματα έτσι στη θολούρα τους. Γιατί ήταν σαφέστατη η έκθεση από διάφορα ερευνητικά κέντρα που έλεγε ότι δεν υπήρχαν στην Ευρώπη αρκετοί τοξικολόγοι για να ελέγξουν όλα αυτά. Δεν είχε στήριξη από πίσω αυτή η έκθεση ανθρωπίνων πόρων για να ασχοληθούν με το πρόβλημα. Και εγώ το θεώρησα πολύ μεγάλη πολιτική ανευθυνότητα αυτό ως πράξη. Επιπλέον κάτι άλλο με ανησυχεί πάρα πολύ. Η υπεραισιοδοξία σας όταν ήρθατε εδώ και σας κάναμε ακρόαση και προφορική εξέταση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που πρότεινε το ΡΙΤΣ, ξέρουμε έχει και ονόματα και ονοματεπώνυμο και ξέρουμε ποιος το προώθησε αυτό το θέμα, το ενθουσιασμό. Αλλά με εκπλήσει. Βλέπετε το άρθρο που δημοσιεύθηκε στο ε, περιοδικό Nature που λέει ότι δεν υπάρχουν υπολογισμοί δεν, μετρήσαμε καλά πόσους τοξικολόγους έχουμε στην Ευρώπη ή τι γίνεται με τα πυραμιτόζωα. Και λέει 54 εκατομμύρια θηλαστικά χρειαζόμαστε. 54 εκατομμύρια θηλαστικά για να ελέγξουμε όλες αυτές τις ουσίες. Και δεν γίνεται ε, παράλληλη έρευνα καινοτόμα για να μην ε, έχουμε έρευνα σε πειραματόζωα. Και ρωτώ, ποιος θα είναι υπεύθυνο αν πάνε στραβά αυτά όλα. Ποιο θα αναλάβει τι ευθύνε απέναντι σε εταιρείε που δεν προλαβαίνουν, Ποιο αναλαμβάνει την ευθύνη στι εταιρείε που σηκώνονται και φεύγουν. Είναι τεράστιο θέμα, πολιτικό. Είμαστε σε ένα πολιτικό σύστημα όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν λογοδοτεί για τις πράξεις τη. Αυτό με ανησυχεί εμένα βαθύτατα. Θα πρέπει να πούμε στου κυρίους αυτού να πάτε στο δικαστήριο, στο ΔΕΚ και θα έχουμε μια νέα απάντηση για το πώς ε, θα ε, έχουν, ε, θα δικαιώνονται οι πολίτες απέναντι σε μια κακοφτιαγμένη νομοθεσία. Τι γίνεται λοιπόν, σας ερωτώ. Πολλές εταιρείε δυσκολεύονται, δεν μπορούν να φτάσουν, θα μπορούν να προσφύγουν και εις βάρος ποιου και πού. Δεύτερον, έχετε υπολογίσει, γνωρίζετε εταιρείε που έχουν σηκωθεί και έχουν φύγει από την Ευρώπη. Ευχαριστώ. Α, συγγνώμη, έχω κι άλλο. Τελευταίο το Nature ζητάει ένα δικαιοστάσιο, ένα μορατόριο. Εσείς τι λέτε γι' αυτό. Η κυρία Κλάς, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Η Κριστίνα Κουτιέρες αναφέρθηκε στα πολλά προβλήματα που ήδη είχαμε ε, εντοπίσει τότε. Οι άνθρωποι σε μας όταν υπάρχουν προβλήματα με την καταχώρηση κάποιων ε, εταιριών, τη γραφειοκρατία και ε, τις δαπάνες. Είναι προβλήματα που συζητήσαμε τότε. Δεν θα σταματήσουμε να ασχολούμαστε με το θέμα και να θέτουμε ερωτήσεις. Είπατε ότι υπολογίζεται σε μεγάλο φόρτο εργασίας. Δεν είπατε ευθέω ότι ζητάτε περισσότερα χρήματα, αν και ο πρόεδρος αναφέρθηκε στο ότι ε, πήκε εκείνη τη στιγμή στην αίθουσα η συγγήτρια για το θέμα αυτό. Θα θέλαμε να ξέρουμε τι σκοπεύετε να κάνετε με αυτό. Θα αυξήσετε τα τέλη ή θα ζητήσετε περισσότερα χρήματα από τον προϋπολογισμό. Άλλη ερώτηση είναι η συνεργασία με τα κράτη-μέλη. Συμμετέχουν τα κράτη-μέλη σε πολλές επιτροπές. Βρίσκεται ότι αυτό είναι αποτελεσματικό, είναι χρήσιμο ή είναι απλά πολύπλοκο και μπερδεύει τα πράγματα. Είπατε επίσης ότι έχει προσθεθεί μια νέα αρμοδιότητα στις εργασίες της υπηρεσίας σας ε, όσον αφορά τον κανονισμό για τα βιοκτώνα. Η υπηρεσία σας συμμετείχε στην πρόταση της Κομισιόν για τον κανονισμό για τα βιοκτώνα. Είσαστε νέα υπηρεσία, ωστόσο Μπορούμε να επωφεληθούμε από τις εμπειρίες σας ε, της χρονιάς αυτής στον κανονισμό για τα βιοκτώνα. Ευχαριστώ. Παρακαλώ, αν θέλετε να απαντήσετε κύριε Ντάνσερτ σε αυτό το νέο γύρο των ερωτήσεων. Thank you. Promote innovation. Σας ευχαριστώ. Προώθηση της καινοτομίας ε, και οι ουσίες που προκαλούν σημαντικές ανησυχίες. Ήδη έχουμε ενδείξεις ότι οι επιχειρήσεις αντιδρούν στον κατάλογο των υποψήφιων ουσιών. Με τα safety data sheets, με τα φυλάδια που περιέχουν τα, τις ουσίες αυτές οι επιχειρήσεις εξετάζουν αν οι ουσίες αυτές χρησιμοποιούνται στα μείγματά τους και ήδη σκέφτονται πώς θα αντικαταστήσουν τις επικίνδυνες ουσίες. Πιστεύω λοιπόν ότι υπάρχει θετική εξέλιξη στον τομέα αυτών. Βλέπουμε δηλαδή το αποτέλεσμα των νομοθετικών αυτών μέσων. Επίσης βλέπουμε τα αποτελέσματα της καταχώρησης νέων ουσιών. Ακόμα και σε αυτές τις δύσκολες οικονομικά χρονιές, οι επιχειρήσεις συνεχίζουν την καταχώρηση νέων ουσιών που θα διατεθούν στην αγορά. Με τον τρόπο αυτόν λοιπόν, το REACH προωθεί την καινοτομία. Η κοινωνία των πολιτών πώς συμμετέχει. Η κοινωνία των πολιτών συμμετέχει με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Έχουμε πολλές περιπτώσεις όπου γίνονται δημόσιες διαβουλεύσεις. Ήδη αναφέρθηκα στα πειράματα σε ζώα. Αλλά και όταν μπαίνει μια ουσία σε κατάλογο των υποψήφιων ουσιών Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις δηλαδή όπου μπορούν οι επιχειρήσεις να συμμετέχουν στη διαδικασία και να εκφράζουν τις απόψεις τους. Επίσης έχουμε μια πολιτική για τα ενδιαφερόμενα μέρη, για τους stakeholders. ώστε να μπορούμε να λάβουμε υπόψη μας και τις θέσεις των οργανώσεων που εκπροσωπούν το ευρύ κοινό. Επίσης θα δημοσιεύσουμε τις πληροφορίες που θα συλλέξουμε για τις καταχωρήσεις. Θα ξεκινήσουμε μέσα στη χρονιά, πολύ περισσότερες πληροφορίες όμως θα έχουμε τις επόμενες χρονιές, θα δημοσιεύσουμε τις επόμενες χρονιές όπου θα συλλεχθούν και πολύ περισσότερες πληροφορίες. Οι καταναλωτές και άλλες οργανώσεις θα μπορούν να επωφελούνται από τις πληροφορίες αυτές. Άλλη ερώτηση είναι εάν θα αρκούν τα τέλη. Θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε λόγο να πιστεύουμε ότι δεν θα αρκούν τα τέλη. Τα τέλη είναι πολύ χαμηλότερα από αυτό που είχαμε υπολογίσει στην αρχή, διότι τελικά θα γίνουν πολύ λιγότερες καταχωρήσεις αυτή τη στιγμή από αυτούς που έκαναν προκατακτική καταχώρηση. Περιμένουμε όμως πολύ μεγαλύτερο όγκο τελών στο τέλος της επόμενης χρονιάς όταν θα πλησιάζει η προθεσμία. Το εάν οι επιχειρήσεις θα μπορούν να τηρήσουν την προθεσμία αυτή όσον αφορά το θέμα αυτό, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό για τι επιχειρήσει να έχουν μία σαφή προθεσμία στο μέλλον, η οποία να μην μετακινείται με το παραμικρό πρόβλημα. Ουσιαστικά είναι πολύ σημαντικό οι επιχειρήσει να μπορούν να προετοιμαστούν εγκαίρως, ώστε να μπορούν να συμμορφώνονται με την νομοθεσία. Νομίζω ότι έχουμε δώσει ορμή στην όλη διαδικασία στην Ευρώπη. Έχουμε πείσει τον κόσμο να συμμετέχει και να υποβάλει τους σχετικούς φακέλους. Πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό να μην χάσουμε την ορμή αυτή με το να ξανασκεφτούμε τις προθεσμίες, να αλλάξουμε τις προθεσμίες. Αφήνω βέβαια σε εσά να αποφασίσετε αν χρειάζεται ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Εμείς πιστεύουμε ότι χρειάζεται και εργαζόμαστε σκληρά πάνω σε αυτό. Όσον αφορά τα βιοκτώνα. Η υπηρεσία μας έχει δεχθεί να εργαστεί στον τομέα των βιοκτώνων στο μέλλον. Αυτή τη στιγμή Έχουμε επιδοτήσεις μόνο για εργασίες που αφορούν το REACH. Δεν έχουμε πόρους να εργαστούμε πάνω σε τίποτα άλλο πέρα από το REACH. Στο μεταξύ όμως έχουμε συμβάλει και στη δουλειά αυτή για να μπορέσουμε όμως να εργαστούμε πιο ουσιαστικά πάνω στην προετοιμασία των, των βιοκτώνων θα πρέπει να ξεκινήσουμε εγκαίρως την διαδικασία ένταξης των βιοκτώνων στα χημικά πάνω στα οποία εργαζόμαστε. Μου διέφυγε κάτι. Συνεργασία με τα κράτη-μέλη. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Οι εμπειρίες μας ήταν εξαιρετικές. Ουσιαστικά θα πρέπει να συνεργαστούμε με τα κράτη-μέλη όσον αφορά την υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Τα κράτη-μέλη όμως έχουν δουλειά να κάνουν και στον τομέα του ρίτσι. Οι αρμόδιες αρχές τους δηλαδή πρέπει να κάνουν πολλή δουλειά και η αξιολόγηση των ουσιών είναι η πιο πολύπλοκη δουλειά που έχουν να κάνουν. Θα πρέπει να εργαστούν και εμείς τους βοηθάμε όσο μπορούμε περισσότερο. Είναι σημαντικό να διατηρήσουν τους σπόρους που είχαν κατά την προηγούμενη θητεία, ώστε να μπορούν να κάνουν τη δουλειά αυτή που αφορά το REACH. Συνεργαζόμαστε με τις αρχές επιβολής του νόμου, ώστε να φροντίσουμε να είναι καλά προετοιμασμένες οι αρχές. Κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει μόνο σε στενή συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές στα κράτη-μέλη. Είναι απαραίτητη λοιπόν η συνεργασία. Θα έλεγα ότι μέχρι στιγμής οι εμπειρίες μας ήταν θετικές. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Γενική Διευθυντά. Και τώρα, ορίστε. Άφησα ερώτηση. Πρόεδρε, μπορεί να σας ενδιαφέρει ο πρόεδρος της Τσεχικής Δημοκρατίας μόλις υπέγραψε τη συνθήκη της Λισαβόνας. Ευχαριστώ, Κρίς, για αυτή την ωραία είδηση. Το περιμέναμε, αλλά δεν πάει περιπτώσει. Καλό νέο είναι. Η κυρία Φρανσουάς Γκροστέτ, παρακαλώ. Merci. Alors, je, je crois, euh, Monsieur Directeur, que je vais, je vais reprendre. Κύριε Διευθυντά, νομίζω πως θα επαναλάβω κάποια πράγματα που ήδη υπόθηκαν, αλλά νομίζω πως είναι σημαντικό να επιμείνουμε στις δυσκολίες που αντιμετωπίζονται, γιατί αυτό που θέλαμε όταν δουλέψαμε στο ΡΙΤΣ να μην φτιάξουμε μία ορολογιακή βόμβα. Ακριβώς αυτό πρέπει να αποφύγουμε λοιπόν. Όμως όταν συζητάμε με τις μεγάλες εταιρείες, ε, τις χημικές, με τις μεγάλες επιχειρήσεις, εταιρείες, βιομηχανίες, ε, τις χημικές, μας εξηγούν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν. Δεν αμφισβητούν τους στόχους προς επίτευξη, το ρίτσο δηλαδή καθόλου, όχι. Αλλά ε, οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν και την ανάγκη που έχουν και μπόρεσα να συζητήσω με τέτοιους ανθρώπους να προσλάβουν άτομα ψηλά ως που να ασχολούνται μόνο με αυτό το θέμα καταχώρησης ρίτσο και όταν βρισκόμαστε σε μια περίοδο οικονομικής κρίσης, ε, το ερώτημα που τίθεται λοιπόν είναι η χρηματοδότηση που, πρέπει να, που είναι υποχρεωμένες να αφιερώσουν αυτές οι εταιρείε στην εφαρμογή του REACH, η χρηματοδότηση, αυτά τα χρήματα, εν πάση περιπτώσει, θα χάνουν μεγαλύτερη χρησιμότητα αλλού. Το ίδιο και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, διότι Είχα την ευκαιρία να συζητήσω με μεγάλες εταιρείε που μου λένε, χημικές βιομηχανίες που μου λένε ότι ναι, να το κάνουν, να κάνουν τα πάντα για να βοηθήσουν τις μικρές, αλλά ούτως ή άλλως δεν θα τα καταφέρουν όλες να τηρήσουν το REACH μέσα στις προθεσμίες. Μα λέτε λοιπόν, βεβαίω με καλή θέληση και καλή την πίστη, δεν σα αμφισβητώ καθόλου, αλλά όταν μου λέτε πώ έχουμε φτιάξει, έχουμε προετοιμάσει βοήθεια, γραφεία βοήθεια, ε, άμεση βοήθεια από το, δική σας, ε, το δικό σα οργανισμό και όλα αυτά, το κάθε κράτο μέλο έχει τη δική του, το δικό του γραφείο βοήθεια. Αλλά όταν κανείς καλεί το Εθνικό Γραφείο Βοήθειας, στην πράξη πέφτει πάνω σε operators που δεν απαντούν παρά μόνο με νομικές παραπομπές. Λένε ας πούμε ότι για το τάδε πρέπει να αναφερθεί να πάτε στο άρθρο χ, σημείο ψ, εδάφιο ω. Δηλαδή πρακτικά δεν βοηθάνε. Οι μικρομεσαίες δεν ωφελούνται από τη βοήθεια αυτή. Φοβούμε λοιπόν πως όλα αυτά τα εργαλεία είναι πολύ τεχνοκρατικής φύσης, αλλά όχι αρκετά συγκεκριμένα για να απαντήσουν πραγματικά στα αιτήματα των επιχειρήσεων. Αυτό λοιπόν είναι πρόβλημα και είναι πολύ περίπλοκο. Πολύ περίπλοκο και φτάνει μέσα σε ένα πλαίσιο, όπως σας είπα, οικονομικής κρίσης, όπου η βασική ανησυχία των μικρομεσαίων μας είναι να βρουν αγορές, να επιβιώσουν ορισμένες από αυτές, ενώ εμείς στην ουσία τους φορτώνουμε υπερβολικά στη λειτουργία τους με την εφαρμογή του REACH. Κατανοώ πολύ καλά ότι πρέπει να τηρήσουμε τις προθεσμίες. Εντάξει, είναι μια αρχή, είναι προφανές. Αλλά νομίζω πως θα πρέπει να, έχουμε, να είμαστε αρκετά ευέλικτοι ώστε να λάβουμε υπόψη το σημερινό πλαίσιο και να μην τους πνίξουμε, γιατί την ημέρα που δεν θα έχουμε πλέον επιχειρήσει δεν θα χρειάζεται και να γίνεται και καμιά καταχώρηση. Ευχαριστώ. Η κυρία Γιούτα Χάουκ. Ευχαριστώ πολύ. Δεν ήθελα να μιλήσω καθόλου στη συζήτηση αυτή, αλλά ακούγοντας τους συναδέλφους και τις συναδέλφους, καμιά φορά ερωτώ με πού βρισκόντουσαν όταν είχαμε αποφασίσει το ΡΙΤΣ. Την περασμένη θητεία ήτανε. Ε, και τώρα υπάρχει αυτή η νομοθεσία και ισχύει. Και παρακαλώ και να θυμίσω σε όλους τους συναδέλφους ότι οι μεγάλες πολιτικές ομάδες ε, στην περασμένη θητεία, μάλλον το μεγαλύτερη ομάδα ήταν η ίδια με σήμερα, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Και ήταν πολύ αποφασιστική η στάση της στο τι θα γίνει με το ΡΙΤΣ. Δηλαδή δούλεψαν και αυτοί με αυτό, το πρώτο που θέλω να πω. Το δεύτερο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι συνομοθέτης. Και όταν λέω συν, υπάρχει και άλλος συν νομοθέτης που είναι το Συμβούλιο. Και το Συμβούλιο ακριβώς αυτή τη νομοθεσία ρίτς τη συναποφάσισε. Και στο Συμβούλιο η πλειοψηφία όλων των κυβερνήσεων ήταν δεξιές κυβερνήσεις. Έτσι. Αυτά. Και έτσι έχει τώρα η κατάσταση. Πώς φτάσαμε εδώ. Έχουμε τον κύριο Ντάνσερτ που είναι Γενικός Διευθυντής και έχει ε, το καθήκον να τα διαχειρίζεται. Δεν μπορούμε να του επιρρύπτουμε ευθύνε για την νομοθεσία. Τι θέλαμε εμεί και τι θα θέλαμε εδώ και τι θα θέλαμε εκεί. Μα δεν φταίει ο άνθρωπος γι' αυτό. Δεν έχει νόημα να συζητάμε αυτά. Εγώ θα επιθυμούσα όλοι οι συνάδελφοι να κοιτάξουν λίγο τι έχει κάνει το Συμβούλιο και τι κάνει με τον οργανισμό αυτό. Έχει πετσοκόψει τον προπολογισμό, έχει περικόψει. Το είπε ο Σλούτερο ότι καταφέραμε τώρα να αυξήσουμε σε πρώτη ανάγνωση τα κονδύλια. Να επαναφέρουμε το αρχικό ποσό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συν τα λεγόμενα assigned revenues, ε, τα προβλεπόμενα έσοδα. Συμφώνησαν λοιπόν όλοι οι συνάδελφοι, όλα αυτά ωραία και καλά, αλλά γνωρίζουμε ότι και το επόμενο ε, έτος του προπολογισμού πάλι θα είναι το ταμείο μείον. Παρακαλώ λοιπόν όλους τους συναδέλφους. Κρίμα τώρα που βγήκε ο Φλόρεντς. Γιατί αυτός με εκνεύρισε περισσότερο από όλους τους άλλους. Γιατί είπε ότι έχει τη δυνατότητα να ε, συμμετέχει και να κάνει διαβήματα σε διαφόρους εκπροσώπους του Συμβουλίου για να φροντίσει να είναι σωστή η πρικοδότηση του οργανισμού για να μπορέσει να κάνει σωστά τη δουλειά τους και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όχι μόνο ο οργανισμός ε, ε, να φορτώνεται με επιπλέον αρμοδιότητες. Καταλαβαίνω και αυτό που λέει η κυρία Κλάς. Τι γίνεται με τα βιοκτώνα και θα επιθυμούσαμε αυτό και εκείνο και το άλλο και να κάνει δουλειά και γι' αυτό ο οργανισμός. Μα εμείς φτιάξαμε ένα οργανισμό με συγκεκριμένη δομή και βάση για τη δράση του. Έτσι. Και πάλι νομοθέτημα είναι, νέο νομοθέτημα, να τη δώσουμε και άλλη αρμοδιότητα. Δεν είναι μεταξύ τύρου και αχλαδιού, ας πούμε, βάλε και κάτι ακόμα, βάλε και τα βιοκτώνα. Καλό λοιπόν όλους τους συναδέλφους. Ο, όποιος θεωρεί ότι χωλαίνει το σύστημα κάπου να κάνει ό,τι μπορεί, αλλά να κάνει ό,τι μπορεί προς το Συμβούλιο να κάνει κρούση. Και τα κράτη-μέλη δηλαδή. Ο καθένας από εμά έχει και ιδιαίτερη ευθύνη και καθήκον και εμείς και ε, οι εταιρείες μας να πετύχουν στην προσπάθεια αυτή με το REACH. Ξέρω ότι δεν πρέπει να φροντίζομαι τόσο συναισθηματικά, να είμαι πιο ψυχρή και να λέω εντάξει, το βάλαμε σαν αυλάκι, ε, καταλήξαμε και για τον προπολογισμό, αλλά καμιά φορά δεν καταλαβαίνω τους συναδέλφους. Εγώ έτσι κι αλλιώς αναπληρωματικό μέλος ήμουν εδώ ανέκαθεν Προέρχομαι από μια περιφέρεια που έχει χημική βιομηχανία. Εχθές ε, μίλησα με πολλά διοικητικά συμβούλια και συμβούλια εργαζομένων και δεν άκουσα την παρά μικρή επίκριση. Έτσι, ίσως και αυτό πρέπει να το πούμε καμιά φορά. Δεν έχουμε άλλες ερωτήσεις. Κύριε Διευθυντά, πριν σας δώσουμε το λόγο, θα ήθελα με την άδειά σας να προσθέσω κι εγώ μια ερώτηση. Σε σχέση με τα όσα είπε η κυρία Χάουκ, συμφωνώ αρκετά με την άποψή της. Μπορεί κανείς να καταλάβει τις δυσκολίες των εταιριών, όντως, αλλά θα πρέπει επίσης να θυμίσουμε την αναγκαιότητα του κειμένου και τη σημασία που έχει για τους πολίτες μας, για τη δημόσια υγεία. Τι οικονομίες θα έχουμε από πλευράς δημόσιας υγείας και τι πρόοδο ε, από προϊόντα υποκατάστασης. Λοιπόν, ερωτώ περισσότερο τι χρειάζεστε τώρα για να ανταποκριθείτε στις υποχρεώσεις σας από το κείμενο που, που εμείς ψηφίσαμε και για να ε, σαρκώσετε την αποστολή σας. Κανείς δεν την αμφισβητεί τώρα, να δούμε πώς θα ανταποκριθείτε σε αυτό το έργο. Thank you for this, uh, σας ευχαριστώ για τα λόγια σας. Νομίζω πως εδώ έχουμε μια διαφορά απόψεων για το πώς θα πρέπει να βοηθηθούν οι επιχειρήσεις. Βασικά όμως, θέλω να πω ότι έχουμε και κάποιον εκπρόσωπο του βιομηχανία που μας ακούει. Εμείς είμαστε ένας οργανισμός που δουλεύει χέρι-χέρι με την βιομηχανία καθημερινά. Συζητούμε κάθε δύο εβδομάδες για την πρόοδο που σημειώνεται. Κανένας άλλος οργανισμός δεν το κάνει αυτό τόσο πολύ προσπαθώντας να βοηθήσει τη βιομηχανία να καταλάβει ακριβώς ποιες είναι οι ανάγκες τους και να τους βοηθήσουμε. Πολλούς πόρους αφιερώνουμε σε αυτό το σκοπό. Και επίσης ε, συνεργάζονται στην ανάπτυξη κάθε εγχειριδίου μας, κάθε εργαλείο πληροφορικής, μας στέλνουν τα δικά τους εργαλεία για το δική τους, ε, ε, δικό τους κλάδο, σχολιάζουμε τα δικά τους εγχειρίδια, οπότε νομίζω πως ε, πραγματικά δεν φιδόμεθα ουδεμίας προσπάθειας ώστε να μπορέσουμε να τους βοηθήσουμε όσο γίνεται περισσότερο τις εταιρείε και τις ενώσεις τους. και αυτό αφορά και τις επαφές με τις ενώσεις των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Τους καλούμε στις συνεδριάσεις μας κάθε φορά και τους ε, ε, λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη μας, όσο γίνεται περισσότερο. Εγώ πραγματικά δυσκολεύομαι να δω πού μπορούμε να κάνουμε περισσότερα πράγματα, αλλά καταλαβαίνω φυσικά πως η οικονομική περίσταση είναι πολύ δύσκολη. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Και αυτό έχει προκαλέσει ε, χάσιμο χρόνο, καθυστερήσεις. Και γι' αυτό και σας εξήγησα ότι προσπαθούμε να ανακτήσουμε αυτό το χαμένο καιρό δίνοντάς τους ε, νέα εργαλεία, νέα στοιχεία ώστε να τους βοηθήσουμε να καταρτήσουν το ε, ντοσιέ, τους φακέλους τους. Είμαστε σε επαφή με τις ενώσεις ακόμη περισσότερο και όπως σας είπα εμείς ε, καλούμε όλες αυτές τις ενώσεις ώστε να είμαστε βέβαιοι πως οι μικρομεσαίες έχουν πρόσβαση στα στοιχεία που συγκεντρώνουν τα, οι συμπράξεις Τώρα όσον αφορά τα εθνικά γραφεία βοήθειας προσπάθησα να εξηγήσω τι κάνουμε. Θα προσπαθήσουμε και να τους εκπαιδεύουμε περισσότερο. Θα έρθουν πάλι την επόμενο μήνα στον οργανισμό μας για να μάθουν πώς μπορούν να βοηθηθούν περισσότερο. Έχουμε αναπτύξει και ένα εργαλείο μέσω του οποίου να δίδουμε πολύ πιο συγκεκριμένες απαντήσεις στις ερωτήσεις και επίση, θα πρέπει να μας ε, να, έρχονται σε επαφή μαζί μας και αν είναι οι νομικής φύσης οι ερωτήσεις ε, για την εφαρμογή του REACH ε, να είμαστε σε συζήτηση με την Κομισιόν και η Κομισιόν μας βοηθά στην επίλυση αυτών των θεμάτων για τον επόμενο, το επόμενο διάστημα. Νομίζω ότι με αυτά κάλυψα τις ερωτήσεις που μου υποβλήθηκαν. Εκτός από αυτά που νωρίτερα με ρωτήσατε για την πνευματική ιδιοκτησία. και σε αυτό το πλαίσιο προστατεύουμε την πνευματική ιδιοκτησία, όπως προβλέπεται και από την νομοθεσία, γιατί πρέπει να διασφαλίσουμε το σεβασμό της ασφάλειας καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε τα συστήματά μας να είναι πάντοτε ασφαλή από τις ε, δυσδύσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Δευθυντά, κύριε Ντάντσετ για την εκτενή σας απάντηση στις πολλές μας ερωτήσεις. Βλέπετε ότι ενδιαφέρεται σφόδρα η Επιτροπή μας να παρακολουθεί και να συνοδεύει τις εργασίες σας έχουμε τον Guido Σακώνη και τον Χάρτμοντ Νάσα, δύο νέους συνδέσμους ε, που είμαι βέβαιος ότι θα εξασφαλίζουν αυτό το σύνδεσμο με τον οργανισμό σας. Και επίσης σημειώσαμε ότι μας έχετε προσκαλέσει να δούμε επιτόπου τη δουλειά σας. Οπωσδήποτε το επόμενο διάστημα θα διστάσουμε να αξιοποιήσουμε αυτή τη δυνατότητα. Λοιπόν, ό,τι επιθυμείτε, καλό κουράγιο, καλή δύναμη γιατί είναι πραγματικά ακρογωνιαίος λίθος ο οργανισμός σας στην περιβαλλοντική μας πολιτική, στο Επανειδήν, εδώ στην Επιτροπή μας ή σε εσάς στο Ελσίνκι. Ευχαριστώ. Γεια σας. Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, πάμε στο σημείο 5 αισίως τη μέση της διάταξης και έχουμε προσκαλέσει άλλον έναν οργανισμό Πολύ σημαντικό επίσης και αυτός. Έχουμε λοιπόν τώρα ε, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος της Κοπενχάγης.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 It's just been announced, so uh, it's in a it's in a document. So at the Arctic Council, it will be put on the table. But there's no. Okay. Yeah, ich darf ganz herzlich... Καλώς. Λοιπόν, καλωσορίζω θερμότατα ενώπιόν μας την εκτελεστική διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, κυρία Τζάκλιν Μακλέιντ, και τους συνεργάτες της, Καλώς ορίσατε θερμότατα στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Καλώς όριζω και τον κύριο Λούντο Φαν Χόλτσμπεκ, που είναι αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Και επίσης ε, πρέπει να σας πω ότι έχει εριστεί από το Κοινοβούλιο. Κυρία Μακλέιτ, είστε ε, από τους παλαιότερους οργανισμούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχετε το καθήκον να μας ε, δίνει τις προφορίες που χρειαζόμαστε για να έχουμε καθαρή ατμόσφαιρα, καθαρά νερά, προστασία του κλίματος, ένα σύστημα δορυφορικό για να έχουμε και περισσότερα στοιχεία στη διάθεσή μας. Έχουμε ε, τη μεγάλη διάσκεψη της Κοπενχάγης σε λίγες εβδομάδες και σημειώνουμε με ευγνωμοσύνη ότι θέλετε να μας βοηθήσετε στην προσπάθεια αυτή, αν χρειαστεί, στην επιμελητεία, ε, στην Κοπενχάγη, στην υποδομή. Είναι τεράστια αυτή η διάσκεψη και δεν πρέπει κανείς να την αντέξει κιόλα. Λοιπόν, ενδιαφερόμαστε βεβαίω πολύ να ακούσουμε τι έχετε να μας πείτε πώς ε, είναι οι εργασίες στον οργανισμό σας, πώς έχει εξελιχθεί η εργασίες σας εκεί και πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε γενικότερα άλλο θέλετε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Είναι μεγάλη μου χαρά να βρίσκομαι εδώ σήμερα. Ε, έχω πολλούς φίλους μεταξύ των μελών της ε, ε, Επιτροπής. χαίρομαι που σας ξαναβλέπω και προσθέτω στην καλή συνεργασία μαζί σας, ιδιαίτερα, στους, ιδιαίτερα με τους επανεκλεγόμενους. ελπίζω επίσης να δημιουργήσω νέες φιλίες με ανθρώπους που δεν είχα την ευκαιρία να συναντήσω μέχρι τώρα. Επιτρέψτε μου για αυτούς που ήδη γνωρίζετε την, ε, τον οργανισμό μας ε, να πω λίγα λόγια. Η εντολή του οργανισμού είναι έτσι διατυπωμένη που ουσιαστικά προδικάζει πολύ από τη δουλειά μας. Ε, πράγματι ασχολούμαστε με την ε, αηφόρο ανάπτυξη. Σκοπός μας είναι να πετύχουμε ε, σημαντική και μετρήσιμη βελτίωση του περιβάλλοντος της Ευρώπης και να παρέχουμε έγκαιρες και αξιόπιστες πληροφορίες και θέλω να τονίσω το αξιόπιστες για να για, για να έχει ο κόσμος περισσότερη συνείδηση της σημασίας του περιβάλλοντος για την οικονομία της Ευρώπης. Ε, το, ε, μας ενδιαφέρει πάρα πολύ η στενή συνεργασία μαζί σας, ε, συνεργαζόμαστε συνεχώς στενά μαζί σας και έχω μαζί μου μέρος ε, του προσωπικού μου. Σήμερα συνήθως καθόμαστε εκεί γύρω και ε, θα έχετε την ε, ευκαιρία να συνομιλήσετε και με αυτούς και με μένα. Θα έχουμε και συζητήσεις με τις διάφορες ομάδες και τους εισηγητές. Θα ήθελα να θίξω ιδιαίτερα δύο θέματα. Το ένα έχει να κάνει με την αλλαγή του κλίματος ε, και την επικείμενη ε, ε, συνάρτηση στην Κοπεχάκη και το άλλο είναι η έκθεσή μας για την κατάσταση του περιβάλλοντος που ε, θα ήθελα να τονίσω ιδιαίτερα στα πλαίσια του έκτου ε, προγράμματο ε, πλαισίου. Αυτά λοιπόν είναι τα δύο θέματα που θα να συζητήσω μαζί σα σήμερα. 42 μέρε απομένουν, δεν είναι πολύ χρόνο. Θα γίνει συνάντηση στη Βαρκελόνη. Γίνεται συνάντηση στη Βαρκελόνη και νομίζω ότι το ψήφισμά σα το οποίο θέλω να αναγνωρίσω διότι στοχεύει ψηλά όσον αφορά την ε, τοποθέτηση της Ευρώπης στα θέματα αυτά. Ε, ωστόσο, ε, πιστεύουμε ότι θα υπάρχει πολλή δουλειά που θα πρέπει να γίνει. Τι κάνουμε εμείς λοιπόν μέσα σε όλες αυτές τις συναντήσεις, τις συμβάσεις, τα δεδομένα κλπ. Δουλειά μας είναι να παρέχουμε αξιόπιστες πληροφορίες όσον αφορά το αποτέλεσμα των ε, πολιτικών ε, για την αντιμετώπιση της ε, αλλαγής του κλίματος. Για να μπορεί η ευρωπαϊκή κοινότητα να συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις της σχετικά με την υποβολή εκθέσεων στα πλαίσια του Διεθνούς Καθεστώτος για την Προστασία του Περιβάλλοντος, υποβάλλουμε ετησίως δύο εκθέσεις ε, που υποβάλλεται στο, μέσω της Επιτροπής ε, στο, ε, της Κομισιόν στην σύμβαση του ΟΗΕ για την προστασία του περιβάλλοντος. Πολλοί κόσμος έχει πει ότι οι εξελίξεις που βλέπουμε, ότι η μείωση των εκπομπών του, το αερίου που βλέπουμε είναι μια ανώμαλη κατάσταση λόγω της οικονομικής κρίσης κτλ. Αλλά δεν είναι. Είδαμε κάποιες εκτιμήσεις ε, του Αυγούστου του 2009, πολύ πρόσφατα δεδομένα δηλαδή, λένε ότι οι εκπομπέ μα ε, για τα 27 κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση ε, είναι 10,7% κάτω από το, το επίπεδο του 1990. Ε, ήδη, έχουμε, έχουμε πετύχει 6,2 μείωση. Ε, ξέρω ότι είναι πολλά νούμερα αυτά, αλλά αυτή ουσιαστικά είναι η ουσία της ε, συζήτησης αυτής. Οι εκπομπές μας δηλαδή είναι 10,5% του διεθνούς ε, συνόλου που καλύπτεται από τη Σύμβαση για την Αλλαγή του Κλίματος στο ΙΕ. Ε, αυτό που κάνει η Ευρώπη λοιπόν δεν μπορεί να σταθεί από μόνο του. Σημαντικό όμως είναι να τονίσουμε ότι η Ευρώπη έχει θέσει πολύ, σημαντικούς, πολύ αυστηρούς στόχους και σε πολύ, ε, τους ε, έχει πετύχει και τους έχει ξεπεράσει μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις. Ε, ανά άτομο οι εκπομπές είναι το πιο σημαντικό στοιχείο που έχουμε. Από το 1990 μέχρι το 2007 μειώσαμε τις μέσα σε εκπομπές ανά άτομο από 11,8 σε 10,2 τόνους σε ισοδύναμου ε, διοξιδίου του άνθρακα. Αυτό είναι πάνω από τον ε, παγκόσμιο μέσο όρο που είναι 7 τόνοι, αλλά δείχνει αυτό ότι έχουμε ε, αντιστρέψει την εξέλιξη όσον αφορά τις εκπομπές μας αερίων του θερμοκηπίου και σίγουρα αυτό είναι χαμηλότερο από 15 τόνους που είναι το, ο μέσος όρος για τις ε, βιομηχανικές χώρες. Η ε, Ευρώπη λοιπόν ε, πράγματι έχει πετύχει μείωση των εκπομπών. 79 με 80% για το 2007 ήταν κατανάλωση ενέργειας και οι μεταφορές ιδιαίτερα συνέβαλαν σημαντικά στα στοιχεία αυτά. Έχουμε λοιπόν πολλή δουλειά να κάνουμε με τους συναδέλφους μας στον τομέα των μεταφορών. Έχει αναπτυχθεί και το μερίδιο των αερομεταφορών 6% το 2007. Ε, έχουμε κάνει κάποιες ε, ε, προβλέψεις που δείχνουν προς τα που πηγαίνει η Ευρώπη. Πριν 10 χρόνια, όταν αρχίσαμε πρώτα να λαμβάνουμε στοιχεία, υπήρχε μια κάπως αρνητική προσέγγιση. Η στόχη του Κιώτο ήταν μακρινή. Μέσα στην τελευταία δεκαετία όμως έχουμε φτάσει σε σημείο όπου 10 από τα 15 κράτη-μέλη αναμένεται να πληρώσουν τους στόχους του Κιώτο για το 2000 και τώρα το 2009 θα δείτε την επόμενη εβδομάδα στις 12 Νοεμβρίου που ε, θα ε, ανακοινωθεί η έκθεση θα δείτε ότι όλες οι χώρες μας εκτός από μία ε, θα ε, πληρεί τους στόχους του Κιώτο. Είσαστε οι πρώτοι που θα λάβετε την έκθεση αυτή. Είναι πολύ κρίσιμη η στιγμή αυτή. Μπορεί η Ευρώπη να πει πράγματι ότι έχει πραγματοποιήσει τους στόχους της. Ε, για να ε, σας βοηθήσουμε έχουμε δημιουργήσει και μια διαπαφή ε, μέσω διαδικτύου όπου μπορείτε να δείτε τις πηγές των εκπομπών του θερμοκηπίου και να δείτε τα παρασκήνια. Έχουμε προχωρήσει ένα βήμα πιο πέρα. Πολλοί από εσά θα θεωρείτε ήδη ότι η αλλαγή του κλίματος έχει χτυπήσει την πατρίδα σας. Έχουμε εξετάσει τις συνέπειες και το πόσο ευάλωτη είναι η Ευρώπη. Έχουμε μια μακρά σειρά δικτών. Έξω θα δείτε την τελευταία μας έκθεση την έκθεση για τις Άλπεις. Ε, εδώ πράγματι ε, θα διαβάσετε πολύ σοβαρά πράγματα. Θα δείτε ότι είναι πολύ σοβαρές οι ε, τροποποιήσεις, οι αλλαγές που έχουν γίνει και στη βιοπικιλότητα, στα ύδατα και γενικά στην συγκεκριμένη αυτή η περιφέρεια όσον αφορά δηλαδή την διαχείριση της αλλαγής στους σπόρους. Είδαμε αύξηση της παγκόσμια θερμοκρασία κατά 0,8 βαθμού Κελσίου. Σε περιφερειακό επίπεδο όμω ε, η κατάσταση διαφέρει. Στην Ευρώπη ήδη έχουμε δει μεγαλύτερη αύξηση και στην Αρκτική η αύξηση είναι σχεδόν διπλάσια από ό,τι είναι ο διεθνή μέσο όρο. Εάν λοιπόν μιλάμε για έναν στόχο 2 βαθμών Κελσίου, και η Ευρώπη βρίσκεται κοντά στον έναν βαθμό Κελσίου, μένει άλλος ένας βαθμός. Και ο ένας βαθμός που ήδη έχουμε ζήσει είναι το παράθυρο μέσα στο οποίο έχει ε, αναπτυχθεί όλη η Ευρώπη, η Γεωργία κτλ. Τα τελευταία 10.000 χρόνια είχαμε μια πολύ σταθερή περίοδο και τώρα ε, κινδυνεύουμε να ξεφύγουμε από την κατάσταση, από, ε, από την κατάσταση αυτή. Πολύ ευχαρίστω σα συζητήσω το θέμα αυτό. Βρισκόμαστε ήδη σε πολύ ευάλωτη θέση αν και ε, υπάρχουν διακυμάνσεις σε διάφορες ε, περιοχές. Έχουμε περιοχές ε, όπου υπάρχει κίνδυνος πλημμυρών ή άλλων φυσικών καταστροφών. Και φυσικά στην Αρκτική η προσέγγιση μας θα είναι διαφορετική. Βλέπουμε διαφορά στις βροχοπτώσεις, εάν και θα πρέπει να επιβεβαιώσουμε τα δεδομένα αυτά. Από ό,τι φαίνεται όμως οι μεσογειακές περιοχές έχουν 20% λιγότερη βροχή από ό,τι στη Μεσόγειο. Έχουμε... Ε, αύξηση της στάθμης θάλασσας 3,1 ε, ε, εκατοστά το χρόνο και 3,1 εκατοστά συνολικά και έχουμε δει διάφορα καταστροφικά γεγονότα στην Ακτική βλέπουμε ότι έχει μειωθεί ο όγκος των πάγων κατά 46% και βλέπουμε ότι απειλούνται πολλά οικοσυστήματα, ε, η χλωρίδα και η πανίδα δηλαδή. Δεν ε, μπορούμε να, ε, να εφησυχαστούμε, θα πρέπει να εξετάσουμε όλες τις πολιτικές μας και η δική σας Επιτροπή θα ηγηθεί στις προσαρμογές στην αλλαγή του κλίματος και θα έχει την επισκόψη των εξελίξεων στην πολιτική σε όλη την Ευρώπη. Ακούω όλο και περισσότερο ότι ακούω ότι θα συμμετέχουν όλοι και περισσότεροι στην ε, συνάντηση της Κοπεχάγης. Ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει, ε, έχει φτάσει στο μέσο των στόχων για το 2020. Έχουμε όμως και μία πιθανή μείωση 30% στα πλαίσια της γενικής αυτής παγκόσμιας συμφωνίας και θα ήθελα να αναγνωρίσω αυτό που έχει πει το Κοινοβούλιο σας όσον αφορά του υψηλούς στόχους. Το θέμα όμως είναι η διεθνή συνεργασία. Η αλλαγή του κλίματος ε, έχει να κάνει με την ε, παγκόσμια ρύθμιση, την ε, νομοθεσία. Θα πρέπει λοιπόν οι κυβερνήσει να αναλάβουν ηγετικό ρόλο. Νομίζω ότι αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να βοηθήσουμε στην κατανόηση των λύσεων, να σημειώσουμε βέλτιστες πρακτικές, benchmarking, να δούμε πώς μπορούμε να παράγουμε βιώσιμη ενέργεια, πώς μπορούμε να ορίσουμε τις πράσινες θέσεις απασχόλησης, διότι υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορούν να πάρουν την ετικέτα αυτή, που μπορεί όμως να αποτελούν απλά βραχυπρόθεσμο ε, γέμισμα ε, κενών. Η συνάντηση Κοπεχάγη 15 δεν θα είναι η τελευταία μας λέξη στην αλλαγή του κλίματος. Ε, ο οργανισμός μας όμως θα είναι έτοιμος, ε, άσχετα από το ποιο θα είναι το αποτέλεσμα, ώστε να ε, βοηθήσει στην εφαρμογή, την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων για οποιαδήποτε συμφωνία θα προκύψει. Σίγουρα στο πακέτο κλίματος και ανανεώσιμης ενέργειας θα ισχύει ότι θα πρέπει να ε, φτάσει στα χέρια των πολιτών για να μπορούν να καταλάβουν πώς μπορούν οι πολιτικές να οδηγήσουν σε αλλαγή της κατάστασης. Μας ενδιαφέρει πολύ να ε, ακούσουμε οι ιδέες που θα βοηθήσουν στην ε, επίλυση των προβλημάτων. Θέλουμε να δούμε πού πραγματικά έχουμε σημειώσει πρόοδο. Από την πρακτική πλευρά θα ήθελα να πω ότι κατά τη ε, διάσκεψη για το κλίμα της Κοπεχάγης ε, είσαστε ε, ευπρόσδεκτοι να εργαστείτε στα γραφεία της υπηρεσίας, του οργανισμού μας. Θα... Είσαστε πάρα πολύ βέβαια τώρα πια. Ε, σας προσφέρουμε λοιπόν τη δυνατότητα, σας παρακαλώ να μας ενημερώσετε εγκαίρως, διότι θέλουμε η παραμονή σας στην Κοπεχάγη και στον οργανισμό μας να είναι όσο πιο αποτελεσματική, επικοδομητική ε, και παραγωγική γίνεται. Να κλείσω λέγοντας ότι θα συμμετέχουμε, θα παίξουμε υποστηρικτικό ρόλο θα μιλήσουμε για τους ωκεανούς, ε, τις, τους καταλόγους αερίων του θερμοκηπίου, τις ε, εκπομπές, θα αναπτύσσουμε ένα, ε, ένα σύστημα υπολογισμού των, ε, των εκπομπών του κάθε προσώπου. Μίλησα για την συνάντηση της Κοπεχάγης, θα ήθελα όμως να αναφερθώ και στο πρόγραμμα μας για το 2010, όπου θα βρείτε μεγάλο μέρος της δουλειάς μας ε, που αφορά το έτος βιοπικιλότητας περιέχει όμως ε, και εκθέσεις ε, σχετικά με το περιβάλλον της Ευρώπης. Φέτος είναι κάπως διαφορετική η κατάσταση, διότι έχουμε ακούσει πολλά από τις χώρες σχετικά με τις δικές τους περιφέρειες. Νομίζω ότι είμαστε πολύ πιο αυστηροί όσον αφορά τα αποτελέσματα. Ελπίζω όμως όλα αυτά να συμπέσουν με, την προκαταρκ... με τις προκαταρκτικές εργασίες της Επιτροπής για το πρόγραμμα για το περιβάλλον. Ελπίζω λοιπόν έτσι να έχετε μια επισκόπηση του πώς λειτουργούν οι πολιτικές αυτές. Προσλέπω λοιπόν στην καλή συνεργασία μαζί σας κύριε Πρόεδρε και κύριοι βουλευτές της Επιτροπής Ελπίζω η εμφάνισή μου εδώ να αποτελεί το ξεκίνημα μιας διαδικασίας και ιδιαίτερα ε, προσλέπω στην καλή συνεργασία με τον κύριο Κεμπράντη και ε, θα ήθελα να τον ε, καλέσω στην Κοπεχάγη, αν δεν έρχεται ούτως ή άλλως για τη διάσκεψη. Θα καλώ όμως όλους σας να επισκεφτείτε τον οργανισμό μας. Όπως σας είπα, είμαι στη διάθεσή σας και ανά πάσα στιγμή θα χαρώ να σας δεχτώ στην Κοπεχάγη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Μακλέιτ. Είπατε ότι έχετε εδώ παλιούς φίλους και νέους θα κάνετε τώρα, γιατί πραγματικά εγγράφετε το έργο σας στα πλαίσια των δικών μας εργασιών και της στήριξή μας. Μου είπατε κάτι ενδιαφέρον στην αρχή, ότι είστε σε επαφή με τον οργανισμό ε, για το διάστημα, διότι οι ε, κυβερνήτες αεροσκαφών ε, όταν πετάνε γύρω από την υδρόγειο ε, έχουν ενδιαφέρουσες εμπειρίες. Το ίδιο ισχύει και με τους ε, κυβερνήτες πλοίων. Βλέπουν πράγματα στη φύση που εμείς δεν τα βλέπουμε και από τον ουρανό. Και είναι πολύ ενδιαφέρον να μας τα πείτε και αυτά πράγματα που να καταγράψουμε κι εμείς για τις αλλαγές. Είπατε για την κλιματική αλλαγή 0,8 βαθμοί Κελσίου, θα πει ο άλλος σιγά την αλλαγή. Αλλά στην Αρκτική διπλασιάζεται αυτό και πολλαπλασιάζεται και από πλευράς δραματικών συνεπειών και μόλις επιστρέφεται από ε, μια συνεδρίαση της Σύμβασης της Αρκτικής, έτσι δεν είναι, όπου υπάρχει και μια ενδιαφέρουσα είδηση και ευχάριστη ότι επιτρέπεται να συμμετέχει και η Ευρωπαϊκή Ένωση ως ένωση, γιατί μέχρι τότε συμμετέχουν ε, κράτη, έτσι. Και τώρα είναι πρόοδος αυτό να ε, συμμετέχει η Ευρώπη ως Ευρωπαϊκή Ένωση, να έχει μία φωνή και όχι μόνο ε, να εκπροσωπείται από τη Δανία, εκπροσωπείται και, και ποιον άλλον, τη Σουηδία και τη Ρωσία. Είναι το, το ε, Βόρειο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Εντάξει, υπάρχει και ο Καναδάς εκεί και οι Ηνωμένε Πολιτείε, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση ως Ένωση δεν είχε φωνή και δεν είχε και έδρα. Καλό είναι λοιπόν να δούμε πώς μπορούμε όλοι μαζί να προστατεύσουμε το Βόρειο Πόλο. Ε, αναφερθήκατε στον κύριο ε, Γκαμπράντη που είναι και βασικός σύνδεσμός μας και ζήτησε και πρώτος το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ω ε, άτομο επαφή με τον οργανισμό της ε, Κοπενχάγης είχα ένα γεύμα με την κυρία Μακλέιντ και ένα από τα πράγματα που συζητήσαμε ήταν κατά πόσο αυτή η Επιτροπή Περιβάλλοντος χρησιμοποιεί τον οργανισμό περιβάλλοντο με επαρκή τρόπο, με αποτελεσματικό τρόπο. Μας είπε πω κάποια μεμονωμένα μέλη το πράττουν, αλλά ότι θα ήταν καλό αν ολόκληρη η Επιτροπή αλλά και άλλα μεμονωμένα μέλη μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τον οργανισμό με πιο αποτελεσματικό και καρποφορό τρόπο. Θα ήθελα λοιπόν να καλέσω την κυρία Μακλέιντ να εξηγήσει στην Επιτροπή καταρχήν τι μπορεί να κάνει ο οργανισμός για την Επιτροπή και για τα μεμονωμένα μέλη. Έχω ακόμα μια ερώτηση. Εγώ είμαι πεπισμένο ότι η, πραγματική, η μόνη πραγματική λύση για το πρόβλημα του κλίματος είναι η τεχνολογία και η ανάπτυξη νέας τεχνολογίας, αλλά και η διάδοση αυτής. Και θέλω να ρωτήσω την κυρία Μαγκλέιντ αν έχει κάποιες ιδέες για το πώς θα επιταχυνθεί η ανάπτυξη τεχνολογίας και πώς θα επιταχυνθεί και η διάδοση της ολόκληρο τον κόσμο. Τέλος, ε, άκουσα πως ε, τελευταία η Ευρώπη ε, σημειώνει στέρηση στην ανάπτυξη νέας τεχνολογίας και διρωτώ με αν αυτό είναι αλήθεια. Αν αρχίζουμε να, αρχίζουν να μας ξεπερνούν άλλες χώρες όπως η ΕΠΑ ή η Κίνα. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε τις απαντήσεις σας σε αυτές τις ερωτήσεις. Ευχαριστώ κύριε Σίμερ. Ζέμπερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την κυρία Μακλέιτ για τα ενδιαφέροντα αυτά που μας είπε. Θα ήθελα να συνεχίσω εκεί που σταμάτησε ο προοραλή σα. Για εμάς τους Ευρωβουλευτές θα ήταν επιθυμητό η επαφή ε, μεταξύ της δικιάς σας ε, πραγματογνωμοσύνης και της δικιάς μας δουλειά να αλλάξει σημαντικά και να ε, πάρει σάρκα και οστά στην πράξη. Να μην σας ρωτάμε εμείς για προφορίες. Να έρχεστε εσείς να μας βοηθάτε, αν είμαστε εισηγητές, σκιώδη εισηγητές, να μας εξυπηρετείτε με κάποια βασική προφόρηση για να εμβαθύνουμε στη συνεργασία μας. Στην καθημερινή πολιτική δουλειά που έχουμε δεν ευκαιρούμε πάντα, ούτε έχουμε το χρόνο, ούτε τη δυνατότητα, ούτε και τη βούληση να μπούμε σε διάβλους επικοινωνίας δύσκολους και μακροσκελής. Παρακαλώ, ρωτήστε τους Γενικού σα διευθυντέ, πώ γίνεται να βελτιωθεί καλύτερα να λειτουργεί επικοινωνία με συγκεκριμένες ε, προτάσεις. Γιατί σήμερα νομίζω χωλαίνουν τα πράγματα, δεν είναι απολύτω ικανοποιητικά. Παρακαλώ το ελέγξουμε αυτό, τι μπορούμε να κάνουμε. Τώρα, για την κλιματική αλλαγή. Όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχει η μέση θερμοκρασία παγκόσμια. Ε, έχει αυξηθεί βεβαίως και έχει αυξηθεί ε, και ε, η παραγωγή διοξιδίου του άνθρακα. Αλλά αυτή η αναγωγή, ε, το ένα προς ένα, χρειάζεται εξέταση και έλεγχο. Και θα παρακαλούσα να κάνετε κάποιες προσπάθειες υποστήριξης, γιατί ακούω και επιστημονικές φωνές προς άλλη κατεύθυνση και θα πρέπει να βεβαιωθούμε απολύτως. Όταν κάνουμε τόσο ε, σημαντικές και βαθιές τομές στη ε, βιομηχανία μας και στην οικονομία μας. Επίσης, ξέρουμε ότι αυξάνεται η θερμοκρασία και χρειάζεται προσαρμογή αλλά για την περίφημη συγκράτηση ή περιορισμό το mitigation υπάρχει ακόμα ένα ερωτηματικό και χρειάζεται πολιτικές προτεραιότητες και υποστήριξη από εσά με επιστημονικά δεδομένα, επιστημονικά στοιχεία. Παρακαλώ αυτό να μας βοηθήσετε για να ε, μπορέσουμε να καλύψουμε τα κενά που έχουμε στην επικοινωνία και στην πληροφόρηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Εστρέλα. Σας ευχαριστώ. Και εγώ θα ξεκινήσω ευχαριστώντας την κυρία Μακλέιντ για την παρέμβασή της και για την αισιοδοξία που μας έφερε σε σχέση με τις προσδοκίες τήρησης ε, του πρωτοκόλλου του Κιώτο. Εγώ θα ήθελα να εκφράσω παρόμοια αισιοδοξία και σε σχέση με τις ε, προσδοκίες ε, που έχουμε από την ε, διάσκεψη της Κοπεχάγης. Όμως όταν είπατε πως όλα τα κράτη-μέλη θα καταφέρουν να τηρήσουν το Κιώτο εκτός από ένα, θεωρείτε, μιλήσατε για την Ευρωπαϊκή Ένωση των 15 ή των 27. Γιατί στην προηγούμενη έκθεση ε, τάσεων και προεκβολών Λέγατε ότι μόλις τέσσερα κράτη-μέλη είχαν ε, φτάσει στα όρια του Κιώτου το 2006, ότι υπήρχαν τρία που απήγαν πολύ από την επίτευξη των στόχων αυτών και ότι τα υπόλοιπα πίστευαν ή, εν πάση περιπτώσει, κατέβαλαν προσπάθειες για να ε, επιτύχουν τους στόχους. Τώρα φαίνεται ότι σε αυτά τα τελευταία χρόνια η κατάσταση βελτιώθηκε ε, σε πολύ μεγάλο βαθμό. Μακάρι να έχει γίνει αυτό, γιατί έτσι μπορούμε να σκεφτόμαστε το μέλλον με μεγαλύτερη αισιοδοξία. Η δικιά μου ερώτηση αφορούσε την κατάσταση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. ποια είναι η εξέλιξη που υπήρξε σε σχέση με την τελευταία έκθεση, τη σχετική έκθεση. Και τέλος, μιλήσατε για τις μεταφορές και για το βάρος των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που προέρχονται από τις μεταφορές. Υπήρξε λοιπόν σε αυτό το τομέα κάποια εξέλιξη θετική. Γιατί στην προηγούμενη έκθεση γινόταν μια πρόβλεψη ότι για να επιτευχθούν επιτευχθεί μάλλον η μείωση του 20% αυτό θα δυστυχούσε στο να σταματήσουν όλες οι εκπομπές που οφείλονται στις μεταφορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα οι επιστήμονες λένε ότι αυτό δεν αρκεί. Και βέβαια θεωρώ ότι είναι αδύνατο να περιορίσουμε τόσο δραστικά τις εκπομπές ε, των αερίων του θερμοκηπίου που προέρχονται από τις μεταφορές. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ah, sì, scusi. Allora, io non sono così soddisfatto ο κύριος Ρώση. Εγώ δεν είμαι πολύ ευχαριστημένος από την παρέμβαση της Γενικής Διευθύντριας ε, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, γιατί δεν είπε ούτε μία λέξη για τα αποτελέσματα αυτού που κοστίζει πολύ στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή τις εκπομπές από πλευράς των επιχειρήσεων. Δεν άκουσα ούτε μια λέξη για το πόσες επιχειρήσεις κλείσανε στην Ευρώπη, πόσες χιλιάδες άνθρωποι βρεθήκαν χωρίς μισθό. Ακριβώς λόγω των υπερβολικών πιέσεων σε μια τέτοια περίοδο απέναντι στις επιχειρήσεις και τις εταιρείες, όχι μόνο τις Ιταλικές αλλά τις Ευρωπαϊκές γενικότερα. Εμείς είμαστε βουλευτέ, καθημερινά δεχόμαστε εκπροσώπους τη βιομηχανία, αλλά και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και όλων όλοι αδιακρίτως ε, κλαίνε και οδύρονται ότι αν προχωρήσουμε με αυτόν τον τρόπο θα κλείσουν και άλλες εταιρείε, θα πάνε σε άλλες χώρες. Οπότε αγαπητή κυρία Διευθυντά, η μείωση για την οποία μιλήσατε που δεν είναι και τόσο ψηλή σε σχέση με το 90% είναι και αυτή συνδέεται και με τις εταιρείες που κλείσανε ή που μετεγκαταστάθηκαν. Πήγαν αλλού να δουλέψουν και μολύνουν τις άλλες χώρες αλλά χάσανε οι δικοί μας εδώ τις θέσεις απασχόλησή τους. Και νομίζω πως αυτό το ξέρετε πολύ καλά. Γιατί δεν μας το λέτε, γιατί σε αυτά τα στοιχεία τα μερικώς θετικά για την Ευρώπη όσον αφορά την μείωση των ε, εκπομπών δεν βάζετε και αυτά τα τόσο σοβαρά αρνητικά στοιχεία τα οποία μιλούν για ένα σωρό κόσμο που έχασε τη δουλειά του. Μιλήσατε και γίνεται υπέροχο ψήφισμα της Επιτροπής της εδώ που ψηφίστηκε σχεδόν ε, ομόφωνα μία μόνο ψήφο αρνητική, τη δική μου, ως τμήμα της αντιπροσωπείας της Λέγκα Νόρτ. Γιατί εμείς εκείνο το, τα, εκείνα τα ωραία 30 εκατομμύρια ε, ευρώ, ε, ευρώ ετησίως δεν τα δίναμε στις αναπτυσσόμενες χώρες για να ανταγωνιστούν τις δικές μας επιχειρήσεις, αλλά τα είχαμε δώσει στις δικές μας επιχειρήσεις, γιατί με αυτά τα λεφτά μπορεί και να μείωναν τις εκπομπές χωρίς να διώξουν κανέναν, χωρίς να κατεβάσουν τα ρολά. Γιατί οι εταιρείε που κλείνουν και πάνε απλώ να μολύνουν μια άλλη χώρα δεν σημαίνει πως γενικά κάνουν οικονομία στις εκπομπές ρήπων. Όχι, λιγότερες εκπομπές εδώ και περισσότερες σε, σε άλλες χώρες εκτός Ένωσης. Είναι μια γραμμή λοιπόν που εμεί εδώ στη Λέγκα Νόρτ δεν συμφωνούμε καθόλου. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, μια λεξούλα θα μπορούσατε να μα πείτε ότι χάνουμε θέσει απασχόληση, δεν ξέρουμε πότε θα τι ξαναβρούμε. Εντάξει, όλοι στο κάτω-κάτω είμαστε υπέρ του περιβάλλοντο και εγώ προσωπικά ανέκαθεν ναι, ήμουν υπέρ. Αλλά πρέπει να βάζουμε και κάποια όρια. Να σκεφτούμε λίγο και τη συνείδησή μα και να δούμε σε μια τέτοια φάση όπου 30% των εργαζομένων τη Ευρώπη δυσκολεύονται να βγάλουν το μήνα, εάν χρειάζεται τόσο πολύ να επιμένουμε και να χάνουμε και άλλους βιομηχανικού πόλους που δίνουν δουλειά, θέσεις απασχόλησης. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Ρώση, οι εταιρείε που κλείνουν τώρα κλείνουν περισσότερο λόγω της κερδοσκοπίας των χρηματιστηρίων και των τραπεζών και λιγότερο από το πακέτο πολέμηση της κλιματικής αλλαγής που δεν έχει αρχίσει καν να ισχύει. Το 2013 θα μας έρθει. Έτσι, να λέμε και τα πράγματα με το όνομά τους. Και όταν αποδίδουμε ευθύνε. Ελπίζουμε το 2013 να έχει ανακάμψει η οικονομία και να έχουν έρθει άλλοι καιροί. Και στην Κοπεχάγη βεβαίως και άλλοι, η ΙΠΑ, η Ιαπωνία, η Κίνα, η Ινδία να μας ακολουθήσουν. Και αυτό είναι κριτήριο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, σαφώς, για να πάμε στο 30%. Παρόλο που θα μας έλεγε η επιστήμη, όχι, 40%. Αλλά εντάξει, δεν παίζουμε και την κολοκυθιά και πρέπει να έχουμε υπόψη μας και τις πραγματικότητες και τι μπορούμε να αντέξουμε στην Ευρώπη ως τόπο παραγωγής. Καλά, δεν θέλω να προεξοφλήσω την απάντησή σας. Εσείς απαντήσετε κυρία Μακλέιντ, όχι εγώ. Κρήτον μας τώρα, τελευταίος και μετά απαντήστε. Thank you, Mr. President and uh, Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Μακλέιντ, ε, χαίρομαι που σας ξαναβλέπω στο Κοινοβούλιο. Και επίση ήθελα να σας ευχαριστήσω για την σημερινή σας παρουσίαση αλλά και για το καταπληκτικό έργο που έχετε κάνει για τις Άλπεις. Ε, Μόλις το είδα σύντομα, αλλά πραγματικά είναι εντυπωσιακή η κλίμακα του αντικτύπου στα ευρωπαϊκά ποτάμια και την πρόσβαση στο νερό. Γι' αυτό και θα ήθελα να εστιάσω και στην προσοχή στο για τον μαύρο άνθρακα που παράγεται από τις ε, εξατμίσεις κτλ. Σε μια πρόσφατη συζήτηση ε, για τα Ιμαλάια φαίνεται πως ε, ο μαύρος άνθρακας προκαλεί πολύ γρήγορη στήξη των παγετώνων σε επηρεάζει, ένα σωρό ποτάμια όπως ο Γιάντζι, ο Σαουίν, τεράστια ποτάμια. Δηλαδή βασικά επηρεάζει το νερό ολόκληρης της Ασίας και την πρόσβαση των ανθρώπων σε αυτό. σε περίπτωση που ο μαύρος άνθρακας δεν συμπεριληφθεί σε κάποια συμφωνία στην Κοπενχάγη, εσείς μπορείτε να μας πείτε αν όντως ε, συμβάλλει στο λιώσιμο των παγετώνων στις Άλπες, έχετε σχετικά στοιχεία, μπορείτε να κάνετε οποιασδήποτε πολιτικές προτάσεις για αυτό το θέμα. Σας ευχαριστώ. Πρώτες απαντήσεις μπορούμε να έχουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα προσπαθήσω να απαντήσω στην κάθε μία ερώτηση όσο γίνεται με μεγαλύτερη ακρίβεια. υπάρχουν κάποιες γενικές παρατηρήσεις που θέλω να κάνω καταρχήν. Πώς μπορούμε εμείς ε, να είμαστε πιο άμεση και πιο, να έχουμε μια πιο άμεση επαφή μαζί σας ε, και επικοινωνία, χωρίς τώρα να ανοίξουμε το φράγμα, ε, θέλω να πω ότι είμαστε πάντοτε στη διάθεσή σα όσον αφορά ένα συγκεκριμένο αίτημα για ενημέρωση και όπω σα ανέφερα και προηγουμένω, θα είμαστε σε κάθε συναντήσή σας, ε, συνάντηση τη της Επιτροπής εννοώ, συνεδρίαση, είμαστε πάντοτε λοιπόν εδώ για να μπορείτε να μα απευθύνετε αιτήματα. Για πιο ουσιαστική δουλειά, α πούμε για να στρίξουμε για του εισηγητές, έχουμε φτιάξει με τη γραμματεία ένα τρόπο για να μπορούμε να δουλέψουμε και να οργανώσουμε την εργασία μας ε, για πιο μεγάλες αναλύσεις, πιο εμπεριστατωμένες αναλύσεις. Επίσης, συχνά μπορούμε να σας δείξουμε σημεία όπου συγκεντρώνονται αυτά τα στοιχεία. Δηλαδή, μπορεί να μην κάνουμε εμεί οι ίδιοι πάντα αυτή τη δουλειά, αλλά σίγουρα να σας δώσουμε ονόματα, και ε, συγκεκριμένα σημεία όπου γίνεται αυτή η δουλειά. Είναι μια, μια προσέγγιση open gate, ανοιχτών πυλών, αντί να συνεργαζόμαστε μόνο με τον, ε, με τον ε, εισηγητή. Πραγματικά, εγώ θα ήθελα να είναι πιο πολύ η συνεργασία μας. Τώρα, για να έρθω τώρα στη τεχνολογία και του ένα-δύο μελητέ που αναφέρθηκαν σε αυτό. Πολύ ενδιαφέρουσα συνεδρίαση είχαμε την περασμένη εβδομάδα με τη ΣΥΠΑ. Μία διάσκεψη κορυφή είχαμε με τη ΣΥΠΑ για την έρευνα. Και φυσικά προέκυψε και το θέμα τη τεχνολογία. Ήταν ε, σαφέ ότι η ισορροπία που καθορίζει τη διαφορά ανάμεσα στη ΣΥΠΑ και στην ΕΕ είναι λόγω τη διαφοροποίηση των δαπανών στην έρευνα και ανάπτυξη στο στρατιωτικό τομέα σε αντίθεση με τον πολιτικό. Δηλαδή είναι ένας αντικατοπτρισμός ο μία το άλλο και μπορούμε να πούμε ότι είναι κακό ή καλό για την ΣΥΠΑ, αλλά τελικά ο ρόλος της τεχνολογίας και η ανάπτυξη της τεχνολογίας γίνεται πολύ πιο γρήγορα γιατί υπάρχει πιο συντονισμένη προσπάθεια για την επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων. Αυτό μπορείτε να το θεωρήσετε ως το υπόβαθρο για τα όσα θα σας πω τώρα. Έχουμε πάρα πολλές παγκοσμιοποιημένες ε, επιχειρήσεις που δουλεύουν πολύ καλά εκτός Ευρώπης και τουλάχιστον να πω κάποια σχόλια για τα, τα ιδιαίτερα παθιασμένη παρέμβαση του κυρίου Ρώση, την οποία εκτιμώ. Αλλά επειδή είμαστε σε διάλογο με εταιρείε όπως η Siemens, η Philips, η GI και η General Electric και άλλες από τη δική μας περιοχή εδώ, είναι σαφές ότι περνάμε μία μεγάλη αλλαγή τόσο όσον αφορά την επίλυση των δικών μας προβλημάτων στην Ευρώπη, δηλαδή μια γυρασμένη υποδομή η οποία δεν ταιριάζει απόλυτα στους σκοπούς της, είτε είναι η οι κλιματικέ αλλαγέ δεν είναι οι τηλεπικοινωνίες, η ενέργεια. Ένα σωρό πράγματα θέλουμε να κάνουμε και να φορτώσουμε την υποδομή μα, είτε είναι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια από τοπικέ πηγέ και ούτω καθεξή. Χρειάζεται δηλαδή μια εκβάθρον αλλαγή σε ολόκληρη την Ευρώπη, στην τεχνολογία μα και στι βασικέ μα υποδομέ. Αλλά φυσικά υπάρχει καθυστέρηση ανάμεσα στην κινητοποίηση αυτή τη τεχνολογία, διασφαλίζοντα την νομιμότητα και του κανονισμού σε όλε τι χώρε που θα διασφαλίζουν αυτή τη δυνατότητα, τα στάνταρ για τις πράσινες θέσεις απασχόλησης, αλλά βασικά για την απασχόληση. Εγώ φυσικά δεν έχω έτοιμη λύση για να μην απολύεται ο κόσμος και δεν είναι και δουλειά μου, δεν είναι δουλειά του δικού μας οργανισμού. Εκεί που μπορούμε να παίξουμε ρόλο, και αυτό που νομίζω πως καταλάβα, κατάλαβα από τα όσα είπατε, είναι ότι αυτό που χάνουμε, είναι το τι θα χάσουμε αν δεν έχουμε καλή περιβαλλοντική νομοθεσία. Εάν βάλετε ότι αν, αν, αν φτιάξουμε αυτή την ομοθεσία για τον εθνικό, ε, την οδηγία για τις εθνικές εκπομπές, 46 δις θα από το Εθνικό Σύστημα Υγείας των χωρών. Αυτή είναι ε, η έρευνα, η μελέτη αξιολόγησης. Είτε ο κόσμος είναι πλήρως απασχολούμενο, είτε είναι μερικώς απασχολούμενο, ένα από αυτά που πρέπει εμείς να κάνουμε είναι να διασφαλίσουμε ότι το περιβάλλον δεν επιδεινώνεται και άρα ε, είναι πιθανότερο πως ο κόσμος δεν θα έτυχε να αντιμετωπίσει δύο καταστροφές στον κόσμο του, δηλαδή να τουλάχιστον αποφύγει την αρρώστια. οι περιβαλλοντικές συνθήκες δεν αρκούν, στο, δεν, δεν, δεν μπορούν να αντισταθούν στις κλιματικές αλλαγές. Επίσης διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν πολλές κοινότητες οι οποίες ε, ε, δημιουργούν αυτό, βιώσιμη μάλλον απασχόληση, παράχουν τρόφιμα έναν διαφορετικό τρόπο με τον οποίο λειτουργούν και οι τοπικές οικονομίες. Εγώ πιστεύω και θα πρέπει να είμαι πολύ ειλικρινής ότι υπάρχει πολύ μεγαλύτερο δυναμικό εντός του συστήματος που θα πρέπει να διασφαλίσει την μακροπρόθεσμη απασχόληση αλλά θα πρέπει να συνοδεύεται από επενδύσεις σε νέες υποδομές και νέους τρόπους ε, αντιμετώπισης των κλιματικών αλλαγών και προσαρμογής σε, σε αυτές. Να στραφώ τώρα στο, στη σχέση αιτίου αποτελέσματος και κατά πόσο έχουμε ακόμα κοινωνίες μας που αρνούνται τις αλλαγές. Ναι, μπορούν να υπάρχουν κάποιες χώρες που να διστάζουν για κάποια συγκεκριμένα θέματα και εγώ είμαι πάντοτε υπέρ των να γίνεται ε, επιστημονικός διάλογος όταν έχουμε κάποια βεβαιότητα για ορισμένα θέματα. Αλλά η σχέση αιτιατού είναι αδιαμφισβήτητη. Η αντίδραση των ε, ανθρώπων ε, στον πλανήτη, ε, στην βιομηχανική περιοχή, είναι να αυξήσουν τα αέρια του θερμοκηπίου και τη συγκέντρωση αυτών. Είμαι βέβαιη και πιστεύω πως θα μπορεί κανείς να βρει ακόμα κάποιους ανθρώπους που πιστεύουν ότι η γη είναι επίπεδη. Αλλά αυτό που μπορώ να σας πω με βεβαιότητα πως ολόκληρη την Ευρώπη ήδη υπάρχουν εμφανείς επιπτώσεις της θέρμανσης του πλανήτη. Τώρα, τα διάφορα αέρια, ο μαύρος άνθρακας και τα λοιπά συγκεκριμένα θέματα. Ναι, δουλεύουμε πολύ στενά, συνεργαζόμαστε με ένα πολύ ευρύ φάσμα ερευνητών. Είμαστε διεθνεί, σε αυτό, δεν, ε, δεν, δεν συνεργαζόμαστε μόνο με τους Ευρωπαίους συναδέλφου και θα σας πω ότι στο καλάθι των αερίων αυτά που εμπίπτουν περισσότερο στο θέμα τη ποιότητα του αέρα, δηλαδή τα σωματίδια, ο μαύρο άνθρακα κτλ. Αυτά ήδη συμβάλλουν στις στην κλιματική αλλαγή και στην θέρμανση του πλανήτη. Αλλά οι επιπτώσεις τους είναι ελάχιστες σε σχέση με τα γνωστά αέρια που συμβάλλουν στη θέρμανση του πλανήτη, όπως το μεθάνιο, το μονοξίδιο του άνθρακα, το μονοξίδιο του θείου κτλ. Ε, μπορούμε λοιπόν να επιβάλλουμε κάποια πράγματα, αλλά σε πολύ μικρό βαθμό. Όταν όμως πέφτουν σε πολύ μεγάλες ποσότητες, όπως ο Μαύρο άνθρακα, σε περιοχές όπου αυτό που είναι σημαντικό είναι η επιφάνεια αντανάκλαση, ώστε να διατηρείται η, η ψυχρότητα του, της περιοχής. Εκεί βλέπουμε όντως στα Ιμαλάια ε, έχει το ίδιο, τις ίδιες επιπτώσεις και στις Άλπες είχε το ίδιο, τις ίδιες επιπτώσεις. Αλλά πολλά από αυτά που συμβαίνουν στη Ιμαλάια έχουν να κάνουν μόνο με το παγκόσμιο φαινόμενο των αερίων του θερμοκηπίου. Και ε, υπάρχει ε, σοβαρή βεβαιότητα για το ότι συμβαίνει ε, στα Ιμαλάια έχει άμεση σύνδεση με αυτά που συμβαίνουν στη λεκάνη του Αμαζονίου. Και μάλιστα υπάρχουν πράγματα τα οποία ελπίζαμε πως πραγματικά δεν θα γίνουν. Αυτές οι ευρείες ε, συνδέσεις σε ολόκληρο τον πλανήτη. Η ξύρανση του Αμαζονίου είναι αυτή που προκαλεί τις επιπτώσεις αυτές στο οροπέδιο του Θιβέτ και στα Ιμαλάια. Για να είμαι πιο συγκεκριμένη για το Κιώτο, Έχετε δίκιο. Είναι στο πλαίσιο των 27, ε, της Ευρώπης των 27 που έχουμε τα πιο θετικά αποτελέσματα. Αλλά εμείς έχουμε δώσει τα όργανα τα οποία οι χώρες χρησιμοποιούν. Έχουμε μια συμφωνία και γι' αυτό και θα επιτύχουμε τους στόχους του Κιώτο, γιατί ακριβώς χρησιμοποιήσαμε το CDM και άλλα ε, εργαλεία. Αλλά επιτόπου και εξετάζοντας τις εγκαταστάσεις είδαμε πως ε, σταδιακά γίνεται μια αντικατάσταση και μια μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα ε, και αποδοτικότητα. Φαίνεται να υπάρχει ένα, μια μεγάλη διαφορά ανάμεσα στους τομείς, στους πρωτοπόρους και στους άλλους που είναι πιο αργοί στις νέες τεχνολογίες. Ορισμένοι όμως κλάδοι δείχνουν ήδη πως όχι μόνο ε, θα πετύχουν τους στόχους του Κιώτο, αλλά μπορούν και να τους ξεπεράσουν με βάση πολλές εγκαταστάσεις όσον αφορά την αποτελεσματικότητα στην ενέργεια και άρα στη ε, μείωση των εκπομπών. Είμαι λοιπόν αισιόδοξη γιατί μπορώ να δω τα στοιχεία επιτόπου για πολλές χώρες, αλλά μπορώ επίσης να δω και συλλογικά τα στοιχεία υπό την κατανομή του φόρτου. Έχουμε ένα πακέτο το οποίο θα πρέπει να ε, το επενέσουμε, αλλά πάντοτε βέβαια υπάρχει χώρος για βελτίωση. Νομίζω πως απάντησα σε όλα σας τα ερωτήματα, αλλά αν κάτι ξέχασε παρακαλώ να μου το θυμίσετε. Α, ναι, η τεχνολογία και η διάδοσή της ε, ήταν μια τελευταία ερώτηση και η επιτάχυνση να επανέλθω στην, στο θέμα αυτό. Αν με ρωτούσατε σήμερα πού χρειάζεται η ευρωπαϊκή τεχνολογία, μάλλον πού βρίσκεται η ευρωπαϊκή τεχνολογία σε παγκόσμιο επίπεδο, εδώ, σε βαθμολογία, δεν είναι πολύ μπροστά. Έχουμε την Ιαπωνία, την Νότια Κορέα, συμβαίνουν πολλά πράγματα παγκοσμίω. Αλλά αυτά που χρειαζεται η ευρωπαικη τεχνολογια μαλλον που βρισκεται η ευρωπαικη τεχνολογια σε παγκοσμιο επιπεδο σε βαθμολογια δεν ειναι πολυ μπροστα εχουμε την ιαπωνια την νοτια κορεα συμβαινουν πολλα πραγματα παγκοσμιω αλλα αυτα που συμβαινουν στην Ευρώπη και που δεν συμβαίνει αλλού, ε, και αυτό δεν καθοδηγείται από την νομοθεσία, δεν είναι υποχρεωτικό. Είναι το γεγονό ότι πολλέ εταιρείε τώρα συγκεντρώνονται, δημιουργούν ένα πράγμα αυτό που ε, εγώ θα νομούσα από την αρχή μέχρι το τέλο. Λύσει δηλαδή ολοκληρωμένε από τα κτίρια, με τη συγκεκριμένη τεχνολογία, στι πόλει που φτιάχνει, στι ε, δρόμου που και τα μέσα μεταφορά που χρησιμοποιεί. Και γενικά πιστεύω πω η Ευρώπη είναι πολύ μπροστά όσον αφορά αυτή την ολοκληρωμένη σκέψη. Και ηρωνικά ε, δεν έχουμε κατάλληλη νομοθεσία για να το στηρίξουμε αυτό, γιατί δεν έχουμε κάνει αρκετά για να ολοκληρωθεί, να ενταχθεί η πολιτική μεταφορών στην περιφερειακή πολιτική. Ίσως εκεί λοιπόν πιστεύω θα έπρεπε να αφιερώσουμε μεγαλύτερη προσοχή, να συγκεντρώσουμε πληροφορίες για το τι μπορεί να αποδώσει η ολοκλήρωση όσον αφορά την επάρκεια σε νερό, σε ενέργεια και ε, από πλευράς κοινωνικο-οικονομικών ωφελών. Σα Σας ευχαριστώ, κυρία ε, Διευθύντρια. Ο Σλούτερ τώρα. Uh, σας ευχαριστώ και πάλι που ήρθατε. Δεν συμμερίζομαι την αισιόδοξη θέση σας για τα στοιχεία που μας δώσατε. Από ό,τι κατάλαβε, μόνο μία χώρα δεν ε, πληρεί τους στόχους του Κιώτο. Κάτι παρεξήγησα, διότι βλέπω ότι η Αυστρία απέχει 24% από το, απήχε πέρσι 24% από το στόχο, η, η, Ιρλανδία 11%, το Λουξεμβούργο 26%, το, η Πορτογαλία 9%, η Ισπανία 37% μακριά από το στόχο πέρσι. Όλες αυτές οι χώρες τι ευκαιρία έχουν να πετύχουν τους στόχους εν καιρός και τι είδους μέτρα προτείνεται για να τις αναγκάσουμε. Διότι είναι αναγκασμένε ε, σύμφωνα με του κανόνε Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πώς μπορούν λοιπόν όλες αυτές οι χώρες να φτάσουν του στόχους του Κιώτο. Διότι ε, αν δεν του φτάσουν, ε, δεν θα έχουμε καλή διαπραγματευτική θέση στην Κοπεχάγη. Και επίσης όσον αφορά τη συνολική μείωση των εκπομπών, το 1990 οι εκπομπές για τη Γερμανία αν δούμε τη μείωση από το 1990 στη Γερμανία, ε, η μείωση της Γερμανίας είναι μεγαλύτερη από ότι ε, στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρώτον, επειδή είναι πολύ καλή η πολιτική, ε, αλλά και δεύτερον λόγω της αποβημηχανοποίησης της Ανατολικής Γερμανίας. Αυτό όμως μία φορά γίνεται πόσο μεγάλο μέρος των στόχων μας έχουμε πετύχει με τους συνηθισμένους τρόπους. διότι από τον Απρίλιο 2008 μέχρι 2009 είχαμε και μείωση λόγω της οικονομικής κρίσης. Πώς θα πετύχουμε το υπόλοιπο, διότι έχουμε πολύ, ε, καλό, πολύ ευνοϊκό έτος σε σύγκριση το 1990. Το υπόλοιπο όμως θα είναι το πιο δύσκολο κομμάτι. Και τι γίνεται με τα εισαγόμενα προϊόντα ναι, 10,5% των παγκοσμίων ε, εκπομπών, αλλά αν υπολογίσουμε και τα, τα εισαγόμενα προϊόντα, ε, ξεπερνάμε κατά πολύ το 10,5% λόγω της κατανάλωσής μας. Και βέβαια υπάρχει και το πρόβλημα των τομέων που δεν συμπεριλαμβάνονται στο Κιώτο, που αυξάνονται. Συγγνώμη που σας ε, χαλάω τα, τη διάθεση, αλλά για να πετύχουμε τους στόχους μας θα πρέπει να δούμε τα προβλήματα αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Αυτή τη βδομάδα θα μιλήσουμε για τη διάσκεψη της Κοπεχάγης. Αύριο θα συναντηθούμε με τον ε, Επίτροπο Σταύρο Δήμα. Στην ημερήσια διάταξη βλέπω αρκετά θέματα που συνδέονται άμεσα μεταξύ τους. Το αναφέρω αυτό εδώ, διότι αυτά που άκουσα από σας ε, κύριε Διευθύντρια στηρίζουν τη θέση μου. Ήταν πολύ ενδιαφέρον να ακούσουμε τέτοιες αξιόπιστες και επίκαιρες πληροφορίες. Από το 1990 είχαμε μείωση των εκπομπών. Δέκα τόνους κατά κεφαλήν ε, που είναι Πολύ καλό στοιχείο σε σύγκριση με άλλες ε, ε, ε, βιομηχανικές χώρες. Όπως υπόθηκε, τα 15 κράτη-μέλη από ένα πληρούν τους στόχους του Κιώτο. Υπάρχει όμως και ένα άλλο σημαντικό νούμερο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ευθύνεται για το 10,5 των παγκοσμίων εκπομπών. Δεν υπάρχουν τοπικές λύσεις στα παγκόσμια προβλήματα. Το 10,5% είναι το μερίδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να προτείνει μόνο εγχώριες λύσεις, εσωτερικές λύσεις. Όταν συζητήσαμε το σχέδιο του ψηφίσματος για τη διάσκεψη της Κοπεχάγης, 7 στους 10 ομιλητές μίλησαν για την ευθύνη των Ηνωμένων Πολιτειών ο Αντιπρόεδρος έκανε μια πολύ ωραία πρόταση στο Στρασβούργο είπε ότι υπάρχει διαφορά στην οτροπία του Αμερικανικού κοινού και της Αμερικανικής κυβέρνησης. Ίσως θα μπορούσαμε να του στείλουμε προτάσεις. Εμείς είμαστε άμεσα εκλεγμένοι από το Ευρωπαϊκό Κοινό και, η, και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έχει πολύ ισχυρή εκπροσώπηση στη διάσκεψη της Κοπεχάγης. Η αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου θα έχει ισχυρή θέση αν έχουμε να παρουσιάσουμε καλά αποτελέσματα. Το, η μείωση 20% ήταν φιλόδοξος στόχος, ε, ο δρόμο που ακολουθούμε είναι ο σωστός. Ε, η λύση δεν είναι να αυξήσουμε το όριο στο 20% με βάση τα επιτεύγματά μας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορεί στην Κοπενχάγη να πει ότι ζητάμε από τις Ηνωμένε Πολιτείες να κόψουν τις εκπομπές τους, να μειώσουν τις εκπομπές τους. Μια ισχυρή αντιπροσωπεία της του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα μπορέσει να ε, ε σχεδόν να απαιτήσει από τις Ευρωπαϊκές Ένωσης. Δεν θέλω να πω να ε, απαιτήσει ή να εξαναγκάσει, αλλά θα μπορέσει να ασκήσει πίεση στις ΗΠΑ για να μειώσει τις εκπομπές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριο Ζιλ Παρνιού. Μάλιστα, κυρία Πρόεδρε. Κυρία Γενική Διευθύντρια, με μεγάλη χαρά σας γνωρίζω και ως νέος Ευρωβουλευτής, με μεγάλη χαρά προσβλέπω στη συνεργασία μαζί σας. Η κυρία Λεπάζ, όπως και εγώ, ε, κλεγόμαστε στη μεγάλη περιφέρεια της βορειοδυτικής Γαλλίας και θα χρειαστούμε την εμπειρογνωμοσύνη σας, διότι στη Γαλλία υπάρχουν πολλοί επιστήμονες που παραλίγο να γίνουν και υπουργοί, που βρίσκονται στο αντίθετο άκρο, στον αντίποδα των όσων μας λέτε εσείς, δυστυχώς. Και στην αρχή και στη δευτερολογία σας. Λοιπόν, χρειαζόμαστε αυτή την πραγματογνωμοσύνη, αυτή της ποιότητας που παρέχετε εσείς ως Διευθύντρια του Οργανισμού της Κοπενχάγης. Επιτρέψτε μου λοιπόν να κάνω τις εξή τέσσερις παρακαλώ ερωτήσεις, πολύ σύντομα. Πρώτη ερώτηση ε, για τους δύο βαθμούς Κελσίου. Έχω εδώ κάποια συμπεράσματα του Συμβουλίου Υπουργών των Βρυξελών τις προάλλες 29 ε, ε, και 30 Οκτωβρίου και κάθε φορά επανέρχονται σε αυτή τη βούληση που θα πρέπει να έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τους δύο βαθμούς. Και σε σχέση με τα όσα είπατε στην αρχή για το 0,8 αύξηση βαθμού Κελσίου τα τελευταία χρόνια, ε, πώς θα γίνει αυτό τώρα, πώς είναι δυνατόν να έχουμε πιο συγκεκριμένες προτάσεις, να πούμε όχι από τώρα δύο βαθμοί, αλλά η διαφορά από το 0,8 και συν 2, όπως είπατε προηγουμένως. Δηλαδή να επανέλθουν ε, ε, στην επιστημονική αλήθεια αυτά τα δεδομένα. Ερώτηση δεύτερη. Στο ίδιο Συμβούλιο αναφέρθηκε ότι για τη διακυβέρνηση χρειάζεται ένα θεσμικό αρχιτεκτόνημα πριν τη χρηματοδότηση και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ε, λέει ότι θα πρέπει να γίνει ένα φόρουμ υψηλού επίπεδου υπό την αιγίδα λέει των Ηνωμένων Εθνών. Ο δικός σας οργανισμός. Πώς μπορεί να εγγραφεί σε αυτή την προσπάθεια διακυβέρνησης μαζί μας έτσι ώστε να αναπτύξουμε και όλες τις ε, εμπειρογνωμοσύνες και όλη τη γνώση που μπορεί να έχετε φύση και θέση. Ερώτηση τρίτη. Δημόσια χρηματοδότηση. Και εδώ το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το εξέτασε αυτό το θέμα. Εσείς πώς το βλέπετε. Είναι σημαντικό να θυμίσει κανείς σε σχέση με τα όσα ακούγονται που είναι έτσι, τελείως ε, άστοχα αυτά που είπε ο κύριος Ρώση και χαίρομαι για την πρώτη απάντηση που του έδωσε ο κύριος Λάινεν. Αλλά ε, βλέπουμε όμως ότι υπάρχει ανάγκη για διεθνή δημόσια χρηματοδότηση που να λαμβάνει υπόψη και τις αναπτυσσόμενες χώρες. Ε, να υπάρχει αυτή η ισόρροπη ανάπτυξη. Αυτό ισχύει για τη δημόσια χρηματοδότηση, επαναλαμβάνω, ε, όπως είπε ε, περασμένη εβδομάδα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, αλλά και για την ιδιωτική. Έτσι θα μπορούσατε να μας κάνετε μερικά σχόλια και να μας πείτε και την αίσθησή σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Ζιλ. Η Καθλίν Βαν Ευχαριστώ Πρόεδρε. Συγχαρητήρια και για τα όσα μας είπατε. Πολύ αισιόδοξα ήταν και πολύ ε, εύστοχα. Και καλό είναι να δείχνουμε και τέτοια αισιοδοξία παραμονέ Κοπεχάης. Δεν βλάπτει. Τούτου λεχθέντος, θα ήθελα να μου επιβεβαιώσετε, σωστά κατάλαβα αυτό που λέτε, ότι στα 15 κράτη-μέλη με εξαίρεση ένα κράτος ε, τηρεί τους στόχους του Κιώτο, ανεξάρτητα από την οικονομική ύφεση που ζούμε τώρα. Με άλλα λόγια, όταν ανακάμψει η οικονομία με το καλό, που σιγά σιγά ξεκινάει, τότε δεν θα έχουμε προβλήματα. Θα φτάσουμε στους στόχους μας. Σωστά το κατάλαβα αυτό. Σωστά το άκουσα. Μπορείτε να μου το επιβεβαιώσετε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και αυτό σημαίνει ότι ένας από τους σημαντικούς στόχους είναι ότι μπορούμε να ε, συνδυάσουμε την οικονομική πρόοδο ε, με ε, τα θέματα του διοξιδίου του άνθρακα. Κάτι άλλο που είναι πολύ μεγάλη πρόκληση, καλά έτσι κι αλλιώς είναι μεγάλη πρόκληση το κλίμα, αλλά εγώ δεν είμαι τόσο πεσιόδοξη για τη βιομηχανία μας. Μπορεί να σας φαίνεται περίεργο, αλλά έχω την εντυπωσιότητα ότι στους μεγάλους κλάδους της οικονομίας υπάρχει η βούληση και η πεποίθηση να προχωρήσουν βέβαια με την απαραίτητη υποστήριξη της τεχνολογίας να κάνουν τις μεταρρυθμίσεις που χρειάζεται. Αυτό δεν ισχύει για τις μεταφορές, το είπατε κι εσείς η ίδια. Πέντε χρόνια ήμουν υπουργό μεταφορών και ε, πραγματικά προσκρούει κανείς σε ένα τείχος απογοήτευσης και δεν καταφέραμε να το τρυπήσουμε αυτό. Δεν μπορούσαμε να αλλάξουμε την ε, νοοτροπία. Ε, σιγά σιγά στη μεταφορά των επιβατών κάτι κάναμε, δημόσιες συγκοινωνίες ή άλλες συγκοινωνίες, αλλαγή τεχνολογίας, αλλά στις οδικές μεταφορές τείχος πραγματικά. Και σας ερωτώ, έχετε ιδέες σε ευρωπαϊκό επίπεδο πώς μπορούμε να αντιστρέψουμε αυτή την τάση. Όντως και αυτό πρόκληση είναι. Στη συνέχεια έχουμε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και θέλω να ρωτήσω κυρίως τι γίνεται στα κράτη-μέλη. Υπάρχουν πολύ μεγάλες διαφορές και στα 15 σε ό,τι αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και δεν έχει σχέση αυτό με τους ιδίους πόρους κάθε χώρας, αλλά ε, με την πολιτική που ασκεί. Η δική μου χώρα, ε, το Βέλγιο, πραγματικά έχει πολύ κακές επιδόσεις. Αλλά ακόμα, ε, δούμε τι γίνεται στη Γερμανία, ε, που δεν είναι και πιο λιόλου στη χώρα, εντάξει, καταλαβαίνετε. Εκεί να δείτε βροχή. Αλλά η Γερμανία έχει πάρα πολύ καλύτερες επιδόσεις. Η δική σας υπηρεσία, ο οργανισμός σας έχει καλά στοιχεία, στατιστικά, όχι απλώς κάποια αθροίσματα δεδομένων, αλλά στοιχεία που να μας βοηθήσουν να εντοπίσουμε γιατί υπάρχουν αυτές οι διαφορές και πού ε, οφείλονται, για να μπορέσουμε να πιοέσουμε ή να πείσουμε τα κράτη-μέλη να κάνουν πολύ περισσότερα και να ποντάρουν πολύ περισσότερο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Γιατί η πίεση θα πρέπει να έρθει από το κράτος πρώτα απ' όλα. Ευχαριστώ. Dernière question avant de vous donner la parole et de <laughs> redonner la parole à nos collègues. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Τρεμόπουλος. Ευχαριστώ. I'll speak in ε, Greek language. σήμερα στην ε, Βαρκελόνη το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μίλησε για πολιτικά δεσμευτική δήλωση, declaration. Βλέπουμε μια διαρκή προσπάθεια να υποβαθμιστεί η νομική δέσμευση που θα απορρέει από το COP15, γιατί ακριβώς στην αρχή μιλούσαμε για συνθήκη, για τρίτη, μετά για πλαίσιο, framework, και τώρα μιλάμε για αυτή την πολιτικά δεσμευτική δήλωση, την declaration. Τι συμβαίνει ακριβώς, ποια είναι η δική σας γνώμη. Και ακόμη, πώς κρίνεται το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν προωθεί πιο φιλόδοξους στόχους, καθώς όπως έχει δηλώσει η Επιτροπή IPPC, πρέπει να μειώσουμε τις εκπομπές κατά 40% μέχρι το 2020 και 80% μέχρι το 2050. Ευχαριστώ. Madame Ευχαριστώ, κυρία Μακλέιτ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να διευκρινίσω τι θα περιέχεται στην έκθεση της επόμενης εβδομάδας, γιατί δεν έχω ε, αντίγραφό της μπροστά μου. Εν μέρη, αυτό θα απαντήσει στην ερώτηση του Κάρλ που είναι όντως πολύ σωστή. Φυσικά θα πρέπει να κάνουμε πολύ περισσότερα. Να πω καταρχήν ότι όχι δεν συμπεριλαμβάνει τις επιπτώσεις των εισαγωγών και της κατανάλωσης. Είναι λοιπόν απόλυτα σαφές ότι κάνουμε το ελάχιστο όσον αφορά το σύνολο των ε, εκπομπών του θερμοκηπίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και, του, ε, ε, και της επακέντρωσης του προβλήματος στο επίπεδο των οικοκυριών. Θα, μπορεί, θα μπορούσε λοιπόν να είναι κανείς πολύ απεσιόδοξος. Εάν όμως θεωρήσουμε ότι θα έχουμε μεγαλύτερο αποτέλεσμα αν εξετάσουμε την βιομηχανία ως επίκεντρο των προσπαθειών μας, Νομίζω ότι αυτό που έχουμε μπροστά μας αποτελεί πολύ λογική ομάδα πολιτικών και στόχων. Δεν λέω λοιπόν ότι δεν μπορούμε να καταφέρουμε κάτι καλύτερο σε επίπεδο νοικοκυριών και ατομική κατανάλωσης. Δεν έχουμε λύσει όμως το πρόβλημα του αποτελέσματος rebound, δηλαδή αν ε, βελτιώσουμε ε, τα μοτίβα κατανάλωσης ε, και αυτό μεταφράζεται σε περισσότερα χρήματα στην τσέπη μας, τότε μπορεί να ξαναεπενδυθούν τα χρήματα αυτά η ε, βιομηχανία ενδιαφέρεται για κάτι τέτοιο. Δηλαδή, εάν ε, εξοικονομήσουν κάποια πράγματα, ε, τότε θα, θα μπορούν να, τα, να ξαναεπενδύσουν τους ε, πόρους ε, αυτούς για να βελτιώσουν ακόμα περισσότερο την αποτελεσματικότητά τους. Αυτό ως σκέψη. Υπάρχουν πάντως προγράμματα κινήτρων. Να επανέλθω στα νούμερα. Η έκθεση της επόμενης εβδομάδας επικεντρώνεται στις στα 27 κράτη-μέλη. Φυσικά κάποια από τα κράτη αυτά δεν έχουν στόχους του Κιώτο, αλλά τα, τα 15 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν θυμάμαι, νομίζω ότι εσεί μου, ε, μου κάνατε τη σχετική ερώτηση. Μιλάμε για τις 15 ε, ευρωπαϊκές χώρες και από τις χώρες αυτές μόνο μία δεν θα έχει πετύχει το στόχο. Δεν είναι αδύνατο κάτι τέτοιο, διότι ε, βλέπουμε τώρα τη χρήση όλων των σχετικών μέσων και βλέπουμε ότι συμπεριλαμβάνεται το σύστημα ε, εμπορίας ε, των εκπομπών, ε, δεν εξετάζεται όμως σε επίπεδο κρατών μελών. Μπορούμε να εργαστούμε μόνο με βάση τα στοιχεία που έχουμε στα χέρια μας. Ε, είμαι όμως ε, πεπισμένη ότι τα στοιχεία αυτά ε, πηγαίνουν προς τη σωστή κατεύθυνση. Βρισκόμαστε στο σημείο αυτό και νομίζω γενικά ότι θα πρέπει να πάτε με αυτοπεποίθηση στην Κοπεχάγη διότι μπορούμε να κάνουμε πολύ περισσότερα, διότι διότι εμείς κάνουμε αυτό που πρέπει, έτσι μπορούμε λοιπόν να ζητήσουμε και από άλλους να το κάνουν ο κύριος Ρώση ξεκίνησε μια συζήτηση σχετικά με τη διαρροή του άνθρακα, τη μετακατάσταση των εκπομπών. Δεν νομίζω ότι θα έχουμε μια ε, τεράστια φυγή ε, βιομηχανιών και οι ε, επικεφαλείς της βιομηχανίας αρνούνται ότι ότι έχουν μεταφέρει τα εργοστάσια τους άλλου. Κοιτάξτε τις επιχειρήσεις αυτές και σχηματίστε τη δική σας άποψη. Νομίζω όμως ότι πολλές από αυτές τις βιομηχανίες θα ήθελαν να συζητήσουν το, το θέμα αυτό μαζί σας. Είτε ε, μετράμε το διοξείδιο του άνθρακα είτε ε, μετράμε ε, άλλους παράγοντες και πόσο μάλλον να εξετάζουμε και την Ινδία και την Κίνα. Πολύ θα χαρώ να επισκεφτώ την βορειοδυτική Γαλλία, να φάω και μύδια. Πολύ ευχαριστώ θα έρθω. Να φάω και στρίδια. Παρατήρηση εκτός μικροφώνου, δεν την ακούσαμε. Θα έρθω την κατάλληλη εποχή, λέει ο αλλά ε, να σοβαρευτούμε. Μιλάμε για τον στόχο των 2 βαθμών Κελσίου. Θίξατε το θέμα αυτό, πρόκειται για παγκόσμιο στόχο. Και είναι η καλύτερη προσπάθεια ε, της επιστημονικής κοινότητας. Όταν μιλάμε για 450 μέρη ανά εκατομμύριο, αυτό μας δίνει μόνο 50% ε, δυνατότητα να πετύχουμε το στόχο μας. Ε, βέβαια, αυτό είναι πολύ συνδυσμένο όταν αγοράζει κανείς ασφάλιση. Όταν μιλάμε για τους δύο βαθμούς Κελσίου, ένας βαθμός απομένει. Και όπως σας είπα, η Αρκτική ήδη έχει ξεπεράσει τα όρια και η Ευρώπη ακόμα κοντεύει να ξεπεράσει τον έναν βαθμό Κελσίου. Το να διατηρήσουμε δηλαδή την αύξηση στους δύο βαθμούς Κελσίου σημαίνει ότι θα πρέπει να εργαστούμε πάρα πολύ σκληρά και φυσικά δεν μπορούμε να το κάνουμε μόνοι μας. Αρκετοί από εσά ε, ανέφεραν ότι ευθυνόμαστε για το 10,5 των ε, παγκοσμίων εκπομπών και μάλλον θα πρέπει να συνεργαστούμε ακόμα πιο στενά με τους διεθνείς μας εταίρους. Όσον αφορά τα χρηματοοικονομικά, φυσικά μας ενδιαφέρει, ε, παρότι δεν είναι το κύριο θέμα του οργανισμού μας ε, η, ε, η διεθνής χρηματοοικονομική κατάσταση. Φυσικά ε, θέλουμε να δούμε πώς μπορούμε να επωφεληθούμε καλύτερα από ένα ε, χρηματοοικονομικό πακέτο. Τα, οι δαπάνες αυξάνονται κάθε μέρα και οτιδήποτε κάνουμε σήμερα αποτελεί ασφάλιση ώστε να πληρώνουμε λιγότερα στο μέλλον και όσον αφορά ε, ανθρώπινες ζωές και όσον αφορά τη στήριξη της οικονομίας. Νομίζω ότι η ευρωπαϊκή θέση να υπάρχει ένα ε, γρήγορο χρηματοοικονομικό πακέτο και μετά ένα πιο μακροπρόθεσμο αποτελεί πολύ σωστή προσέγγιση. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντική η χρηματοδότηση του δημοσίου τομέα. Δεν θα πρέπει να υποτιμηθεί ως καταλήτης για τις ιδιωτικές επενδύσεις. Και θα ήθελα να τονίσω την ανάγκη των ε, συμπράξεων με τον ιδιωτικό τομέα που χρειάζεται να γνωρίζουν ε, ότι λειτουργούν μέσα σε ένα γνωστό πλαίσιο. Όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, Υπάρχει ένας μεγάλος όγκος δουλειάς που έχει γίνει, που συνεχίζουμε να επικαιροποιούμε, που έχει να κάνει με τις ανανεώσιμες ε, πηγές ενέργειας και τη χρήση τους ε, στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Μιλάμε για αιωλική ενέργεια, βιομάζα, θα υποβάλουμε έκθεση για τις θαλάσσιες μορφές ενέργειας και Θέλουμε να διατηρήσουμε την ορμή που υπάρχει στον τομέα αυτό και να αναλύσουμε περαιτέρω γιατί υπάρχει μεγαλύτερη χρήση των ε, μορφών αυτών ενέργειας σε κάποιες χώρες και το θέμα ε, δεν, ε, είναι αφο... δεν αποκλειστικά τεχνολογικό ή οικονομικό, έχει να κάνει και με την αποδοχή του κόσμου στις διάφορες χώρες. Στις αρχές της χρονιάς υποβάλαμε μια έκθεση, δημοσιεύσαμε μια έκθεση για την αιωλική ενέργεια και είδαμε ότι ε, υπάρχει δυνατότητα παραγωγής 8 φορές της ενέργειας της Ευρώπης ε, με την αιωλική ενέργεια. Υπάρχουν βέβαια κάποιοι περιορισμοί, προστασία ε, οικοσυστημάτων κλπ. Με τους περιορισμούς αυτούς μειώνεται στο, στις δύο φορές, στο διπλάσιο της ενέργειας της Ευρώπης. Υπάρχει λοιπόν αντίσταση από το κοινό, η δυνατότητα όμως υπάρχει θα πρέπει να εξετάσουμε το θέμα αυτό. Επίσης, πολύ θα θέλαμε να έχουμε μια συζήτηση ε, σχετικά με την ε, ιδέα ότι θα μπορούσαμε, αν για παράδειγμα υπάρχει ένα παρομετρικό ε, χαμηλό στον Ατλαντικό και υπάρχει ε, άνεμος από τη δικιά μας μεριά, θα πρέπει να υπάρξει εξισορρόπηση των διαφόρων μορφών εναλλακτική ενέργειας. Επίσης θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι ε, το... Το όσον αφορά το συνεχές ε, ρεύμα θα πρέπει να ε, το έχουμε και αυτό υπόψη. Θα μπορούσε, θα μπορούσε να συνδεθεί η Δανία για παράδειγμα τις ΗΠΑ μέσω καλωδίων στη Βόρεια Θάλασσα. Είναι πολύ, ε, το Ηνωμένο Βασίλειο, συγγνώμη. να σας δώσω μια ιδέα τις Ηνωμένε Πολιτείες υπάρχουν 293 ε, κρατικοί και ομοσπονδιακοί κανονισμοί που εμποδίζουν την εξάπλωση των ανανεώσιμων ε, μορφών ενέργειας. Αυτό όμως παρόλα αυτά γίνεται. Υπάρχουν τρόποι δηλαδή. Να πω επίσης ότι δεν έχω παρακολουθήσει το τι πραγματοποιείται αυτή τη στιγμή στην Βαρκελόνη. Δεν μπορώ λοιπόν να σχολιάσω. Ε, Πολύ ευχαριστώ όμως μετά τη σημερινή συνεδρίαση θα ενημερωθώ και θα επανέλθω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Διευθύντρια. Thank you, Madam Chairman, and thank you. Ο κύριος Μπας σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ στην προηγούμενη δουλειά μου χρησιμοποιούσα πάρα πολύ τις εκθέσεις σας και ήταν πάρα πολύ χρήσιμες για μένα, πολύτιμες. Τώρα ε, βλέπω το πρόγραμμα εργασίας σας για το 2010 και θέλω να δούμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τις σχέσεις μας, τις επαφές μας, τι κάνετε εσείς εκεί και τι χρειαζόμαστε εμείς για τη χάραξη πολιτικής. Βέβαια είναι πολλοί στόχοι, μιλάμε για πολλούς στόχους και μέχρι τώρα για την ενέργεια και την ενεργειακή πολιτική όλα αυτά καλά, αλλά τώρα το μεγάλο θέμα είναι η υλοποίηση και η υλοποίηση όλων αυτών μετά το 2020, γιατί του χρόνου τον Ιούνιο τα 27 κράτη-μέλη θα φέρουν τα σχέδια εφαρμογή και θα κοιτάξουμε μέχρι το 2020 τι θα κάνουμε και πώς θα φτάσουμε στους στόχους. Ωραία, αλλά ξέρουμε ότι όλα αυτά δεν φτάνουν. Μιλάμε για μια νέα ανανεώσιμη πράσινη οικονομία. Μετά το 2020 τι μέλη γενέστε. Καλό θα ήταν λοιπόν να γίνει μια τέτοια ανάλυση. Ποια είναι τα πολιτικά εμπόδια ή φραγμοί που πρέπει να πέσουν, τι πολιτικέ ε, χρειάζονται, τι επενδύσει, για να πάμε σε πιο μακρόπνοα σχέδια ας πούμε, πώς θα γίνει αυτή η μετάβαση και στον ηλεκτρισμό, ε, στα νέα σχέδια, τι επενδύσεις χρειαζόμαστε τώρα, να μην μας γίνει αμονή ιδέα ο στόχος του 2020 και μετά τι. Γιατί είναι πολύ επικίνδυνο κατά την άποψή μου. Έχουμε κολλήσει εκεί ε, μέχρι το 2020 και μετά δεν θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Και μια επιπλέον συγκεκριμένη ερώτηση Άλλο θέμα πολύ σημαντικό για μας, ε, το Κοινοβούλιο του χρόνου, είναι τα βιοκαύσιμα, βιομάζα κτλ. Και μιλάμε πολύ για την ε, έμεση αλλαγή χρήση γη εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι κάνετε, λοιπόν, χαίρομαι πάρα πολύ για τα όσα ήδη έχετε κάνει για τα βιοκαύσιμα, αλλά αυτές οι έμεσε αλλαγέ χρήση γη Ευρω... εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση, επαναλαμβάνω, πώ μπορούν να αποφευθούν τι κάνει ο οργανισμός σας λοιπόν για να προετοιμάσει την επόμενη χρονιά και σε αυτό το συγκεκριμένο και πολύ σημαντικό πεδίο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ η Πρόεδρος. Ο κύριος Κυλακάκης παρακαλώ. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Μακλέιτ για την παρουσίασή σας. Εγώ έχω δύο ειδικές ερωτήσεις. Ερώτηση πρώτη. Γνωρίζουμε ήδη από τώρα ότι ό,τι και αν κάνουμε σήμερα για συγκράτηση της κλιματικής αλλαγής, για τα επόμενα 20, 30, ίσως και 40 χρόνια θα πρέπει να προσαρμοστούμε σε κλιματική αλλαγή στην οποία ήδη είμαστε προγραμματισμένοι και εγκλωβισμένοι. Η έκθεσή σας είναι εξαιρετική και την είδα για τη σάλπης για την περιφερειακή ε, κλιματική αλλαγή και προσαρμογή και διερωτώ με μήπως το 2010 θα μπορούσαμε να δούμε ε, το ίδιο θέμα για την Νότια Ευρώπη και ε, τις ε, των βασών. Διότι όπως γνωρίζετε έχουμε εγκρίνει ένα ψήφισμα με 640 ψήφους υπέρ στο Κοινοβούλιο. Ανησυχούμε πάρα πολύ για τις δασικές πυρκαγιές ε, και αυτά συμβαίνουν τώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι δε προβλέψεις λέγουν ότι θα επιδεινωθεί η κατάσταση τα επόμενα χρόνια και έχουμε 30-40 χρόνια μπροστά μας τέτοιων εξελίξεων. Έτσι. Αυτή είναι η πρώτη μου ερώτηση. Ερώτηση δεύτερη. Ε, φορά ένα ευρύτερο πλαίσιο. Μιλήστε πολύ για τις μεταφορές. Εξ όσων εγώ καταλαβαίνω, στις μεταφορές έχουμε μεγάλο πρόβλημα, αλλά πολύ διαφορετικές πολιτικές ανακλάδο που δίνει το Συμβούλιο. Το Συμβούλιο τώρα εγκρίνει, ας πούμε, μείον 20% για τις θαλάσσιες μεταφορές, μείον 10% για τις αερομεταφορές για το σιδηρόδρομο. Όχι άμεσα μεν, αλλά έμεσα έχει ήδη ενταχθεί σε ένα πάρα πολύ σκληρό μέτρο πολιτικής, διότι είναι ηλεκτροκίνητα τα τρένα και στις οδικές μεταφορές τίποτα. Ανοιχτά όλα, στον αέρα. Ερωτήσεις λοιπόν δύο έχω σχέση, σχέση με αυτό. Πρώτον, έχετε στοιχεία πώς να το πω, για τη, σχέση, τη σχετική συμμετοχή του κάθε κλάδου στη ρήπανση. Η χειρότερη ρήπανση την προκαλούν οι θαλάσσιες μεταφορές ή μήπως οι αεροπορικές ή μήπως οι οδικές. Τι πταίει περισσότερο και πώς ανταγωνίζονται μεταξύ τους αυτοί οι κλάδοι, γιατί είναι ανταγωνιστικοί μεταξύ τους. Και αν έχουμε διαφορετικές πολιτικές για το πώς θα τις αντιμετωπίσουμε τελικά, μπορεί να είναι ε, το αποτέλεσμα όχι επιθυμητό και παρενέργειες και από πλευράς δίπασης και από πλευράς οικονομικής. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Σίλντερς. Ευχαριστώ. Βρίσκω την ε, εισήγησή σας εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και καλωσορίζω την προσφορά σας για εμπειρογνώμονες που θα στηρίξουν τη δουλειά μας. Εγώ είμαι νέα ευρωβουλευτής από την Ελλανδία και είμαι ευτυχής που επιτέλους υπογράφηκε και από την Τσεχία η νέα συνθήκη και οι επιπτώσεις στις, ε, στο κλίμα θα είναι σημαντικές. Θέλω και εγώ να ρωτήσω για τα βιοκαύσιμα και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Δεν χρειάζεται να τα επαναλάβω λοιπόν, τα είπαν και άλλοι ομιλητές και θα περιμένω την απάντησή σας ευχαριστώ. Η κυρία Μισελ Ριβάζη. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ κυρία Διευθύντρια. Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω αν έχετε δεδομένα για τη σύγκριση των στρατηγικών των διαφόρων χωρών για την μείωση ε, των αερίων του θερμοκηπίου. Γιατί το παράδειγμα, ας πούμε, του φόρου άνθρακα. Το ότι επιβάλλει κανείς ένα φόρο άνθρακα που υπάρχει στη Γερμανία, για παράδειγμα, στην Αγγλία και τώρα το φτιάχνουν και το ίδιο και στη Γαλλία. Έχει σημαντικό αντίκτυπο στην μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Και έπειτα, ε, εσείς τι πιστεύετε για αυτή την ε, χρήση αυτού του φόρου χωρί να λαμβάνουμε υπόψη την ενέργεια. Γιατί ο φόρος για τον άνθρακα χρησιμοποιεί μόνο την ε, ορυκτή ενέργεια. Αλλά δεν ε, χρησιμοποιεί άλλου είδου ενέργεια όπως η ηλεκτρισμός που σε αντιστάθμισμα θα αναπτύξει την ηλεκτρική θέρμανση και την πυρηνική ενέργεια. Δηλαδή τελικά πάλι θα αυξηθούν τα αέρια του θερμοκηπίου. Δεύτερο θέμα Συχνά γίνεται λόγος για τις ε, οδικές μεταφορές, κυρίως μέσω των ε, φορτηγών, που συμβάλλουν στις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου. Τι πιστεύετε για τους φόρους άνθρακα στα σύνορα. Αντί να συγκρίνουμε το μεταφορές με τις ε, θαλάσσιες και με τις οδικές μεταφορές, υπάρχει ένα πράγμα φρικτό στο σύστημά μας, ότι ορισμένα προϊόντα, να δώσω ένα παράδειγμα ας πούμε για το ΕΝΔΡΗ στη Γαλλία, πάει στην Κίνα, από την Κίνα γίνει στην Κίνα, μετατρέπεται σε παρκέ και επανέρχεται στην Κίνα, ε, στη Γαλλία, συγγνώμη. Δεν είναι φρικτό αυτό το πράγμα. Στη, στο πλαίσιο ενός φόρου του άνθρακα στα σύνορα να υπάρχει ένα αποτρεκτικό τέτοιο αποτέλεσμα για να μειωθεί οι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα που επηρεάζει, επηρεάζεται από τις οδικές και από τις ε, υπόλοιπες ε, μεταφορές. Ε, τώρα, Λέμε για μείωση των αερίων του θερμοκηπίου. Εσείς τι πιστεύετε, γιατί εγώ νομίζω ότι είναι αυτό ένα εργοστάσιο αερίων. Αυτή την αποθήκευση του διοξιδίου του άνθρακα υπογείως. Τι γίνεται με την έρευνα σχετικά. Θα είμαστε έτοιμοι δεδομένων των προθεσμιών που πρέπει πραγματικά να μειώσουμε με δρακόντια μέτρα τα... τις εκπομπές αερίων. Τι επιπτώσεις θα έχει η υπόγεια αποθήκευση. Ευχαριστώ πολύ. Τελευταία παρέμβαση η κυρία Λεπάζ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κυρία Διευθύντρια. Δύο σύντομε παρατηρήσει. Πρώτο, για τα όσα είπε κάποιο συνάδελφο προηγουμένω για την πρόσβαση στι πληροφορίε του οργανισμού. Για μα είναι ένα στοιχείο θεμελιώδε και το παρελθόν είχα την ευκαιρία να δουλέψω πάνω σε δικά σα έγγραφα πώς μπορούμε να φτιάξουμε ένα σύστημα που θα επιτρέπει σε καθέναν από τους ευρωβουλευτέ που το επιθυμεί να ε, πάει πολύ γρήγορα και να βρει αυτό που χρειάζεται. Να, δεν ξέρω, να είναι συνδρομητή σε κάποιο <laughs> site, κάποιες διευκολύνσει για να μπορούμε να δουλέψουμε πιο γρήγορα. Είναι μια λεπτομέρεια βέβαια μπορεί να σα φαίνεται δευτερεύουσα σημασία, αλλά από την άποψη ενό ευρωβουλευτή δεν είναι και τόσο λεπτομέρεια. Τώρα, για την ουσία, και για το θέμα της προσαρμογής της κλιματικής αλλαγής. Να βάλουμε, δηλαδή, ε, να μπούμε σε ένα ρυθμό για να αλλάξουμε τον τρόπο παραγωγής, να αλλάξουμε τον τρόπο ζωής μας, να συνειδητοποιήσουμε ακριβώς πόσα πράγματα θα αλλάξουν για μας. Και άρα να δουλέψουμε για την ε, δημιουργία σχεδίων προσαρμογής ε, για τις κλιματικές αλλαγές. Με αντικειμενικά στοιχεία που θα μπορούσατε εσείς να μας δώσετε, ίσως θα ήταν ε, το πιο χρήσιμο, το πιο πρακτικό που θα μπορούσαμε να κάνουμε προς όλους τους φορείς. Είτε είναι η επιχειρήση, είτε είναι η κοινωνία των πολιτών, γιατί ακριβώς είναι ένα μέτρο, ένα τρόπος μάλλον, για να ενημερώσουμε για το τι θα συμβεί και για να προσαρμοστούμε και να με έχει και προσωπικό συμφέρον κάτι τέτοιο, να είμαστε έτοιμοι για αυτές τις μετατροπές που σίγουρα θα τις βιώσουμε, γιατί πέρα από την εξαίρετη έκθεση για, τον, για τις άλπες, να μας πείτε τι σκουπεύει να κάνει προς αυτή την κατεύθυνση ο οργανισμός. Ορίστε. Τελευταίος γύρος από ερωτήσεων, θέλουμε τις απαντήσεις σας. Σας ευχαριστώ. Πλάκα έχει. Πλάκα έχει. Απαντάς όλες αυτές τις ερωτήσεις. Ωραία. Λοιπόν, αρχίζω από τα βιοκαύσιμα και γενικότερα ε, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τη χρήση γης. Μου λένε υπεύθυνα ότι τα βιοκαύσιμα της νέας γενεάς, της δεύτερης γενεάς θα βγουν του χρόνου. Τι σημαίνει αυτό. Ενδεχομένως να έχουμε και τρίτη γενεά. Ε, υπάρχει σημαντική βελτίωση στην καταλητική δράση και στο τι θα αποδώσουν. Ε, χαίρομαι πάρα πολύ. Ωραίο είναι αυτό. Εντάξει, αυτό ήταν το πρώτο. Και το δεύτερο, και θα το γνωρίζετε όλοι πολύ καλά, γιατί ήταν μια συζήτηση που ακούστηκε μετά το στόχο, γιατί υπόθηκε ότι ο στόχος μπορεί να ήταν ε, όχι ο αηφόρος και θα αυξηθεί η ζήτηση και τι σημαίνει αυτό για άλλα μέρη του κόσμου. Κοιτάξτε, έχουμε όλο και περισσότεροι επιρροή και σταματούν τα βιοκαύσιμα αυτά από το να εισέρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί τα συζητάμε και σε θέματα εμπορίου, αλλά ακόμα υπάρχει πολύ μεγάλη δυνατότητα να χρησιμοποιούμε βιοκαύσιμα για την οικονομία των καυσίμων. Αλλά χρησιμοποιώντας βιοκαύσιμα σημαίνει ότι από κάπου αλλού θα στερηθεί αυτό ε, ε, δηλαδή, ε, αν θέλουμε ε, να καλλιεργούμε φυτά για βιοκαύσιμα, για βιομάζα, να φτιάξετε ένα εργοστάσιο δίπλα ακριβώς, για να είναι μικρές οι αποστάσεις. Και το θέμα της χρήσης γης. Βλέπουμε αποψήλωση δασών. Δεν θυμάμαι τα τελευταία στοιχεία, αλλά νομίζω 30 με 40% των δασών παγκοσμίω έχουν αποψηλωθεί το τελευταίο αιώνα. Είναι τεράστια αυτή η κάλυψη που χάνουμε και όταν κανείς χάνει δάσος, χάνει ε, δυνατότητα και του εδάφους δυνατότητα να συγκρατεί διοξίδιο του άνθρακος και να απορροφά. Και τα τελευταία 20 χρόνια περίπου έχουμε χάσει, αν δεν απατώμε, 15% της δυνατότητας των εδαφών να απορροφούν το διοξίδιο του άνθρακα. Και αυτό πάει και στους ωκεανούς. Δηλαδή το θέμα δεν είναι μόνο τα δέντρα που χάνουμε, αλλά η δυνατότητα λειτουργίας του οικοσυστήματος γενικά. Αυτό όταν το συζητήσαμε ε, πέρσι, τα βιοκαύσιμα και φέτος, δεν το λάβαμε υπόψη. Το θέμα της χρήση γη για μας είναι το πιο ε, ουσιαστικό και η δική μα συνεισφορά από τον οργανισμό και πραγματικά δεσμεύομαι ενώπιον σας είναι το εξή. Στην Ευρώπη ελπίζω μέχρι τα τέλη του έτους να έχουμε αυτή την ήρεμη επανάσταση, ελπίζω, στη στατιστική. Διότι ακούσαμε ε, τον επικεφαλής της Eurostat να αναφέρεται εκτενώς στο θέμα αυτό και σε συμφωνία με τον ΟΗΕ ότι θα υπάρχει ε, περιβαλλοντική λογιστική και θα χρησιμοποιείται παράλληλα με την κανονική οικονομική λογιστική. Ε, αυτό καμιά φορά το ονομάζουν πέρα από το ΑΕΠ. Δεν είναι μόνο αυτό όμως. Ε, μιλάμε για την απασχόληση, μιλάμε ας πούμε για τους αριθμούς, για τη ε, δημιουργία του ΑΕΠ. Θα πρέπει να μπει και το περιβάλλον ως παράμετρος. Και επανέρχομαι σε αυτό που ρώτησε ο Καλ Σλούτερ. Θα πρέπει να δώσουμε κίνητρα στον κόσμο, να ενθαρρύνουμε για αλλαγή του μοντέλου κατανάλωσης. Να πούμε λοιπόν τι κάνουμε, πώς καταναλώνουμε, μπορέσουμε να καταφέρουμε η Ευρώπη και οι Εθνικές Στατιστικές Υπηρεσίες και η Eurostat να καταλάβουν ότι βάζουμε και μια περιβαλλοντική λογιστική και είμαστε τμήμα των υπολογισμών για να δούμε τι γίνεται με τη χρήση γης, με την αλλαγή στη χρήση γης, τι γίνεται με τη, τη, λογιστική των υδάτων και, ε, ε, ή των δασικών πυρχαγιών όπως είπατε, αλλά ξέρουμε και πού είναι το νερό, έτσι για να δούμε τι γίνεται με τον υδροφόρο ορίζοντα και τις υπόγειες δεξαμενές. Είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά, αλλά θα πρέπει να αλλάξει ο διάλογος που γίνεται παγκοσμίως. Και γιατί λέω παγκοσμίως, διότι η υπηρεσία μας, ο οργανισμός στην Κοπεχάγη, μαζί με τους συναδέλφους μας στη Βραζιλία και παντού στον κόσμο, θα ε, συζητήσουν για το πώς παγκοσμιμοποιείται αυτή η υπόθεση. Γιατί μιλάμε για τη διαρροή ε, βιομηχανιών που παράγουν πολύ διοξίδιο του άνθρακα ή για τις δασικές πυρκαγιές, θα υπάρχει μια παγκόσμια δυνατότητα συζήτησης και σύγκρισης. Και αυτή είναι η άλλη πλευρά του νομίσματος κλιματικής αλλαγής. Για να ε, λογοδοτούμε κιόλα για το τι κάνουμε, ποιοι είναι οι πόροι, από πού τους βρίσκουμε για να είναι φόρος η οικονομία, αλλά και τι χάνονται, ε, ας πούμε, στα παρθένα δάση, τα τροπικά. Δηλαδή, standards, πρότυπες, προδιαγραφές ε, για ε, λογιστική περιβάλλοντος αλλά και λογιστική των υδάτων. Θα συγκλονιστείτε να δείτε πώς στην Ευρώπη έχουμε ε, χρησιμοποιήσει το νερό και για τα εδάφη και για την ποιότητα της ατμόσφαιρας και τα λοιπά. Κάτι άλλο που θα κάνουμε τα επόμενα χρόνια είναι να συνδέσουμε την παγκόσμια παρακολούθηση και συστήματα ασφαλείας που συνδέονται με φυσικούς πόρους και πάλι μέτρηση των φυσικών πόρων με το Γαλιλαίο να βρούμε έναν τρόπο να είμαστε πολύ πιο ακριβείς στις μεταφορές μας. Κάτι που δεν έχουν οι μεταφορές είναι ένας καλός μηχανισμός ε, εντοπισμού. Ε, καλή ευρωβινιέτα, αλλά τι γίνεται με το καμποτάζ, ας πούμε, τι γίνεται με τα φορτηγά που πηγαίνουν έρχονται άδεια και μεταφέρουν αέρα πολλές εταιρείες πάνε ένα προϊόν από ένα μέρος της Ευρώπης σε ένα άλλο και γυρνάνε άδεια μετά. Γιατί δεν υπάρχει τρόπος να ε, γίνει μεταφορά με άλλο εμπόρευμα. Αυτό θα πρέπει ε, να το αντιμετωπίσουμε. Το, ο Γαλιλαίος λοιπόν και το GMES μπορούν να μας βοηθήσουν έτσι ώστε στο μέλλον να έχουμε μια λογική πολιτική για τις μεταφορές. Τώρα για τα ποσοστά. Ήταν σωστά τα νούμερα που είπατε για τις θαλάσσιες αερομεταφορές και τις υδρομικές και για την Ευρώπη και παγκοσμίω. Έχετε δίκιο. Ε, οι μεταφορές εμπορευμάτων όμως είναι δύσκολο να αντιμετωπιστούν, αλλά είπαμε θα πρέπει να βάλουμε όρια Στι εκπομπές ε, στο ίδιο το φορτηγό. Ήδη βλέπουμε να αλλάζουν οι στόλοι. Ε, το CCS λειτουργεί η δέσμευση και αποθήκευση του άνθρακα. Ελπίζω, έχουμε οδηγία ολόκληρη, αλλά χρειάζεται τώρα πολύ μεγάλη προσπάθεια το επόμενο διάστημα. Επιλέγονται τα έργα και η τεχνολογία ε, πραγματικά προχωρεί μέσα από μελέτες αντικτύπου και θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και να υπαγρυπνούμε. Τώρα για το φόρο στα σύνορα δεν ξέρω, δασμούς. Το θέμα είναι να παρακολουθήσουμε, να ελέγχουμε πώ είναι οι ροέ των μεταφορών εμπορευμάτων. Και επανέρχομαι σε αυτό που είπε η Κορίν Λεπάζ. Θα μπορούσαμε ε, να έχουμε καλύτερη επικοινωνία, μα είναι δωρεάν στη διάθεση ε, όλων ε, η πληροφόρηση. Προσπαθούμε να μεταφράζουμε ό,τι μπορούμε. Αν είχαμε και περισσότερα χρήματα θα μεταφράζαμε ακόμα περισσότερα. Προσβλέπουμε και ε, επαφιόμαστε στα κράτη-μέλη μας για να μεταφράζουμε αλλά και να ενημερώνουμε τις πληροφορίε. Δεν φτιάχνουμε μόνο εκθέσεις, δεν βγάζουμε εκθέσεις, αλλά και δεδομένα με τρόπο που μπορείτε εσεί να τα χειρίζεστε και να είναι πολύ πιο χρήσιμα στο PDA, στο τηλέφωνο σας ο καθένας ε, με προειδοποιήσεις, με νέα στοιχεία και τις επόμενες εβδομάδες θα λασάρουμε το Ion Earth, δηλαδή στην ιστοσελίδα σας, αλλά και στους προσωπικούς σας υπολογιστές ή στις μηχανές σας, θα έχουμε τα νέα στοιχεία για διοξίδια του θείου, του αζότου, του σωματίδια, ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, του νερού. Θα σας έρχονται τα στοιχεία και θα μπορείτε και εσείς να μας ενημερώνετε και οι πολίτες. Δηλαδή, ε, βαθμία και σταδιακά λανσάρουμε τεχνολογία για να μπορείτε και εσείς να μας ενημερώνετε και με ένα feedback. Πράγματι πιστεύω ότι θα αλλάξει ο κόσμος του χρόνου, ο τρόπος που θα ενημερωνόμαστε και για να έχετε έτσι χρήσιμα στοιχεία. Σας ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις σας, πολύ ενδιαφέρουσες. Βλέπω ένα χεράκι να σηκώνετε. Α, για τις δασοπυρκαγιές, ναι. Ε, στο πρόγραμμα ε, του χρόνου έχουμε μια δραστηριότητα για την πολιτική προστασία και ιδιαίτερα διαχείριση των θεομηνιών ε, για την πρόληψη. Βλέπουμε ότι οι δασικές πυρκαγιές και η λειψιδρία είναι από μόνο του θεομηνία αν δεν υπάρχει ε, σχεδιασμός αλλά θα πρέπει επί τόπου να υπάρχουν οι κατάλληλοι μηχανισμοί αντίδραση με σωστή πληροφόρηση και ενημέρωση την ώρα που συμβαίνουν όλα αυτά. Και αυτά μπαίνουν στο πρόγραμμα του GMES. Θα επανέλθω λοιπόν, ε, επενδύσαμε στην Ευρώπη για να κάνουμε λειτουργικό αυτό το σύστημα και το δορυφορικό και άλλα. Η δουλειά μας τώρα είναι με τα ερευνητικά κέντρα και τα κράτη-μέλη να βάλουμε πολύ περισσότερη ενέργεια στην προσαρμογή, στην επιχειρησιακή δυνατότητα ε, σε θέματα ξηρασίας, δασικών πυρκαγιών και όλα αυτά. Είναι στο πρόγραμμα εργασίας και ελπίζουμε του χρόνου να συνεχίσουμε και να εντατικοποιούμε αυτά ε, που κάνουμε. Και να ξέρει και το κοινό ότι πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο ζούμε στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Ήταν πολύ κατατοπιστική η συζήτηση, νομίζω, και πολύ πιστική. Πολύ καλή δουλειά. Θα τα πούμε στην Κοπεχάγη το αργότερο, κατά τη διάρκεια της διάσκεψης για το κλίμα και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Ε, θα τα πούμε σύντομα. Μην φύγουν τα μέλη, παρακαλώ, γιατί έχουμε μία ερώτηση ακόμα ακούστηκε, εκφράστηκε επιθυμία από πολλές πλευρές η ψηφοφορία για τον κατάλογο της διαρροής του διοξιδίου του άνθρακα να αναβληθεί, carbon leakage. Ε, τώρα όμως θα πρέπει να σκεφτούμε ποια θα ήταν η σωστή και η κατάλληλη μέθοδος να γίνει αυτό. Μερικοί πήγανε στι Ηνωμένε Πολιτείε την ε, περασμένη εβδομάδα και δεν είχαν χρόνο να το μελετήσουν. Έχουμε πραγματογνωμοσύνη και της νομικής υπηρεσίας, γνωμοδότηση. Άλλοι θέλουν να ακούσουν και τον Επίτροπο, τον κύριο Δήμα. Λοιπόν, μία δυνατότητα είναι να αναβληθεί για την Πέμπτη το πρωί στις 10 και οι άλλοι να το αφήσουμε όπως είναι αύριο, αλλά ξέρω εγώ 12 και 4, 12 και 20, όταν θα έχουμε ακούσει τον κύριο Δήμα. Εγώ θα πρότεινα να ε, ψηφίσουμε αύριο, γιατί θα είναι παρόντα όλα τα μέλη έτσι κι αλλιώς το 6 έχει διαγραφεί, τα καλλιντικά φύγανε. Στι 9 ε, η ώρα θα αρχίσουμε αμέσω τη συζήτηση, μετά θα έρθει ο κύριο Δήμα και μετά θα ψηφίσουμε. Συμφωνείτε? Ωραία. Καλώ. Πριν το μεσημεριανό διάλειμμα, λοιπόν, μετά τον κύριο Δήμα, 12 και κάτι, εν πάση περιπτώσει 12 και 20, μπορούμε να ψηφίσουμε. Θα στείλουμε και ένα email προειδοποίηση, να το ξέρετε όλοι. Ευχαριστώ πολύ. Ραντεβού αύριο το πρωί στι 9.